Muy buenas tardes. Les agradezco que tomen... Καθίστε παρακαλώ για να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. A Σας ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι, τα πρώτα μου λόγια απευθύνονται σε όλους εσάς. Θέλω να σας καλωσορίσω εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το να έχουμε την υλοποίηση μιας διακοινοβουλευτικής συνεδρίασης είναι κάτι εξαιρετικό. Είναι εξαιρετικό για πολλούς λόγους και θα επικεντρωθώ σε δύο. Καταρχήν, επειδή συνεδριάζουμε σε, αυτό το, σε αυτή την αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συμμετέχουν 46 μέλη των Εθνικών Κοινοβούλιων που προέρχονται από 26 ε, κοινοβούλια από 21 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εγώ πιστεύω ότι ήδη αυτός ο αριθμός ε, είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικός και μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι εξαιρετικές οι περιστάσεις. Αλλά επίσης είναι εξαιρετικό το ότι μπορούμε να έχουμε την δυνατότητα να συζητήσουμε με την παρουσία της ε, κυρίας Επιτρόπου, της κυρίας Δαμανάκη, που την ευχαριστώ πάρα πολύ που παρευρίσκεται σήμερα εδώ. Όπως πάντα προσπαθεί να έρχεται εδώ ε, ενωπιών μας γιατί αυτή η συζήτηση που θα κάνουμε σήμερα είναι θεμελιώδη σε μια κέρια χρονική στιγμή για την Ευρωπαϊκή Αλία καθώς ε, τώρα υλοποιούμε ένα προβληματισμό για την κοινή αλληλευτική πολιτική και θέλουμε να δούμε ποιο θα είναι το μέλλον αυτού του τομέα τα επόμενα έτη. Και σας ευχαριστώ ε, για την προσπάθειά σας ε, να έλθετε εδώ, να παρευρεθείτε σε αυτή τη συνεδρίαση. Είμαι πεπισμένος ότι θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Είναι το πιο αξιόλογο μέσο που μπορούμε να έχουμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή η ανταλλαγή απόψεων ε, μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έτσι ώστε από κοινού να μπορέσουμε να καταλήξουμε στην καλύτερη δυνατή μεταρρύθμιση. Και θα σας πω πώς ε, θα λάβει η χώρα αυτή η συνεδρίαση. Γιατί εμείς επιθυμούμε να πάρουν το λόγο όσο το δυνατόν περισσότεροι βουλευτές, ε, κυρίως από τα Εθνικά Κοινοβούλια που παρευρισκόνται σήμερα εδώ. Έτσι λοιπόν, όταν εγώ θα ολοκληρώσω την παρουσίαση αυτή, θα πάρει το λόγο η κυρία Επίτροπος και θα μιλήσει περίπου για 15 λεπτά. Στην συνέχεια θα έχουμε μία ανταλλαγή απόψεων και αλλάξαμε τον αρχικό συνδυασμό γιατί θεωρήσαμε ότι ήταν σημαντικό η κυρία Επιτροπός να έχει τη δυνατότητα να απαντήσει στις ερωτήσεις που μπορείτε να τις θέσετε για μισή ώρα περίπου. Και στη συνέχεια θα περάσουμε Δηλαδή αφού θα μας εγκαταλείψει η κυρία Επίτροπος ε, θα περάσουμε στο επόμενο μέρος της συζήτησης, ε, θα πάρουν το λόγο οι εισηγητές στα διάφορα πάνελ και θα έχουμε το ίδιο σύστημα. Μία παρέμβαση περίπου 10 λεπτών για κάθε έναν από τους εισηγητές ε, και κατόπιν θα έχουμε μία σειρά ερωταπαντήσεων που θα διαρκέσει 30-35 λεπτά. Αυτό και για τα τρία πάνελ που έχουμε προβλέψει και στη συνέχεια θα εξάγουμε και συμπεράσματα. Τώρα, πώς ε, θα γίνει η συζήτηση ή οι ερωταπαντήσεις. Θα θέλαμε, όπως είπα και πριν, όλοι να μπορέσουν να πάρουν το λόγο, αλλά δεν θα είναι εύκολο. Έτσι λοιπόν σας ζητώ να συνεργαστείτε, να σεβαστείτε το χρόνο. Όποιος λάβει το λόγο Ξέρετε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ποτέ δεν ξαπερνάμε το 1,5, το πολύ δύο λεπτά. Και αν ε, δεν σεβαστείτε το χρόνο θα πρέπει να σας ευχαρίσω το λόγο. Δύο λεπτά νομίζω ότι είναι αρκετός χρόνος ε, για να μπορέσετε να εκφράσετε τις ανησυχίες σας ή να θέσετε τις ερωτήσεις σας. Είναι αλήθεια, δεν ε, είναι επαρκές ο χρόνος για να προβληματιστούμε επαρκώς επί του θέματος, αλλά το πολύ δύο λεπτά θα έχετε χρόνο στη διάθεσή σας. Και Τώρα, διατύπωση των ερωτήσεων. Για να μην ε, σηκώνετε το χέρι, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας να διακρίνουμε ποιος ζητάει το λόγο. Έχετε στα, μπροστά σας, ενώπιόν σας, ε, τέσσερα χαρτιά. Ένα κίτρινο, ένα άσπρο, ένα πράσινο και ένα πορτοκαλί. Με αυτά μπορείτε να δηλώσετε αν θέλετε το λόγο ή αν θέλετε να κάνετε ερώτηση για το λευκό χαρτί, ερώτηση προς την κυρία Επίτροπο. Αν θέλει λοιπόν ε, κάποιος να θέσει ερώτηση στην Επίτροπο, να συμπληρώσει το έγγραφο, θα το πάρουν οι αρμόδιοι και κατόπιν θα φέρουν σε εμάς αυτά τα χαρτιά για να κάνουμε και εμείς τον κατάλογο. Τώρα το κίτρινο χαρτί θα είναι για ερωτήσεις στην κυρία Ρόντουστ ε, για το βασικό κανονισμό, το πορτοκαλί χαρτάκι για τη συζήτηση για την ΚΟΑ ε, και τη συζήτηση που έχουμε τον κύριο Στεβίνσον και το πράσινο για το Ταμείο ε, για το οποίο είναι ο κύριο Κάντε και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσα και Τώρα βέβαια ε, κάποιος ε, δεν μπορεί να παρουσιάσει και τα τέσσερα χαρτάκια να θέσει τέσσερι ερωτήσει, να περιοριστούμε σε ένα. Και κατόπιν, αν δούμε ότι έχουμε χρόνο και δυνατότητα για περισσότερε ερωτήσει, τότε θα δώσουμε την ευκαιρία σε όλου, όσου το επιθυμούν. Και γι' αυτό επαναλαμβάνω, είναι σημαντικό να σεβαστούμε όσο το δυνατόν περισσότερο το χρόνο και να περιοριστείτε στα δύο λεπτά ο καθένας. Αυτό για τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων. Τώρα, για τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, φυσικά θα έχετε και εσείς την ευκαιρία να θέσετε ερωτήσει, αν το επιθυμείτε. Έχουμε προβλέψει ένα σύστημα για δύο, ε, δύο άτομα από τα Εθνικά Κοινοβούλια και από τις γερουσίες και ένα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έτσι λοιπόν ε, μας ενδιαφέρει να κάνουν ερωτήσεις περισσότερο τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων που είναι σε επίσκεψη. Και αν κάποιο θέλει να θέσει μια ερώτηση κατά τη διάρκεια λοιπόν της συζήτησης, να συμπληρώσει το κατάλληλο χαρτάκι και αν δεν θέλετε να θέσετε κάποια ερώτηση, αν δεν έχετε κάποια αμφιβολία, να ξεκινήσουμε. Να δώσουμε το λόγο στην ε, κυρία Δαμανάκη. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Thank you, President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που διοργανώσατε τη σημερινή συνεδρίαση και μου δώσατε την ευκαιρία να παρευρεθώ ενώπιόν σας. Αξιότιμοι βουλευτές ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αξιότιμοι βουλευτές των Εθνικών Κοινοβουλίων, θα ήθελα να σας καλωσορίσω να καλωσορίσω του βουλευτέ των Εθνικών Κοινοβουλίων όλους ιδιαίτερω. Όπω είπα τον Οκτώβριο όταν συναντηθήκαμε για τελευταία φορά, Είμαι πεπισμένη ότι η μεγαλύτερη συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων θα αναβαθμίσει την ποιότητα και τη φύση αυτή τη μεταρρύθμισης. Εν ολίγης, θεωρώ ότι δεν μπορεί να προχωρήσει η μεταρρύθμιση αν δεν εμπλακούν και συμμετάσχουν ενεργά τα Εθνικά Κοινοβούλια. Γι' αυτό το λόγο Προσκαλέσαμε εκπροσώπου των Εθνικών Κοινοβουλίων σήμερα, γι' αυτό το λόγο ήδη μετέβην σε διάφορα εθνικά κοινοβούλια και σκοπεύω να επισκεφθώ πολλά εθνικά κοινοβούλια ακόμη προτού εγκριθούν οι προτάσει τη Επιτροπή. Σε δύο εβδομάδε θα πάω στην Ιταλία, παραδείγματο χάρη. Ελπίζω ότι όλα τα εθνικά κοινοβούλια θα μου απευθύνουν πρόσκληση για διάλογο. Έχω ήδη καταγράψει τις απόψεις που έχετε εκφράσει μέχρι τούδε. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρατήρησα τα όσα σας απασχολούν και εν γέννη θεωρώ ότι υπάρχει συνένεση περί της ανάγκης μεταρρύθμισης που παρατηρείται στην Ένωση. Όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει να στραφούμε προς μια πιο βιώσιμη προσέγγιση. Η χρηστή ε, οικονομική επίδοση της βιομηχανίας μπορεί να προέρχεται μόνο από υγιή ε, ηχθιαποθέμε. Αυτά αυτή είναι η γενική προσέγγιση. Πιστεύω ότι υπάρχει συνένεση, όπερ και με χαροποιεί σίγουρα. Κάποιοι θα επιθυμούσαν ακόμη πιο φιλόδοξες προτάσεις. Έχω λάβει συγκεκριμένα εισηγήσει ε, που προτείνουν μια, ένα πιο φιλόδοξο, αν θέλετε, προσανατολισμό. Άλλοι είναι ικανοποιημένοι με την καθεστική ατάξη, άλλοι πάλι απευθύνουν επικρίσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θεωρούν ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε καλύτερα μια ε, σταδιακή προσέγγιση. Πάντως υπάρχει ένας κοινός παρονομαστή, δηλαδή όλοι θέλουν με αυτήν την μεταρρύθμιση να ανατρέψουμε ε, την παρακμή του κλάδου. Πιστεύω ότι αυτό συνιστά κοινό στόχο για όλους. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο κοινός παρονομαστής σε συνδυασμό δε με την προσοχή και την αφοσίωσή σας ε, για αυτό το θέμα. Θεωρώ ότι ε, υπάρχει υλικό ώστε να οικοδομήσουμε μια ευρύτερη συνένεση θα εξετάσουμε κάποια από τα πλέον αφιλεγόμενα ζητήματα για να έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε εις βάθος. Μία επίκριση που ακούω επανειλημμένα και διαβάζω σε διάφορες γνωμοδοτήσεις ε, σχετίζεται με τον δεσμευτικό, υποχρεωτικό χαρακτήρα των προτινόμενων αλλαγών. Ας δούμε παραδείγματο χάρη τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση που πρέπει να επιτευχθεί μέχρι το 2015. Οι πλήστοι συμφωνούν, αλλά θα ήθελαν να προσθέσουν στα αγγλικά το where possible, όπου δει. Σχετικά με την απαγόρευση απορρίψεων, λέτε ναι επί της αρχής, αλλά ζητάτε περισσότερο χρόνο και περισσότερη ευελίξη τα Μεταβιβάσιμες ε, ε, εκχωρήσεις, ε, μάλιστα, εδώ... Υπάρχουν περισσότεροι που δεν συμφωνούν με αυτήν την αλλαγή. Άλλοι συμφωνούν με την αλλαγή, δεν θέλουν να είναι υποχρεωτική διάταξη. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι χρειαζόμαστε μια πιο δεσμευτική προσέγγιση κατά την μεταρρυθμιστική αυτή προσπάθεια. Για ποιο λόγο, διότι ε, ε, θεωρώ και τώρα απευθύνομαι στου βουλευτέ των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πιστεύω ότι δεν μπορούμε παρά να υπομιστούμε πολιτικέ ευθύνε. Δεν μπορούμε να τα αφήνουμε όλα για τα παιδιά μα, για τι επόμενε ε, γενιέ. Πολλοί από εσά υποβάλλουν προτάσει για να συμπεριλάβουμε τις μαγικές λέξεις στη μεταρρύθμιση. Where possible, όπου δει. Μα τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει ε, να ε, εισαγωγή μιας αλλαγής όπου δει. Μάλιστα, μπορεί να σημαίνει ε, ότι θα την εγκρίνουμε την αλλαγή. Μπορεί όμως να σημαίνει ε, ποτέ ε, όταν λέμε όπου όπου, όπου είναι εφικτό, ε, είναι ασαφή η διατύπωση και δεν είναι βιώσιμη εναλλακτική λύση. Δεν έχουμε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ούτε και συγκεκριμένο στόχο υλοποίηση. Όσο εξακολουθούν να ισχύουν αυτό, θα μεταθέτουμε διαρκώ τη μεταρρύθμιση και θα αποτύχει παταγωδό. Ήδη το έχουμε κάνει αυτό επί σειρά ετών. Ήρθε η ώρα λοιπόν να αποκτήσουμε κάποιου δεσμευτικού στόχου. Και εγώ θα ήθελα σήμερα να συζητήσουμε ποιοι ακριβώ θα είναι αυτοί οι δεσμευτικοί στόχοι. Νομίζω ότι μπορούμε να το συζητήσουμε μεταξύ μας. Πιστεύω επίσης ότι μπορούμε να βρούμε ε, κοινά σημεία, αλλά είναι ξεκάθαρο και θέλω εξ αρχή να το διευκρινίσω ότι αν δεν έχουμε συγκεκριμένου στόχου θα αποτύχουμε. Ξέρω, γνωρίζω ότι οι στόχοι τη πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι δύσκολοι, είναι αυστηροί και ορισμένοι πιστεύουν ότι είναι πρόωρα όλα αυτά. Αλλά είναι ο μόνο τρόπο, είναι ο μονόδρομο για να επιτύχουμε βιώσιμη διαχείριση των αποθεμάτων. Η βιώσιμη διαχείριση είναι κατεπήγον θέμα. Ε, χρειαζόμαστε ένα σαφή οδικό χάρτη με ρεαλιστικού ε, με ρεαλιστικά ορόσημα ε, και σταδιακά ορόσημα. Θα ήθελα να εξηγήσω γιατί αν μεταθέσουμε τη μεταρρύθμιση τότε μετά από μία πενταετία ή μία δεκαετία τότε θα είναι ακόμη δυσχερέστερη η μεταρρύθμιση. Δεν θα είναι ευκολότερη, θα είναι δυσχερέστερη διότι θα έχουν στο μεταξύ συσσωρευτεί τα προβλήματα και θα έχουν μεγεθυνθεί. Γι' αυτό το λόγο τώρα είναι η ώρα να δράσουμε. Ας πάρουμε τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Ε, στα αγγλικά. Εάν ε, σκοπεύουμε να επιτύχουμε τα ε, επιθυμητά επίπεδα για όλα τα αποθέματα, ε, πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε μια καταλεκτική ημερομηνία. Κάποιοι κρίνουν ότι δεν πρέπει να είναι το 2015 η προθέσμια μας. Εγώ θα διαφωνήσω και για τρεις λόγους. Ο πρώτος είναι ότι οι προσπάθειες για να επιτύχουμε τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση έχει ήδη υλοποιηθεί για κάποια από τα αποθέματα. Από 38 ε, αποθέματα το 2009 κρίναμε ότι μόνο 5 ήταν σε μη βιώσιμα επίπεδα. Ε, τώρα, σήμερα, έχουμε φτάσει στα 20 αποθέματα. Έχει σημειωθεί πρόοδο και υποπίεση κιόλα. Όταν εγώ ανέλαβα το αξίωμά μου, το Συμβουλίο ήταν κατηγορηματικά αντίθετο. Βήμα-βήμα όμω το καταφέραμε. Μπορούμε να διασχίσουμε και την υπόλοιπη απόσταση. Ε, επίσης, ο μπακαλιάρο για την Ανατολική Βαλτική. Η μεγάλη υπεραλίευση μέχρι νόση και τώρα έχει φτάσει σε βιώσιμα επίπεδα. Το ίδιο ισχύει ε, για τον ε, Βισκαϊκό κόλπο, για τη διάφορα ψάρια όπως η Ρέγκα ή ο Εγκλεφίνος. Έχουμε επανέφερει τα αποθέματα σε βιώσιμα επίπεδα και άρα μπορούμε να σημειώσουμε και άλλη πρόοδο. Ο, δεύτερον, ο λόγος όταν μειώνεται η ελιευτική ικανότητα, μεγαλώνουν τα ψάρια σε μέγεθο και σε βάρο. Επίση, είναι ευκολότερο να αλλιευθούν και μειώνεται το κόστο, αυξάνοντα ταυτόχρονα το κέρδο ε, του κλάδου. Ε, αυτό το μήνα ε, ένα ίδρυμα που ονομάζεται New Economics Foundation ε, μας υπενθύμησε και πάλι πόσο σημαντικό είναι να έχουμε μια χρηστή και βιώσιμη διαχείριση των αλλιευτικών πόρων. Λένε ότι στην Ευρώπη των 27 κάθε χρόνο θα μπορούσε ο κλάδος ε, να έχει 1,8 δις ευρώ επιπρόσθετα, δηλαδή επί τρία οι επιδοτήσεις που δίνουμε τώρα και θα καταλήξουμε σε 83.000 νέες θέσεις απασχόλησης

83.000 ε, θέσεις ε, απασχόλησης ε, αν επαναφέρουμε τα αποθέματα σε μέγιστα, στη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Με το τωρινό οικονομικό δυσχερές περιβάλλον καταλαβαίνετε ότι πρέπει να δράξουμε τις ευκαιρίες. Δεν μπορούμε να μεταθέσουμε την προσπάθεια. Επίσης, μέχρι το 2015 έχουμε τη νομική υποχρέωση να αποκαταστήσουμε τα αποθέματα βάσει τη σύμβαση του ΙΕ και το δίκαιο της θάλασσας καθώς και το πλάνο του Johannesburg για την υλοποίηση αυτών των των αποφάσεων. Θέλουμε να δείξουμε στη διεθνή κοινότητα ότι σηκώνουμε τα χέρια ψηλά όταν ε, ταυτόχρονα ζητάμε ηγετικό ρόλο για την Ευρωπαϊκή Ένωση για ένα καλύτερο περιβάλλον. Αν θέλουμε να έχουμε ηγετικό ρόλο, λοιπόν πρέπει να εφαρμόζουμε και όλε τι αποφάσει. Θα ήθελα τώρα να, να περάσω σε ένα διαφορετικό θέμα, την απαγόρευση απορρίψεων. Σταδιακά θα υλοποιηθεί. Αυτό σα διαβεβαιώ δεν γίνεται νυχθημερών να εφαρμοστούν αυτά, το γνωρίζω αυτό, ξέρω ότι χρειαζόμαστε περισσότερε ε, λύσει για τεχνική αρρωγή. Συμφώνω, πρέπει να είναι σταδιακή η προσέγγιση ε, για να υλοποιηθεί τελικά η απαγόρευση Ε, Η κοινή γνώμη είναι κάθετα εναντίον των απορρίψεων. Σήμερα υπάρχουν ε, τουλάχιστον 70 διαφορετικέ πρωτοβουλίε κατά της απόρρεψης ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση από του αλληλεί, παραδείγματο χάρη που ε, βρίσκουν τρόπους για να ε, αλλιεύουν πιο επιλεκτικά ή από λιανοπολιτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ε, ξέρετε τι κάνουν, βγάζουν από τις προμήθειές του συγκεκριμένα είδη όταν απειλούνται τα αποθέματα ή όταν δεν χρησιμοποιούνται επιλεκτικές τεχνικές, αλλιευτικές τεχνικές. Δεν έχουμε εμείς εναλλακτική λύση. Η ίδια η αγορά ε, έχει αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία. Πολλές φορές τις κατακρίνουμε, αλλά τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση κάνουν τη δική μας δουλειά οι ίδιες οι αγορές, οι ηλιανοπολιτές ε, καταγράφουν οι ίδιοι τα απειλούμενα είδη. Ε, και τα αποσύρουν από, τις, ε, από τους προμηθευτικούς ε, καταλόγους τους. Επιπιστεύω ότι είναι πολύ θετικές αυτές οι πρωτοβουλίες και θα πρέπει να υποστηρίξουμε τον κλάδο στην προσπάθειά του. Να υποστηρίξουμε επίσης ε, την επιλεξιμότητα. Χρειαζόμαστε λοιπόν εξοπλισμό μεγαλύτερη επιλεξιμότητα και θα χρηματοδοτήσουμε σε ποσοστό μέχρι 85% και ενίοτε και υψηλότερο ποσοστό από αυτό, ούτως ώστε να προμηθευτούν οι αλληλείς τις το νέο αυτό επιλεκτικό εξοπλισμό. Χρειαζόμαστε λοιπόν ούτω ή άλλω ε, δεσμευτικό στόχο. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε όλα στην ε, βιομηχανία. Έρχονται κάποιοι και μα λένε γιατί πρέπει οπωσδήποτε να είναι υποχρεωτική η απαγόρευση. Α το αφήσουμε, α είναι θελοντικό το σύστημα, μάλιστα, αλλά θα σα το πω ομά. Έχω δει στην πρόταση, στις προτάσεις μάλλον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα τελευταία 7 χρόνια τόσες πολλές φορές αυτό τον όρο απαγόρευση απόρριψης και τίποτα δεν έχει γίνει. Μα αν ακολουθήσουμε λοιπόν την πεπατημένη σε μια πενταετία πάλι εδώ θα είμαστε, μάλλον ε, ο, προκάτω, ο διάδοχός μου θα είναι ή η διάδοχός μου και πάλι θα συζητάτε τι θα κάνουμε με τις απόρριψεις. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε καταληκτική ημερομηνία λοιπόν για την απαγόρευση απόρριψης. Δεν, ε, δεν ε, Μπορούμε να βρίσκουμε συνέχεια δικαιολογίε. Θα δούμε τι είναι ρεαλιστικό. Μπορούμε να το συζητήσουμε ω προ το χρονοδιάγραμμα. Επίση, χρειαζόμαστε λύσει για τη μεικτή αλία, διότι δεν έχουμε επιλύσει ακόμη όλα τα προβλήματα. Σίγουρα θα τα καταφέρουμε, αλλά ξαναλέω, ε, στο κάτω-κάτω της γραφής θα χρειαστούμε οπωσδήποτε ε, δεσμευτικούς στόχους σχετικά τρώμε τις μεταβιβάσιμες ε, παραχωρήσεις. Ξέρω πόσο αμφιλεγόμενο είναι αυτό το θέμα. Ε, και λένε κάποιοι ότι είμαι υπέρ ε, αυτή τη ιδέα γιατί είμαι φιλελεύθερη. Ε, δεν ξέρω αν είμαι φιλελεύθερη. Εγώ δεν βρίσκω ότι είμαι φιλελεύθερη. αλλά στον κανονισμό, στον ισχύοντα κανονισμό, πρώτη φορά υπάρχει ρητή μνήμα της δημόσιας, του δημόσιου ιδιοκτησιακού καθεστώ των ηχθιαποθεμάτων. Το ίδιο ισχύει λοιπόν και για τι εκχωρήσει, μεταβάσιμε εκχωρήσει, για ένα συγκεκριμένο ε, χρονικό διάστημα. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σκοπεύω να κάνω με την απελευθέρωση της αγοράς, τις χρειαζόμαστε αυτές τις μεταβιβάσιμες εκχωρήσει. Τι πρέπει ακριβώς να συζητήσουμε όταν μιλάμε για πλεονάζουσα ε, ε, αλλιευτική ικανότητα των στόλων. Νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε από κοινού λύσεις. Επίσης θα ήθελα να σε ενημερώσω ότι υπάρχουν πάρα πολλές δικλείδες ασφαλείας για τα κράτη-μέλη, αν το επιθυμούν τα κράτη-μέλη, για να αποφύγουμε αυτό που φοβάμαι φοβάστε ε, ότι θα ε, υπάρχει μια κεντρική διαχείριση όλων των δικαιωμάτων. Τα κράτη-μέλη μπορούν να εισαγάγουν επιπρόσθετες δικλείδες ασφαλείας. Θα ήθελα όμως να σας πω το εξή. Αν θέλουμε ε, να εξαιρεθούν οι στόλοι μικρής κλίμακας, 80% των σκαφών θα εκφεύγουν το κανονισμό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι λύσει υπάρχουν. Χρειαζόμαστε όμως τη βοήθειά σας, είναι αναγκαία, ούτως ώστε ε, οι εθνικές αρμόδιες αρχές ή στις εκλογικές περιφέρειές σας να συνειδητοποιήσουν όλοι πόσο κατεπήγον είναι αυτό το ζήτημα. Ε, σίγουρα σε σχέση με τι ημερομηνίες ε, στόχους ε, φαίνονται αυστηρές ε, αλλά θα δείτε μέσα στη συζήτηση ότι είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Είμαι ανοιχτή για οποιαδήποτε, οποιαδήποτε πρόταση διευκόλυνσης της διαδικασίας έχετε. Απευθύνω έκκληση σήμερα προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα Εθνικά Κοινοβούλια, το Συμβούλιο ε, να μας ακολουθήσουν, ε, να θέσουν υψηλότερους στόχους, χωρίς βεβαίως ε, να αντιβαίνουμε και στις επιμέρους διατάξεις της συνθήκης της Λισαβόνας. Για την περιφερειοποίηση έχουμε ένα έγγραφο της Βρετανικής Αντιπροσωπείας, το αξιολογούμε τώρα, το σκεφτόμαστε, αλλά πραγματικά στείλτε μας όλη ε, τη θέση σας ε, γραπτός ε, για αυτό το πολύ συγκεκριμένο θέμα της περιφερειοποίησης της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Εν κατακλείδη, κυρίες και κύριοι, αν είναι να βασιστούμε στην παρελθούσα εμπειρία, θα διαπιστώσουμε ότι διάφορα συστήματα έχουν επινοηθεί για να αποφύγουμε με οποιοδήποτε δυνατό τρόπο τις μεταρρυθμίσεις. Τα νέα χρονοδιαγράμματα θα βοηθήσουν τους επαγγελματίες να συνειδητοποιήσουν ότι θέλουμε να του βοηθήσουμε για να συμμορφωθούν, θα γνωρίζουν τη θέση μα περί βιωσιμότητας. Ε, κανείς ε, δεν μπορεί να αρνηθεί ότι θα είναι κακοτράχαλος ο δρόμος ε, προς την επίτευξη των στόχων, αλλά δεν μπορούμε να αναβάλουμε τη μεταρρύθμιση γιατί θα επιδεινωθεί η κατάσταση. Θα πρέπει να βοηθήσουμε σε αυτή τη μεταβατική περίοδο τους επαγγελματίε εξού και η λειτουργία του νέου ταμείου. Αυτό το νέο ταμείο θα βοηθήσει του αλλήλου να προσαρμοστούν στι νέε απαιτήσει θα προαγάγει τοπικέ πρωτοβουλίε και οι εγχώριε κοινότητε θα, θα μπορέσουν από μόνε του να αναβαθμίσουν την παραγωγική δραστηριότητα. Αν είναι να συγκρατήσετε κάτι από σήμερα είναι το εξή γνωρίζουμε τι μπορεί να παράγει η θάλασσα ε, και η θάλασσα αποφασίζει ποιου ε, πόρου θα μα δώσει, όχι εμείς. Ε, το αντίθετο προσπαθούσαμε να κάνουμε στο παρελθόν και θα πρέπει το ταχύτερο δυνατόν να αλλάξουμε στάση ούτω ώστε να εξασφαλίσουμε την οικονομική ευημερία και βιωσιμότητα του κλάδου και των παράκτιων περιοχών. Σίγουρα θα αποκομίσουμε ωφέλη 135 εκατομμύρια ευρώ, 135 εκατομμύρια ευρώ είναι το επιπρόσθετο κονδύλιο στι τσέπε ε, των ε, αλλιών ε, με τι αυξήσει δηλαδή των ποσοστών που καλύπτουν την περίοδο από το 2011 έω 2012 διαχειριζόμαστε καλύτερα τα αποθέματα και έχουμε ήδη δώσει αυτά τα 135 εκατομμύρια σαλής και μπορούμε να δώσουμε ακόμη περισσότερα με τη δική σας όμως αρρωγή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η εκλογή σας, ο, ο, ο κλάδος ε, της κάθε χώρας να συνειδητοποιήσει ποιος είναι ο τρόπος σκέψης μας. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων και περιμένω με ανυπομονησία τις παρατηρήσεις και ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. <coughs> Ευχαριστώ πολύ την ε, κυρία Επίτροπο για αυτή την παρέμβαση, να περάσουμε ευθύ αμέσω στη συζήτηση με τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων που έχουν ζητήσει το λόγο. την κυρία Μάκιντο ε, θα ξεκινήσουμε από τη Βουλή των Κοινοτήτων. Παρακαλώ. Για δύο λεπτά έχετε το λόγο. I'd uh, like to thank... Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς ε, κύριε ε, Πρόεδρε και την Επίτροπο για την ευκαιρία που μας δίνετε και περιορίζομαι στη νομική βάση. Χαίρομαι διότι η Επίτροπος χαιρέτησε την συμβολή μας και αναζητεί κι άλλες. Πιστεύουμε ότι θα ήταν λάθος να ξανανοίξει η συζήτηση για τη συνθήκη της Λισαβόνας. Και αναγνωρίζομαι την αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής. Θέλουμε να περιορίζεται στο να υπάρξει μια στρατηγική εποπτεία της ευρωπαϊκής πολιτικής αλίας. Πιστεύουμε ότι ο σωστός τρόπος να προχωρήσουμε είναι να καλέσουμε τα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε συναπόφαση με το Συμβούλιο Υπουργών ώστε να συμφωνήσουν στην τροποποίηση των συγκεκριμένων κανονισμών που εξετάζουμε σήμερα. Πιστεύουμε ότι έτσι είναι θεμητό να προχωρήσουμε, είναι ένας καινοτόμος τρόπος, καινούριο και λύνει το πρόβλημα που παρουσίασε η κυρία Δαμανάκη όταν ε, ήρθε σε εμά ε, στη Βουλή των Λόρδων ότι πρέπει να λειτουργήσουμε στα πλαίσια της νομικής βάσης της συνθήκης της Λισαβόνας. Ε, υπάρχουν αντίγραφα, αντίτυπα για όλους που είναι παρόντες σήμερα και πιστεύω ότι θα υπάρξει θετική ανταπόκριση στις προτάσεις μας. Επίσης, αναγνωρίζοντας τη νομική βάση, συμφωνούμε με τα συμπεράσματα της Επιτρόπου ότι θα πρέπει να δουλεύουμε πάνω σε στέρεη επιστημονική βάση εις ό,τι αφορά τις απορρίψεις, την μέγιστη ευβιώσιμη απόδοση, τις ε, μεταβιβάσιμες ε, εκχωρήσεις. Πιστεύουμε ότι η μεγαλύτερη παραχώρηση που μπορούμε να κάνουμε είναι να τροποποιήσουμε τους κανονισμούς και να δουλέψουμε θετικά στα πλαίσια της συνθήκης της Λισαβόνας, αλλά με μια καινούργια νομική βάση. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Γιάντσεβα τώρα από το Βουλγαρικό Κοινοβουλίο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία ε, Επίτροπε. Η Βουλγαρία θέσπισε την, ε, την πρόταση για την ε, μεταρρύθμιση της κοινή αλλιευτικής πολιτικής και θεωρεί ότι είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι περιφερειακές οργανώσεις, η ανταλλαγή των ορθών πρακτικών και η επιστημονική έρευνα. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να οργανωθεί η επιτυχή συνεργασία μεταξύ όλων των παραευξήνιων χωρών. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι ο εύξηνος πόντος είναι μια θάλασσα ε, που γειτονεύει και με τρίτες χώρες και χρειάζεται γι' αυτό να υπάρχει σωστή βάση δεδομένων για τη θάλασσα αυτή. Χρειάζονται εδώ επιστημονικά στοιχεία. Ήθελα λοιπόν να πω ότι γι' αυτό δεν συμφωνούμε με την αυτόματη μείωση τον ε, τάξ ε, κατά 25%. Επίσης δεν πιστεύουμε ότι θα ήταν καλή ιδέα να μειώσουμε ανεφόρον ε, τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση μέχρι το 2015. Συμφωνούμε με την απαγόρευση της απόρριψης, γιατί αν λύσουμε το θέμα των απορρίψεων, θα συμβάλλουμε στην μεγαλύτερη υπευθυνότητα των επιχειρηματιών και των δραστηριο... όσων δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να μειώσουμε την γραφειοκρατία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Μιράντα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να απευθύνω στον κύριο Επίτροπο μια ερώτηση που έχει επανεληφθεί και στο παρελθόν. Ε, έχετε επισκεφθεί και την Γαλλική και σας έχουν ξαναθέσει αυτή την ερώτηση σε σχέση με την αναγνώριση της ερασιτεχνικής αλίας. Όπως ξέρετε, η προτινόμενη ε, μεταρρύθμιση της κοινή συλλευτική πολιτικής έχει ως στόχο να ε, διασφαλίσει την αηφόρο αλία και να διασφαλίσει την πρόσβαση στην αλία των διάφορων ειδών, σεβόμενοι του ε, κοινωνικούς και περιφαλλοντικούς και κοινωνικού παράγοντε. Και ε, όμως ε, δεν αναγνωρίζεται η αλία, η ερασιτεχνική, η μικρή, η αλία μικρής κλίμακας και η αλία των θαλάσσιων οργανισμών. Εμείς θα θέλαμε να αναγνωριστεί στο πλαίσιο της πρότασης της νομοθετικής και εγώ είμαι και η συγγήτρια της γνωμοδότησης για την περιφερειακή ανάπτυξη και θα τονιστεί αυτό το θέμα. Η έλλειψη λοιπόν της αναγνώρισης της ερασιτεχνικής αλίας, αν και η κυρία Επίτροπος ε, μας είπε ότι σίγουρα θα αναγνωριστεί μέσω από άλλες έμεσες πολιτικές είναι κάτι ανησυχητικό κατά τη γνώμη μας. Αυτό μας είπε ο κλάδος από τη Γαλλικία πριν 1,5 χρόνο περίπου ε, στην πόλη της Κορούνια υπεγράφει μια δήλωση της Κορούνια που έθεσε την ερασιτεχνική αιλία στην καρδιά της μεταρρύθμισης της κινησιλευτικής πολιτικής και οργανώσεις ε, του κλάδου αλλά και οργανώσεις περιβαλλοντικές ε, δεσμεύτηκαν να αναλάβουν κάποιες κοινέ δράσεις και εκεί αναφερόταν η ιδέα ότι στο μελλοντικό ταμείο για την αιλία να υπάρξουν κάποια μέτρα στήριξης, κάποια βασικά μέτρα και να υπάρχει ένα ελάχιστο κατόφλι έτσι ώστε η αεραστεχνική αλία να προστατεύεται. Θα, η κυρία Επίτροπος ε, στις ε, διαπραγματεύσεις με τα κράτη-μέλη και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα προτείνει μέσα στο Ταμείο να υπάρχει δυνατότητα για ένα ελάχιστο κατόφλι για να υπάρχει αναγνώριση και της αεραστεχνική αλίας. Ευχαριστώ πολύ ο κύριο Αλόνσο από την Βουλή από το Εθνικό Κοινοβούλιο της Ισπανίας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Καταρχήν, ε, μια αξιολόγηση σε σχέση με την ελευτική πολιτική, η οποία έχει φυσικά θετικές στοιχείες, αλλά σε αυτά τα δύο λεπτά δεν ε, μπορώ να τα αναφέρω, θα αναφερθώ μόνο στα αρνητικά. Καταρχήν, εμείς ε, από την σοσιαλιστική ομάδα ε, θεωρούμε ότι το θέμα της κοινωνικής διάστασης στον τομέα της ηλίας ε, δεν έχει καλυφθεί πλήρως στο έγγραφο, όπως πρέπει. Δηλαδή, δεν λαμβάνονται επαρκώς υπόψη και νομίζω ότι με περιορισμένο τρόπο λαμβάνεται υπόψη συνέπειες που μπορεί να έχουν ορισμένα μέτρα. Ξέρουμε ότι υπάρχει τελευταία βελτίωση Όμω, ορισμένα από τα κριτήρια που έχετε συμπεριλάβει θεωρούμε ότι θα έπρεπε να εφαρμοστούν ε, με μεγαλύτερη ευελιξία και με περισσότερο σταδιακό χαρακτήρα για να μην έχουν τόσο αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία και στην απασχόληση σε ορισμένε περιοχέ τη χώρα μα. Έτσι λοιπόν ε, θα θέλαμε να σα ζητήσουμε να σκεφτείτε σε σχέση με την μέγιστη βιώσιμη απόδοση ε, που θα μπορούσε να, να διευρυνθεί η που προβλέπεται αρχικά στα έγγραφα που έχουμε επιτάπητο και σε σχέση με την εξάλληψη των απορρίψεων. Επίσης ε, θα έπρεπε να προσεγγίσουμε το στόχο αυτό, δηλαδή να έχουμε μια πιο σταδιακή εισαγωγή και προς την κατεύθυνση αυτή θα θέλαμε να σας προτείνουμε μια προθεσμία 10 ετών. Πιστεύουμε ότι θα ήταν κάτι λογικό αυτή η προθεσμία έτσι ώστε να μην έχουμε αρνητικέ επιπτώσει. Και τέλος, γιατί δεν έχω χρόνο, σε σχέση με τις ε, μεταβιβάσεις ε, είναι αυτός ένας μηχανισμός, οι μεταβιβάσιμες παραχωρήσεις που θεωρούμε ότι είναι θετικός ε, για την αλία σε μεγάλη κλίμακα αλλά νομίζω ότι είναι προφανές ότι τουλάχιστον στην Ισπανία αυτό είναι ένα σύστημα που αν εφαρμοστεί γενικά θα έθετε σε κίνδυνο την είναι ερασιτεχνική αλεία. Έτσι λοιπόν θέλουμε να σας ζητήσουμε να εξετάσετε τη δυνατότητα να θεσπίσετε μια διαδικασία που να αποκλείει, που να δίνει μάλλον την αρμοδιότητα να αποκλείουν αυτή την αλεία. Ευχαριστούμε κύριος Βίλουγκ από τη Φιλανδία. Mr. Chairman, dear κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Επίτροπε, η Φιλανδία συμφωνεί με τις μασικές γραμμές της πρότασης και χαίρομαι διότι έθεσε η Επίτροπος το θέμα της περιφερειοποίησης, γιατί είμαστε υπέρ εμείς. Πρέπει να διασφαλίζεται ότι η περιφερειοποίηση όμως θα λειτουργεί στην πράξη αυτό είναι το βασικό. Ο κανονισμός, υπ' αυτή την έννοια, θα πρέπει να προβλέπει διακριτική ευχέρεια ώστε τα κράτη-μέλη να αποφασίζουν επιτεχνικών και άλλων θεμάτων διαχείρισης ε, της αλληλεία, λαμβάνοντας υπόψη την άποψη των εμπλεκομένων σε περιφερειακό ε, επίπεδο. Όταν έφυγα από την πατρίδα μου χθες, από τη Δυτική Φιλανδία, ε, υπήρχε πάγος μισό μέτρο στο, στη Βαλτική και μισό μέτρο χιόνι. Οι συνθήκες, θέλω να πω, μπορεί να είναι πολύ διαφορετικές και αυτό θα πρέπει σε κάθε χώρα να λαμβάνεται υπόψη. Τώρα, ίσως ό,τι αφορά τις μεταβιβάσιμες αλληλευτικές εκχωρήσεις, θα πρέπει να επαφίενται να αποφασίζονται από τα κράτη-μέλη και να εφαρμόζουν ε, καλύτερα το σύστημα σε μικρή κλίμακα. Τα TFCs λειτουργήσαν καλά στην αλληλεία μεγάλης κλίμακας, αλλά υπάρχουν και πολλοί αλληλείς ε, που δεν μπορούν να υπαχθούν σε αυτό το καθεστώς. Και η, τώρα η υποχρέωση εκφόρτωσης ή απαγόρευση της απόρριψης. Πώς θα λειτουργήσει το σύστημα αυτό στον ευξηνοπόντο. Είναι ανοιχτό το θέμα. Επίσης αυτή η προϋπόθεση δύσκολα θα λειτουργησει το συστημα αυτο στον πόντο. ειναι ανοιχτο το θεμα επισης αυτη η προυποθεση δυσκολα θα εφαρμοζεται στη μικρή αλία και στη μικρή κλίμακα αλία. Αυτό το πρόβλημα θα πρέπει να λυθεί. Τέλος αλλά πολύ σημαντικό, κάθε άσκοπο πως διοικητικός φόρτος θα πρέπει να καταργηθεί στις μικρής κλίμακας αλία, αλλιώς δεν θα μείνει κανένας αλιέας να δραστηριοποιείται στην ακτή της ε, Φιλανδίας. Ευχαριστώ κυρία Γκαρσία Γέρο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν ε, θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρωτοβουλία και θέλω να καλωσορίσω όλους τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια των κρατών μελών. Πιστεύω ότι τέτοιες ε, συναντήσεις δεν είναι καρποφόρες για όλους. Έχω μία ερώτηση για την κυρία Επίτροπο. Όπως ε, γνωρίζετε, η θέση της Ισπανικής Αντιπροσωπείας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι θετική σε σχέση με τη μεταρρύθμιση, αν και υπάρχουν βέβαια κάποιες αποχρώσεις ε, και ε, εργαζόμαστε επί αυτών για την τελική έκθεση. Υπάρχουν κάποιες ανησυχίες αφενός είναι σαφές ότι ο στόχος είναι ότι πρέπει να υλοποιηθεί αυτή η μεταρρύθμιση και βέβαια πιστεύω ότι σε καμία περίπτωση ε, δεν αναφερθερόμαστε μόνο στο περιβαλλοντικό παράγοντα, αλλά έχουμε και τον κοινωνικό και τον οικονομικό παράγοντα και αυτοί οι τρεις στόχοι αλληλοσυνδέονται για να έχουμε πραγματική ανάπτυξη μιας ε, κοινή ελευτικής πολιτικής. Αν θέλουμε κάτι τέτοιο να είναι δυνατό. Και πρέπει αυτό να ελοπιθεί και με τη συμμετοχή του κλάδου, με το διάλογο με τον κλάδο. Ε, πρέπει να συνεργαστεί και ο κλάδος, διαφορετικά θα έχουμε ε, μια μετα μεταρρύθμιση που θα μείνει στα χαρτιά, κατά τη γνώμη μου. Όμως, ε, για να μην μιλήσουμε για μία ακόμη αποτυχία, ε, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με την πλεονάζουσα ελευτική ικανότητα και πώς θα καταπολεμήσουμε την ε, άναρχη και παράνομη αλία. Επίσης, έχουμε το θέμα της προθεσμίας για την εξάλληψη των απορρίψεων και ξέρετε ότι δεν μπορούμε ε, να έχουμε τις ίδιες προθεσμίες για τη Μεσόγειο όπως έχουμε για την Νορβηγία. το χάρη η Νορβηγία χρειάστηκε 20 χρόνια για πολύ λιγότερα είδη. Έτσι λοιπόν πρέπει να υπάρχει ευελιξία τη στιγμή που θα αναπτυχθούν τα διάφορα μέτρα. Και επίσης ε, μιλάμε και για την ποιότητα, μιλάμε για τον καταναλωτή. Ο Ευρωπαίος καταναλωτής ε, καταναλώνει το 65% ψάρια εισαγωγή ε, και δεν ξέρουμε αν γίνονται σεβαστές οι ίδιες εγγύησει. Ε, και τέλος, για το Ταμείο Χρηματοδότησης, ε, είπατε ότι έχουμε αύξηση 135 εκατομμύρια ευρώ. Όμως, εμένα μου φαίνεται ότι δεν επαρκούν αυτή οι πόροι για μια τόσο φιλόδοξη μεταρρυθμισή και προ αυτή την κατεύθυνση σα ρωτώ, Ποιου άλλου μηχανισμού, γιατί βιώνουμε κρίση, όχι μόνο στον τομέα, αλλά πώς ε, ακριβώς ε, ε, αυτοί οι πόροι θα αντιμετωπίσουν μια κύρια ανησυχία, δηλαδή πώς θα ενισχυθεί η αλία μικρής κλίμακας κυρίες τεχνική αλία και πώς θα έχουν οι αλίες αυτοί περισσότερα μέσα για να μπορέσουν να ζουν αξιοπρεπώς αλλά να μπορέσουν και να διαφυλάξουν και το θαλάσσιο περιβάλλον. Πρόεδρος, θα είναι αδύνατο να μπορέσω να δώσω το λόγο στους υπόλοιπους. Κυρία Ντελόκ από το Γαλλικό Κοινοβούλιο. Σας παρακαλώ σεβαστείτε το χρόνο λεπτά. Euh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, από πλευρά τη Βρετάνη, ε, τη Γαλλία, ε, θα δηλώσω τη διαφωνία μου για την ε, μεταρρυθμιστική σα πρόταση, τουλάχιστον σε μεγάλο μέρο, διότι ακολουθεί φιλελεύθερο προσανατολισμό. Από το 90 στη Γαλλία έχουν, έχει καταρρεύσει ο αριθμό των σκαφών και το ίδιο ισχύει και με του λιμένε. Σήμερα ο στόχο σα είναι να μειώσετε κατά το ίμιση, κατά τα δύο τρίτα, τα σκάφη και του αλληλεί για να επιτύχετε την περίφημη μέγιστη βιώσιμη απόδοση μέχρι το 2015. Μα αυτό που είναι κατεπήγον σήμερα είναι να διατηρήσουμε την ικανότητα του κλάδου ω προς τους ανθρώπους που δουλεύουν στον κλάδο και τα σκάφη για να επιβιώσει, να επιβιώσει η δραστηριότητα. Ε, αντίθετα, εσεί προτείνετε να μειωθεί ο αριθμό των αλλιών, ενώ εμεί θέλουμε να ανανεωθεί ο κλάδος. Και δεν αναφέρομαι καν στα κοινωνικά προβλήματα και στα διάφορα προβλήματα που επιζήρει η απελευθέρωση των αγορών. Σήμερα λοιπόν το πρόβλημα δεν είναι οι υπερβολικέ επενδύσει όπω ίσχυε στη δεκαετία του 80 και του 90. Οι υποεπενδύσει είναι το πρόβλημα για τα σκάφη τα οποία είναι απαρχαιωμένα, δεν είναι, είναι προσαρμοσμένα ω προ την ασφάλεια, το περιβάλλον, τι συνθήκε εργασία, τι ε, σημερινέ απαιτήσει. Ε, με, το ζόρι λοιπόν να ε, επιτύχουμε τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση μέχρι το 2015 σίγουρα δεν είναι η ιδανική λύση. Θέλουν διαφοροποιήσει διαφοροποιημένα μέτρα οι αλληλείς. Αυτό ζητάνε διότι και τα ίδια τα οικοσυστήματα είναι διαφοροποιημένα και έτσι πρέπει να οργανώνεται και η αλληλεία. Θα πρέπει να μιλάμε περισσότερο για τους αλληλείς. Όχι μόνο για τα ψάρια, τους αλληλείς, ε, για την, ε, ε τους κοινούς πόρους, πώς μπορούμε να τους μοιραστούμε, πώς μπορούμε να τους διαχειριστούμε για να τους σώσουμε όλους. Και το οικοσύστημα και τα ψάρια και τους ε, ε Ευχαριστώ. Ευχαριστώ από το Ιταλικό Κοινοβούλιο και το <clears throat> Ε, ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Και σας ευχαριστούμε για την ε, παρουσία σας εδώ, γιατί ε, είναι πολύ σημαντική και σας ευχαριστούμε και για την ειλικρινιά σας ε, γιατί ε, γνωρίζουμε ότι με πολύ μεγάλη ευαισθησία μας ακούτε και απαντάτε πρέπει να είμαστε ίσοι, πρέπει να έχουμε ίσους κανόνες και πρέπει να σκεφτόμαστε ότι ε, ε αν ο ένας πρέπει να ε, επιβληθεί στον άλλο, αυτό θα σήμαινε ότι δεν θα ασκευόμασταν ε, τον πολιτισμό του άλλου και θα έπρεπε και να καταργήσουμε διάφορους τόπους ελίε. όμως ε, θέλουμε να είμαστε ίσοι και για να βελτιώσουμε την προστασία του περιβάλλοντος και τα αποθέματα. Η περιβαλλοντική βιωσιμότητα θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα με την κοινωνική βιωσιμότητα. Θα ήταν μεγάλο λάθος να πιστέψουμε ότι μπορεί η μία προπόθεση να υπερισχύει τις άλλες. Τα ιστορικά αποθέματα θα πρέπει σε περιφερειακό επίπεδο εδώ να γίνονται αντικείμενο και ε, αμέσως θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες τη κάθε περιοχή. Αναφέρομαι στις ε, ε, χώρες της Μεσογείου. Μία από τις ιδιαιτερότητες, το χάρη, είναι να λαμβάνουμε υπόψη την αλία πολλαπλών ειδών και να λαμβάνουμε υπόψη και τις κλιματικές συνθήκες. Θέλουμε να δούμε πώς θα θα ε, βελτιώσουμε τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Ε, καμία διαδρομή που να ε, διαχειρίζεται εντελώ διαφορετικά θέματα σαν ισότιμα δεν μπορούμε να τη σκεφτούμε. Έχουμε ε, την εγκατάλειψη ε, των απορρίψεων είναι κάτι ενδιαφέρον, είναι καινοτόμο, αλλά μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία μόνο για την βιομηχανική αλεία και να ωφελήσει μόνο τη βιομηχανική αλεία. Ε, και δεν θα υπάρχει ιδιαίτερο δυνατότητα για τους μικρούς αλείς και για τα μικρά σκάφη. Πρέπει να αποφύγουμε με τα βάση βασιλευτικές παραχωρήσεις να ε, χρησιμοποιηθούν ε, από τις μεγάλες ε, εταιρείες που όλο και περισσότερο θα τις εκμεταλλεύονται και θα καταστήσουμε καπιταλιστική την αλία. Πρέπει να έχουμε την διαφάνεια και την ετικετοποίηση. Πρέπει να έχουμε τις μεταβάσιμες ελευτικές παραχωρήσεις, αλλά θέλουμε να έχουμε κάπως περισσότερα στοιχεία για να ξέρουμε ξέρουμε πώ όλα αυτά τα στοιχεία θα τα εντάξουμε στην ε, μεταρρύθμιση. Ο κύριο Χάτον από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, e από τη Σκωτία συμφωνώ με πολλά από αυτά που είπε ο Φιλανδός αλλά και ο ε, συνάδελφος από τη Βρετάνη που υπογράμμισε τις γεωγραφικές και άλλες ιδιαιτερότητες και μοναδικότητες που αποτελούν πραγματικότητα στα αλλιευτικά ύδατα και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει μέγιστη αποκέντρωση ως στόχος καθώς προχωρούμε στη μεταρρύθμιση. Βεβαίως αναγνωρίζουμε όλοι ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, την παλαιά εμπειρία της πολιτικής αλληλείας ε, σε κεντρικό επίπεδο η οποία πέτυχε. Επίσης, Καταρχήν τουλάχιστον, και θα εκπλαγείτε με αυτό, συμφωνώ με την προσέγγιση ε, της Βουλής των Κοινοτήτων που προσπαθεί με τις προτάσεις να βρει μια νομική λύση για τα προβλήματα και της αποκέντρωσης μεταξύ άλλων. Βέβαια, ήδη οι νομικοί εμπειρογνώμονες έχουν αμφισβητήσει ορισμένα στοιχεία από την πρόταση που γίνεται. Όμως, ε, είμαστε σε μια παράδοξη θέση αν λέμε, όπως λέμε, ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι με τρόπο που θεωρούμε πρακτικό και εφικτό, πιο λειτουργικό από ό,τι στο παρελθόν, ενώ η κουτή συνθήκη μας δεν μας επιτρέπει να κάνουμε όσα θα θέλαμε. Παράλληλα, με την μεγιστοποίηση της ε, νομικής ερμηνείας των υφισταμένων συνθήκων, θα πρέπει να υπάρξει και η επαρκής πολιτική βούληση, ούτω ώστε με την συναπόφαση να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε πολιτική αλληλείας αποτελεσματική, ε, μια πολιτική για τη διατήρηση, γιατί ε, τα αλλιευτικά κράτη είναι τα πρώτα που θα έχουν να ωφεληθούν από μια τέτοια προσέγγιση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Παπαγεωργίου από το Ελληνικό Κοινοβουλίο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ την κυρία Επίτροπο για την δουλειά που έκανε μέχρι τώρα. Ωστόσο όμως πρέπει να πούμε ότι εμείς ε, ε περιμέναμε μια πιο κοινωνική οπτική στην αναθεώρηση διότι ο τομέας που αποσχολείται, που αποσχολεί τη χώρα μας είναι ένας τεράστιος τομέας και βέβαια ε, μας πρόλαβε η κυρία Επίτροπος για τις επιφυλάξεις που έχουμε, δεν διαφωνούμε με τα τρία ζητήματα που έθιξε. Ωστόσο όμως ε, έχουμε τις επιφυλάξεις μας και στα τρία ζητήματα για την ε, αποτελεσματικότητα αυτών των πολιτικών και για την ολική μέγιστη βιώσιμη ε, απόδοση μέχρι το 2015 και για τις απορρίξεις εφορτώσεις Εδώ θέλω να μείνω κύριε Επίτροπε. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχουμε 17.000 περίπου σκάφη μικρά στη χώρα μας. Έχουμε δεκάδες νησιά. νομίζω ότι θα είναι ατελέσφορο ο έλεγχος, θα χρειαστεί κέντρα διακίνησης ε, εάν δηλαδή ένα σκάφο μικρό βγάζει 5 κιλά ψάρια, θα πρέπει να τα πάει, να ελεγχθούν. Το κόστο αυτού του μηχανισμού ελέγχου πιθανά είναι τεράστιο. Έχουμε ένα πρόβλημα λοιπόν. Επαναλαμβάνω, δεν είμαστε κατά των απορρίψεων επί τη αρχή, αλλά θα χρειαστεί βάσανο και προσπάθεια να δούμε πώ σε κάθε χώρα θα το εξειδικεύσουμε και φυσικά αυτό αφορά και την πολιτική της περιφερειοποίησης. Ε, είναι σωστή η πολιτική μόνο που πρέπει να δούμε τις προϋποθέσεις υλοποίηση, της περιφερειοποίησης για να έχουν αποτέλεσμα ε, αυτές οι πολιτικές οι οποίες επαναλαμβάνω καταρχήν μας βρίσκουν σύμφωνος, διατηρούμε τις επιφυλάξεις, είναι το αντικείμενο, πολύ σωστά και σοφά κυρία Επιτροπή, κυρία Επιτροπή το θέσατε. Ε, δεν είναι τυχαίο και αυτό πρέπει να σας προβληματίσει ότι αυτή είναι η άποψη των περισσότερων και των συνειδημάτων που σας έδεσαν υπόψη. Σας το θέτουμε και εμείς ε, υπόψη σαν ένα προβληματισμό σοβαρό. Θα ήθελα επίσης και να κλείσω για να μην παίρνω από τον χρόνο, να δείτε λίγο στην κατηγορία των υδατοκαλλιεργειών, ιδιαίτερα της λιμνοθάλασσας, ε, κύριε Επίτροπε, πρέπει στον, ε, στον κανονισμό να ληφθεί ιδιαίτερη μέρημνα δίπλα στις υδατοκαλλιέργειες και για τις κλειστές θάλασσες λιμνοθάλασσες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Φερέιρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επίτροπε. Εμείς ε, θα συμφωνήσουμε πολλές από τις επικρίσεις των συναδέλφων ε, σχετικά με το σύνολο των μεταρρυθμιστικών ε, προτάσεων. Πιστεύω ότι ούτως ή άλλως γνωρίζετε τις επικρίσεις. Υπάρχουν δύο βασικά προβλήματα στη μεταρρυθμιστική σας πρόταση. Πρώτον, το ανέφεραν ήδη οι συνάδελφοι, είναι το εξή. Μία αλληλευτική πολιτική δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στην πολιτική διατήρηση των μέσων, των πόρων και των αποθεμάτων. Είναι πολλά περισσότερα από αυτό. Ε, αγνοείται λοιπόν την οικονομική και κοινωνική διάσταση της ε, αλλιευτικής πολιτικής. Ε, δεύτερο σημείο, προσπαθείτε να εφαρμόσετε αυτό το σύστημα των υποχρεωτικών μεταβιβάσεων παραχωρήσεων. Σα κατηγόρησαν ε, ότι είστε φιλελεύθεροι, είπατε ότι εγώ δεν είμαι φιλελεύθερη. Ε, και, κοιτάξτε, αν δεν είστε, το κρύβετε καλά, Επίτροπε. Διότι αυτή η πρόταση που κάνετε ε, διαπνέεται από, μια άκρος φιλε, από ένα άκρο φιλελεύθερο όραμα. διότι χρειαζόμαστε μια πρόταση που θα καλύπτει τι απαιτήσει ε, πραγματικότητα. νομίζω ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να το κάνουν. Χρειαζόμαστε εκβάθρον αναθεώρηση των προτάσεων τη Ευρωπαϊκή επιτροπή Θέλω να σας ρωτήσω τα εξή. Είπατε βάσει των στοιχείων που μας δώσατε ότι 80% ε, των σκαφών ε, θα αποκλειστούν τελικά από αυτό το σύστημα των, μεταβιβάσεων, ε, των μεταβιβάσιμων παραχωρήσεων. Μάλιστα, ω προς τον όγκο των εκφορτωμένων αλλιευμάτων μπορείτε να μας δώσετε στοιχεία. Τι θα γίνει με το νέο σύστημα. Άλλη ερώτηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατίθεται να αναθεωρήσει αυτή την περιοριστική και παραμορφωτική ερμηνεία της κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο ελιευτικός κλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση πέρα από το θέμα του μεγέθους ε, των σκαφών υπάρχει το θέμα της εγκύτητας ε, προς την άκτη, ε, ο αριθμός ημερών εν πλώ, τα, οι αλλιευτικοί εξοπλισμοί, το αν καταναλώνονται νοπά τα ψάρια ή μεταποιούνται, άλλα οικονομικά χαρακτηριστικά του κλάδου κατά την ε, εκμετάλλευση αυτών των αλλιευτικών πόρων. Τι θα συμβεί λοιπόν με αυτό το νέο σύστημα. Θέλω να σα κάνω και άλλε ερωτήσει. Ένα λεπτό, Πρόεδρε, ένα λεπτό. Τελευταία ερώτηση και σταματάω. Η Επιτροπή προτείνει θέσπιση κυρώσεων, να στις πω έτσι, για τα κράτη-μέλη που δεν υποβάλλουν τα δεδομένα που δεν υποβάλλουν τέλος τα δεδομένα όπως ε, θα ήταν υποχρεωμένα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να αυξήσει την συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απόκτηση αυτών των στατιστικών δεδομένων και τι θα γίνει, ε, ποια νέα διάταξη θα ισχύσει με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Θεωρείτε ότι έχετε αποκλειστική αρμοδιότητα, αλλά το κόστος μετακυλίεται στα κράτη-μέλη. Επίτροπε, Κύριε Φεραίρα, νομίζω ότι ξεπεράσατε κατά πολύ το χρόνο σα ε, και έχουμε οκτώ άτομα ακόμα που ζητούν το λόγο. Μάλλον δεν θα προλάβουμε γιατί θα πρέπει να φύγει και η κυρία Επίτροπο και πρέπει να τη δώσουμε και χρόνο να μπορεί να απαντήσει. Ε, θα δώσουμε λοιπόν ε, σε ένα ακόμη συνάδελφο ε, το λόγο και για τους υπόλοιπους αν συμφωνείτε να σας δώσουμε το λόγο κατόπιν, κατά τη διάρκεια των πάνελ. Ο κύριος Σουσικόφσκι από την Πολωνία. Mm, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τώρα, γενικά η πολωνική κυβέρνηση στηρίζει τη μεταρρύθμιση. Υπάρχουν όμως κάποιες λεπτομέρειες ε, που μας ανησυχούν λίγο. Και μιλώ εδώ εξ ονόματος των Πολωνών των πολωνικών οργανώσεων αλλιέων που ανησυχούν με θέματα όπως απαγόρευση των απορρίψεων γιατί πιστεύουμε ότι ναι μεν θα πρέπει να θεσπιστεί αλλά το πρόβλημα είναι πώς θα εξειδικεύσουμε τον τρόπο εφαρμογής ούτω ώστε να στηρίξουμε την παραδοσιακή αλία. Οι μικροί αλίες δεν πρέπει να εξαφανιστούν γιατί αυτή είναι η καρδιά του τομέα. Πρέπει λοιπόν να επιβιώσουν και πρέπει να τους στηρίξουμε. Τώρα, για τα TFC, τις μεταβιβάσιμες αλλιευτικές παραχωρήσεις, και εκεί μπορεί να προκύψουν κάποιες απειλές για τον κλάδο. Δεν πρέπει γι' αυτό πιστεύω να είναι υποχρεωτικές. Και όταν πρόκειται για την ανταγωνιστικότητά μας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, βλέπουμε να ε, εισάγονται νέοι κανονισμοί, και διατάξεις, χωρίς όμως να λαμβάνεται παρκώς υπόψη το θέμα της ανταγωνιστικότητας. Και αυτό σημαίνει ότι χάνουμε μερίδιο διεθνώς. Πρέπει να ακούσουμε περισσότερο τους αλληλείς μας. Ε, η κυρία Επίτροπος επισκέφθηκε την Πολωνία και συνομίλησε με τους αλληλείς μας και γι' αυτό πιστεύω ότι θα λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις μας. Επίσης το θέμα της ε, ε, σήμανσης οι αγοραστές ενδιαφέρονται για την σωστή σήμανση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω λοιπόν ότι τώρα θα ήταν καλό να δώσουμε το λόγο στην κυρία Επίτροπο για να μπορέσει να απαντήσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για αυτή την πολύ αποτελεσματική συζήτηση. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη, καθώς δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο και επίσης θα ακολουθήσουν και παρεμβάσει των εισηγητών. Θα κάνω λοιπόν ορισμένες διευκρίνήσει ε, Καταρχήν βέβαια θέλω να σας ευχαριστήσω για όλες σας ε, τις παρεμβάσεις γιατί ήταν ουσιαστικέ και θεωρώ ότι τα Εθνικά Κοινοβούλια έχουν μελετήσει δεόντως ε, την πρόταση και τώρα έχουμε φτάσει σε ένα οριμοστάδιο να διαπραγματευτούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θέλω λοιπόν καταρχήν να διευκρινίσω ότι πρέπει να εργαστούμε στο πλαίσιο της συνθήκης της Λισαβόνας. Αυτό δεν είναι ένα θέμα ε, να συζητήσουμε εδώ, αν η συνθήκη είναι ανόητη και πρέπει να την ε, τροποποιήσουμε. Φυσικά οι βουλευτές έχουν το δικαίωμα να έχουν τη δική τους άποψη και μπορούν να εργαστούν επ' αυτού. Όμως εγώ θα ήθελα να σας ε, ε παροτρύνω να επικεντρωθούμε στη μεταρρύθμιση. Η μεταρρύθμιση είναι στο πλαίσιο της συνθήκης και καλωσορίζω τις προτάσεις ακόμη και τι αρνητικέ, αλλά στο πλαίσιο τη συνθήκη. Στο πλαίσιο της συνθήκης, ε, όπως σα είπα, εγώ είμαι τη συνθήκη, δεν υποτίθεται ότι εδώ έρχομαι να διαπραγματεύσω τη συνθήκη, αυτό είναι ο ρόλο τη Κομισιόν. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν προσπαθούμε να είμαστε ευέλικτοι, προκειμένου να επιτρέψουμε στα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν ε, ιδιαίτερα διαφορετικέ καταστάσει. Ε, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι έχουμε διαφοροποιημένες καταστάσεις από τη Φιλανδία στη Βουλγαρία ή στην Πολωνία ή στον το Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ιταλία, στη Μεσόγειο. Το κατανοώ αυτό. Αυτή είναι λοιπόν η πρότασή μας. Ε, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με την περιφερειοποίηση και με την αποκέντρωση. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να εξαντλήσουμε τα περιθώρια που μας δίνει η συνθήκη προκειμένου να επιτρέψουμε στα κράτη-μέλη να λάβουν κάποιες αποφάσεις. Ε, υπήρξε λοιπόν μια συζήτηση για τα τεχνικά μέτρα. Αν αυτή η πρόταση υιοθετηθεί, όλα τα τεχνικά μέτρα θα μπορέσουν να εισαχθούν σε περιφερειακό επίπεδο. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη αλλαγή. Ξέρω ότι πολλοί εξημών θα θέλατε περισσότερα, ε, ότι πολλοί εξημών θα θέλατε μια πιο φιλόδοξη πρόταση, αλλά σα παρακαλώ μην υποτιμάτε το τι συμβαίνει υπό τη σημερινή πρόταση, γιατί υπάρχουν το σχάρι όλοι οι κανονισμοί που έχουν να κάνουν με τα τεχνικά μέτρα στη Βαλτική θα εφαρμοστούν και θα εισαχθούν από τα κράτη-μέλη αν φυσικά συμφωνήσουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τι θα συμβεί αν δεν συμφωνήσουν. Αλλά πιστεύω ότι για τη Βαλτική παραδείγματο χάρη Ήδη έχουμε μια καλή κουλτούρα συνεργασίας και μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτή την οδό. Αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για κράτη-μέλη όπως η Γερμανία ή η Πολωνία και κράτη-μέλη όπως η Φιλανδία μπορούν ε, να συζητήσουν ε, και να λάβουν από μόνο τους αποφάσει. Και αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορούμε τώρα να πάμε παραπέρα. Ναι, θα το καλωσόριζα αυτό. Και θα ήθελα να πάμε παραπέρα αν η συνθήκη μας το επιτρέπει. Θέλω να είμαι απόλυτα σαφής γι' αυτό. Έλαβα λοιπόν ήδη την Βρετανική συνεισφορά, όπως ε, ανέφερε, και ε, πρόσωπος ε, της Βουλής των Λόρδων θα ε, προσπαθήσουμε να αξιολογήσουμε αυτήν τη σφορά και αν υπάρχει δυνατότητα θα προσπαθήσω να τη δεκτώ αυτή την πρόταση και επίσης θα προσπαθήσω να δεκτώ όλες τις προτάσεις που μου στέλνετε αν βέβαια είναι συμβατές με τη συνθήκη. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να δώσουμε περισσότερες αρμοδιότητες ε, στα ε, περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια και ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο θα καλωσορίσει αυτή την ιδέα και θα έχουμε και ένα περιφερειακό γνωμοδοτικό συμβούλιο για τον αυξηνοπόντο αν είναι δυνατόν το συντομότερο. Αυτό για την περιφερειοποίηση. Τώρα ας προχωρήσουμε σε ένα άλλο θέμα που είναι πραγματικά επίμαχο και είναι η πλεονάζουσα ικανότητα. Η πλεονέσου ελευτική ικανότητα υπάρχει ή όχι. Υπήρξε μία ερώτηση από ε, το, το μέλος του Γαλλικού Κοινοβουλίου, αν δούμε τη Βρετάνη και την παράκτη Ελία, δεν υπάρχει πλεονάζουσα ικανότητα, αλλά αν ε, συζητήσουμε, κοιτάξτε, ε, έχω πάει εκεί και θα σας πω ότι δεν υπάρχει πλεονάζουσα ικανότητα, αλλά ε, συζητώντα για το γαλλικό στόλο, δεν εφερόμαστε μόνο στην παρακτία αλία. Έχουμε ένα μεγάλο αριθμό γαλλικών σκαφών, τεραστίων σκαφών, ε, που, και ε, εδώ μιλάμε για βιομηχανικό στόλο, δεν μιλάμε για φτωχού ελεί, μιλάμε για στόλο που οικοδομείται, που κατασκευή, που κατασκευάζονται με εκατομμύρια δολάρια χρήματα των φορολογουμένων. Δεν μιλάμε λοιπόν μόνο για του φτωχού ελεί και τα μικρά σκάφη. Σα παρακαλώ, αν ε, πρόκειται παραδείγματο χάρη να εξαιρέσω τα σκάφη μικρή κλίμακα από το σύστημα των παραχωρήσεων, θα εξαιρέσουμε το 80% των σκαφών μα, 80%, αλλά το 60% των εκφορτώσεων θα συμπεριλαμβάνονται στο σύστημα. Γιατί το 60% των εκφορτώσεων ε, ε, λαμβάνονται από το 20% των σκαφών μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν, τι να σας πω, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δεν ε, μπορώ να καταλάβω πώς οι σοσιαλιστές, οι κομμουνιστές, οι φιλελεύθεροι δεν ξέρω ε, πώς δεν μπορούν να καταλάβουν ότι το 20% των σκαφών μας ε, φτάνουν στο ποσοστό του 60% των εκφορτώσεων. Πρέπει να έχουμε μια πολιτική και για αυτούς. Έτσι λοιπόν θα το αντιμετωπίσω. Θα προσπαθήσω να βρω μια ειδική μεταχείριση για τα σκάφη μικρής κλίμακας και μπορούμε να συζητήσουμε μεταξύ μας ποια θα είναι η κατάλληλη μεταχείριση για Αλλά δεν μπορώ να έχω την ίδια μεταχείριση για αυτά τα μεγάλα σκάφη. Αυτή είναι η ιδέα που έχουμε κατά νου. Υπάρχουν. Λοιπόν, εδώ κάποιε συζητήσει. Ποιο είναι ο ορισμό για το small scale vessel, για το σκάφο μικρή κλίμακα. Ε, τώρα είναι σχετικά στενός ορισμός, αφορά το μήκος του σκάφους και το είδος των εργαλείων. Έτσι λοιπόν μιλάμε για 12 μέτρα αλλά όχι για σειρώμενα εργαλεία, μόνο ε, εργαλεία που είναι φιλικά προς το περιβάλλον και είναι επιλεκτικά. Υπάρχουν λοιπόν ορισμένες ιδέες ε, και κάποια θέματα για να έχουμε νέου ορισμούς. Θέλω να σας πω ότι αυτό δεν μπορώ να το υιοθετήσω και θα σας πω γιατί. Καταρχήν χρειαζόμαστε ένα πολύ σαφή ορισμό και που θα είναι εύκολο να τον ελέγξουμε. Παραδείγματο χάρη υπάρχουν προτάσεις να έχουμε κάποιους ορισμούς ε, για την περιοχή αλίας ή για τις αποστάσεις από την ακτή, από την ακτογραμμή. Αλλά πώς μπορούμε να το ελέγξουμε αυτό. Ήδη Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα σε σχέση με την απαγόρευση των απορρίψεων για να το ελέγξουμε και δεν ε, μπορούμε να προσθέσουμε περισσότερες παραμέτρους εδώ. Άλλο πρόβλημα είναι το εξής. Θα η ειδική μεταχείριση και ειδική χρηματοδότηση για τα σκάφη μικρής κλίμακας. Εδώ, υπό αυτούς τους ορισμούς, ε, θα έχουμε αυτή την ειδική μεταχείριση για το 80% των σκαφών μας. Αν θα διευρύνουμε αυτόν τον ορισμό, τότε θα έχουμε το 90% των σκαφών. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε πολιτική. 90% των σκαφών, τίποτα δεν σημαίνει αυτό. Σημαίνει τίποτα. Έτσι λοιπόν πρέπει να σας πείσω ότι πρέπει να εμείνουμε σε αυτόν τον ορισμό. Τι θα γίνει τώρα με τα σκάφη αλίας μικρής κλίμακας. Υπήρξε μία πρόταση να έχουμε κάποια κονδύλια ειδικά για τέτοια μικρά σκάφη. Θα καλωσόριζα μία τέτοια πρόταση από την Επιτροπή, την Περιφερειακή την Επιτροπή, ε, που είναι αρμόδια για την Περιφερειακή Πολιτική, για το Κοινοβούλιο. Αλλά θα πρέπει να το δούμε αυτό και θα πρέπει να το συζητήσουμε με τα κράτη-μέλη, γιατί για να είμαι ειλικρινή μαζί σα, πολλά κράτη-μέλη δεν συμφωνούν με αυτή την ιδέα να έχουμε δική μεταχείριση για την αλληλεία μικρή κλίμακα. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι λοιπόν χρειαζόμαστε ένα περιθώριο ελιγμών και διαπραγμάτευσης. Και σας μιλώ πολύ ανοιχτά. Ε, αυτή είναι η κατάσταση. Εσείς θα αποφασίσετε. Εγώ θα προτείνω τελικά, αλλά εσείς θα αποφασίσετε. Αλλά έτσι εσείς ε, θα λάβετε τις αποφάσεις στην Επιτροπή σας και κατόπιν στην Ολομέλεια για το θέμα αυτό. Θέλω λοιπόν να είμαι απολύτω ανοιχτή, ειλικρινής μαζί σας. Αν υπάρχει καλύτερη λύση, να τη δούμε. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε σκάφη μικρής κλίμακας και έχουμε ειδική μεταχείριση, καλύτερη χρηματοδότηση και καλύτερες ιδέες και μιλάμε για το 80% σκαφών μας. Τώρα, για τις τύψεις, τις μεταβάσιμες ελευτικές παραχωρήσεις, δεν υπάρχει πρόθεση από την πλευρά μας ε, να παρέμβουν εδώ οι τράπεζες. Μιλάμε για τους πλειοκτήτες. Αυτό είναι απόλυτα σαφές. Μιλάμε για τις παραχωρήσεις, ε, μιλάμε για τις κυβερνήσεις ε, και ε, για τους ιδιώτες των και θα δοθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ένα δικαίωμα σε ένα πλειοκτήτη να αυξηση Αυτή είναι η πρότασή μας. Έτσι λοιπόν πρέπει να διαλέξουμε εδώ. Θέλουμε τα κράτη-μέλη να το εφαρμόσουν αυτό όπως θέλουν ή θέλουμε δικλείδες ασφαλείας. Αυτό είναι κάτι που θέλω να συζητήσω μαζί σας και περιμένω τις δικές σας τροπολογίες. Αλλά δεν ε, μιλάμε εδώ για τράπεζα σε καμία περίπτωση. Δεν ε, μιλάμε για ε, για, συγγνώμη για ταμεία. μιλάμε εδώ για πλειοκτήτες και για το δικαίωμα το δικό τους να εμπορευτούν υπό πολύ αυστηρές προϋποθέσεις. Αυτή είναι η πρόταση, αλλά φυσικά τελικά θα δούμε τι θα αποφασίσουν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Σε σχέση τώρα με το άχθος και την γραφειοκρατία, συμφωνώ με όλες τις προτάσεις ε, της γραφειοκρατίας και τα Αν έχετε λοιπόν τροπολογίες παρακαλώ να μου τις στείλετε και ευχαρίστω θα τις δεχτώ. Θα τις υιοθετήσω. Τώρα για τις απορρίψεις. Καταλαβαίνω ότι χρειαζόμαστε μια λογική προθεσμία και μια ρεαλιστική πρόταση. Θα καλωσορίσω τι προτάσει σας. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε μια συμφωνία εδώ. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να εφαρμόσουμε στη Μεσόγειο ε, μια απαγόρευση απορριψίων για τους μικτούς τύπους αλίας. Και να είμαι και εδώ ειλικρινή. Επιτρέψτε μα να βρούμε λύση εδώ. Τι συμβαίνει στη Μεσόγειο, αυτό που συμβαίνει στη Μεσόγειο δεν είναι ότι έχουμε πάρα πολλές απορρίψεις, γιατί έχουμε μεκτό τύπο αλίας ε, σε μεγάλο βαθμό στο ε, Μεσόγειο, εκτός ίσως από τον τόνο. Μιλάμε λοιπόν για μεκτό τύπο αλίας και δεν έχουμε απορρίψει πολλέ. Στι βόρειε θάλασσε έχουμε πολλέ απορρίψει. τι τις στη Μεσόγειο. Εγώ προέρχομαι από τη Μεσόγειο και μπορώ λοιπόν να σα το πω πολύ ανοιχτά. Τρώμε γόνου, ηχθίδια στη Μεσόγειο έχουμε αγορά ηχθιδίων. Τρώμε πολύ μικρά ψάρια. Δεν αφήνουμε τα ψάρια να μεγαλώσουν. Θέλουμε να τα πιάσουμε όταν είναι μικρά. Ηχθίδι, αυτό είναι το πρόβλημα. Έτσι λοιπόν, Γι' αυτό στη Μεσόγειο έχουμε αυτή την ανητική στάση κατά της αποφύγης των απορριψιών γιατί υπάρχει ε, αγορά για τα μικρά καλαμάρια, τα μικρά ψαράκια και αυτό δεν είναι καλό γιατί μεσούσες της κρίσης και όταν τα αποθέματα είναι σε κακή κατάσταση πρέπει να αφήσουμε τα αποθέματα να αναπαραχθούν. Έχουν το δικαίωμα να αναπαραχθούν. Πρέπει να εργαστούμε λοιπόν από κοινού, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα, ναι, να βρούμε ρεαλιστικές λύσει. συμφωνώ, αλλά πρέπει να εργαστούμε από κοινού για να σταματήσουμε αυτή την αγορά εκθηδίων. Εγώ είμαι εδώ και θα καλωσορίσω όλε τι προτάσει που αναφέρονται στου μικρού του από τη Γαλλία, την Ιταλία. Και ήδη πήγα στην Ιταλία και είχα μια πολύ καλή συζήτηση με τον Ιταλό Υπουργό. Ελπίζω ότι το ίδιο θα συμβεί και με του αρμόδιου υπουργού από Ισπανία, Γαλλία. Αλλά σα παρακαλώ, αν βρείτε μια λύση, να τη δω. Και μια τελευταία παρατήρηση για τη χρηματοδότηση και τα κονδύλια. Τώρα, τι προσπαθούμε να κάνουμε με το νέο μέσο χρηματοδότησης. Είναι το εξή. Προσπαθούμε να έχουμε καλύτερη κατανομή των ε, χρημάτων, των πόρων, προκειμένου να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Αυτή είναι η γενική ιδέα. Έτσι λοιπόν δεν λέμε ότι ε, δεν πρόκειται να ξεχρονίσουμε το στόλο μας, θα δώσουμε χρήματα για τον ξεχρονισμό του στόλου, αλλά δεν θα αυξήσουμε την πλεονάζουσα ικανότητα. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα δώσουμε χρήματα για μεγαλύτερες μηχανές, αλλά θα δώσουμε χρήματα για την επιλεκτικότητα των εργαλείων. Και ξέρετε, καταλαβαίνω ότι έχουμε κάποια προβλήματα ε, σε ό,τι αφορά τους ελίς. Θέλουμε να έχουμε καλύτερη κατάρτιση, επαγγελματική κατάρτιση και πρέπει να δώσουμε χρήματα εκεί, αλλά όχι για να έχουμε όλο και μεγαλύτερα σκάφη όπως κάναμε στο παρελθόν. Γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε. Τα χρήματα των φορολογουμένων είναι πολύτιμα και αν δίνουμε όλο ένα και περισσότερα χρήματα, ακόμη και αν δίνουμε όλο ένα και περισσότερα χρήματα, δεν θα περιορίσουμε την πλειονότητα ικανότητα. Γιατί αυτό ήταν το πρόβλημα. Δώσαμε σχεδόν ένα δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία δεκαετία και είμαστε στα ίδια επίπεδα ικανότητα. Ίσως και παραπάνω, λίγο παραπάνω. Πρέπει να βρούμε άλλου τρόπου λοιπόν. Τι θα κάνουμε λοιπόν. θα βοηθήσουμε τους όλους μας να ε, αντιμετωπίσουν αυτή τη μεταβατική περίοδο. Δεν είναι αλήθεια ότι δεν ενδιαφερόμαστε για τους Ελλείς. Ε, Σω να μην είμαι καλή στην επικοινωνία. Ίσως ε, να μην μπορώ να τα πω όπω πρέπει. Αλλά ο βασικό μα κανονισμό, ο κανονισμό για την ετικοθεσία, για τη διάθεση στην αγορά, για την εισαγωγή μεγαλύτερη χρηματοδότηση για τις οργανώσεις παραγωγούς, για διάφορες οργανώσεις, αλλιέ μικρή κλίμακα, όλα αυτά υπάρχουν στην νομοθεσία μας. Ίσως ε, λοιπόν ε, να μην είμαι καλή στην επικοινωνία, σας δώσω ορισμένα παραδείγματα. Φέτος ε, θα δώσουμε στον κλάδο μας 135 εκατομμύρια ευρώ επιπρόσθετα διότι έχουμε φτάσει για κάποια αποθέματα στην μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Αυτό ισχύει για τους αλλήλους στη Μεσόγειο, στη Γαλλία, στη Βαλτική ε, και μιλάμε για τον γάβρο, για τον μπακαλιάρο, για διάφορα ψάρια. Και αυτό δεν έγινε επειδή είναι καλή ή κακή η κακη ή γενναιόδορη τσιγκούνα ή οτιδήποτε συνέβη διότι βελτιώθηκε η κατάσταση. Α συνεργαστούμε λοιπόν για να καταφέρουμε να διανύσουμε την υπόλοιπη απόσταση. Φανταστείτε πόσα εκατομμύρια και πόσε θέσει απασχόληση ε, ε, θα παράγουμε αν συνεχίσουμε να ακολουθούμε αυτό το σύστημα αναβαθμισμένη διαχείριση. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια καλή συνεργασία, ούτω ώστε να βοηθήσουμε του αλληλεί. Ε, ξέρετε από πού έρχομαι, η Μελληνίδα, και ξέρετε ότι η χώρα μου έχει ιδιαίτερα προβλήματα προβλήματα με την κρίση. Φυσικά γνωρίζω την κατάσταση και δεν έρχομαι ως εξωγήινος. Ξέρω πολύ καλά ε, τι αντιμετωπίζουμε και η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερα ε, φαύλο κύκλο. Αλλά ξέρετε, ε, για να διατηρήσουμε την κατάσταση. Αυτό το business as usual το περίφημο δεν είναι το ιδανικό για τους ε, αλληλείς μας. Ε, η διατήρηση της τάξης δεν είναι ιδανική λύση για αυτούς. Πρόεδρε, συζητώ, συγγνώμη, μακρηγόρησα αλλά χρειαζόταν και ελπίζω ότι θα μου υποβάλλετε προτάσεις, ε, τρόπολογίες ε, για οποιοδήποτε επιμέρου στοιχείο του σχεδίου κανονισμού. Ε, ευελπιστώ να έχουμε σύντομα και πάλι την ευκαιρία να συζητήσουμε. Ελπίζω να με προσκαλέσετε και πάλι στο Κοινοβούλιο προτού περατωθεί η πρώτη φάση διαβούλευση με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπο. Λοιπόν, και χωρίς κονοτριβή, να συνεχίσουμε, γιατί όπως βλέπετε δεν έχουμε πολύ χρόνο. Και να περάσουμε στο πρώτο πάνελ για τη μεταρρύθμιση του βασικού κανονισμού. Να δώσουμε το λόγο στην κυρία Λουρίκε Ρόντουστ, η οποία είναι η για το θέμα αυτό. Και όπως είπα, θα έχουμε μια παρέμβαση από την κυρία Ρόντουστ 10 λεπτών και κατόπιν ε, έχουμε περίπου 20 ερωτήσει που έχουν τεθεί για την κυρία Ρόντουστ. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, μάλλον η αποστολή του Πρόεδρου είναι να κόβει χρόνο. Αλλά σα παρακαλώ να προσπαθήσουμε να μην καθυστερήσουμε πάρα πολύ. Έχει το λόγο κύριε Ρόντουστ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, χαίρομαι που βλέπω τόσους ε, εθνικούς εμπειρογνώμονες για να συζητήσουμε για τη μεταρρύθμιση της κοινή αληφτική πολιτικής, η οποία κατά το παρελθόν καθορίζονταν μόνο από την εκτελεστική αρχή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι κυβερνήσει των κρατών μελών από κοινού συνδιαμόρφωναν την πολιτική μας. Δεν είναι μυστικό ότι αυτή η πολιτική δεν είχε ιδιαίτερα επιτυχές αποτέλεσμα. Υπάρχουν πολλά αίτια γι' αυτό. Ένα αίτιο, ένα λόγος είναι ότι οι κυβερνήσεις και ο υπαλληλικό μηχανισμός ίσως ε, να μην θέλουν αλλαγές. Επίσης ε, δεν είναι ε, πολύ, πολύ ε, ευρωπαϊκές κάποιες κυβερνήσεις. Όμως θα πρέπει να έχουμε το γενικό σύνολο υπόψη μας, γιατί τα ψάρια δεν γνωρίζουν εθνικά σύνορα. Χρειάζεται, και γι' αυτό την έχουμε άλλωστε, μια κοινή αλλιευτική πολιτική. Στην Επιτροπή Αλίας εμείς είμαστε έτοιμοι για μεταρρυθμίσεις και θαραλέες, τολμηρές μάλιστα. Η συμμετοχή του Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι μοναδική ευκαιρία λοιπόν για να επεξεργαστούμε μια φιλόδοξη και αποτελεσματική πολιτική. Μόνοι μας δεν μπορούμε όμως. Χρειαζόμαστε συνεργασία ε, με τους εθνικούς βουλευτές. Θα πρέπει όλοι να κινηθούμε προς την ίδια κατεύθυνση. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να ασκήσετε πιέσεις στις εθνικές σας κυβερνήσεις, ώστε οι τελευταίες να μην ακολουθούν μόνο τα εθνικά τους συμφέροντα, αλλά να συμβάλλουν σε μια αποτελεσματική και καλή πολιτική για ολόκληρη την Ευρώπη. Δύο λόγια για την περαιτέρω διαδικασία, την νομοθετική διαδικασία. Αρχές Μαΐου θα επεξεργαστώ το σχέδιο έκθεσής μου ε, με συγκεκριμένες προτάσεις ε, τροποποιητικές στην πρόταση της Κομισιόν. Μετά θα καταθέσουν τροπολογίες οι συνάδελφοι. Ως εισηγήτρια θα προσπαθήσω να βρω καλές συμβιβαστικέ τροπολογίες, να τα συμπεριλάβω όλα. Τον Ιούλιο θα ψηφίσει η Επιτροπή Αλίας. Ε, Ως πρώτο βήμα έχω συντάξει ένα έγγραφο εργασίας όπου παρουσιάζω τις απόψεις μου. Το έγγραφο αυτό αποτελεί την πρώτη βάση συζήτησης. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Θα χαρώ να λάβω παρατηρήσεις, σχόλια, κριτική, ώστε να συντάξω την καλύτερη δυνατή έκθεση. Τέλος θα ήθελα να σας παρουσιάσω τα σημαντικότερα στοιχεία του εγγράφου εργασίας μου. Ε, υποβάλλω 35 συνολικά συγκεκριμένες προτάσεις που αριθμούνται μία προς ε, μία. Ε, τώρα, εις ό,τι αφορά τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές αλλά και φιλόδοξοι. Προτείνω λοιπόν ο στόχος ε, του βασικού κανονισμού να είναι, και να το γράφει αυτό, ότι η βιομάζα των αποθεμάτων θα πρέπει να αυξάνονται σε επίπεδο μέγιστης βιώσιμης απόδοσης. Έχω τροποποιήσει λίγο τη διατύπωση της Κομισιόν. Τα αποθέματα μέχρι το 2015 θα πρέπει να αυξάνονται με βάση τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση όπου είναι βιολογικά δυνατόν, γιατί για κάποια αποθέματα αυτό δεν είναι βιολογικά δυνατό δεν θα πρέπει να θέσουμε ρεαλιστικούς στόχους. Παράλληλα, ο βασικός κανονισμός θα πρέπει να είναι όσο πιο συγκεκριμένος και δεσμευτικός γίνεται. Προτείνω λοιπόν η θνησιμότητα να μειώνεται σε επίπεδο μέγιστης βιώσιμης απόδοσης πάλι μέχρι το 2015. Αυτό θα πρέπει όμως να είναι δεσμευτικό στο βασικό κανονισμό. Το 2015 για τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση ε, είναι εφικτή ε, για όλα τα είδη για όλα τα αποθέματα. Ε, όσο πιο εύκολα έχουμε ανασύσταση, τόσο περισσότερη αλία θα γίνεται. Βεβαίως, τα σκάφη σε μια με, τα βατική περίοδο θα πρέπει να λιεύουν λιγότερο και μάλιστα για κάποια αποθέματα να έχουμε δραστικές μειώσεις. Ε, θα πρέπει γι' αυτό στο μεταβατικό διάστημα να χρηματοδοτήσουμε και να στηρίξουμε τους αλληλείς διότι δεν θα πρέπει κάποιο, κάποια επιχείρηση να κλείσει λόγω των μεταβατικών μέτρων για την ε, απαγόρευση των απορρίψεων. Καταρχήν έχει νόημα να γίνει κάτι τέτοιο, διότι συνολικά θα εκφορτώνονται περισσότερα αλλιεύματα. Δεύτερον, γιατί όλα τα αλλιεύματα θα αφαιρούνται από τις ποσοστώσεις, οπότε θα γίνεται ε, εύκολα μια σωστή διαχείριση των αλλιευμάτων. Τέλος, επειδή τα δεδομένα θα βελτιωθούν πολύ. Θα πρέπει όμως να είναι εφαρμόσιμη η απαγόρευση των απορρίψεων και δεν πρέπει να γίνει αντιπαραγωγική. Προτείνω γι' αυτό λοιπόν η απαγόρευση των απορρίψεων να γίνει σταδιακά με βάση την αλληλεία και όχι τα, ε, είδη. Έτσι λοιπόν με πολυετή σχέδια θα υπάρξει η απαραίτητη προσαρμογή στους κανόνες. Ε, επίσης θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η απαγόρευση των ε, απορρίψεων ε, είναι αντιπαραγωγική. Ε, θα πρέπει να αποδεικνύεται αυτό ως τμήμα της μεταρρύθμισης ή με τη μορφή των κατεξουσιοδότηση πράξεων. Είναι σημαντικό καταρχήν να ισχύει η απαγόρευση των απορρίψεων και μετά με βάση τα επιμέρους είδη και τις επιμέρους μορφές αλίας να υπάρξουν εξαιρέσει, όχι το αντίθετο. Στο έγγραφο εργασίας μου υποβάλλω κάποιες προτάσεις σχετικά με την ρύθμιση της κατανομής των ποσοστώσεων μεταξύ κρατών μελών. Οι προτάσεις αυτές θα πρέπει να είναι το σημείο εκκίνησης μιας συζήτησης. Από κοινού με το Συμβούλιο θα πρέπει να ε, προσπαθήσουμε να βρούμε ένα δικαιότερο αλλά και ε, ρεαλιστικό σύστημα. Πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα τις μεταβιβάσιμες αλλιευτικές εκ ή παραχωρήσεις. Εδώ θα πρέπει να βρούμε ευφυείς λύσεις. Γεγονός είναι ότι υπάρχουν πολλά πιστικά πλεονεκτήματα για ατομικές παραχωρήσεις. Ατομικές, λέω, το λέω αυτό συνειδητά, όχι ατομικές μεταβιβάσιμες εκχωρήσεις. Η τήρηση των, παραχωρή, των ποσοστώσεων από το κράτος μέλος θα ελέγχονται καλύτερα από, το, καλύτερα από το αν υπήρχαν συνολικές ποσοστώσεις για όλο το κράτος. Το κράτος θα πρέπει κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή ε, να κλείσει ε, κάποιες ε, ζώνες αλίας. Και αυτό να γίνεται στην πραγματικότητα. Επίσης υπάρχει το, η άγρα των ψαριών, το race of the fish, γιατί οι αλίες προσπαθούν να αλλιεύουν όσο γίνεται περισσότερο. Ακόμα και κάτω από επικίνδυνες συνθήκες όπως κακοκαιρία. Βγαίνουν τα σκάφη παρόλα αυτά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ατομικές ε, ποσοστώσεις, εκεί μπορεί ο Ελιάς να αποφασίσει ο ίδιος πώς θα αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τις ποσοστώσεις, γιατί η διαπραγματευσιμότητα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Η προσέγγιση μου είναι να πούμε ότι η διαπραγματευσιμότητα θα πρέπει να είναι υποχρεωτική μόνο εκεί όπου υπάρχει πλεονάζουσα ικανότητα και εκεί όπου τα κράτη-μέλη δεν κάνουν τίποτε άλλο για να την μειώσουν την ικανότητα αυτή. Πρώτο βήμα θα πρέπει να ορίσουμε την πλεονάζουσα ικανότητα εκ, νέου. Θα πρέπει να συνδυάζεται, να ισούται με την ικανότητα αλίευσης. Σήμερα η ικανότητα προσδιορίζεται με βάση το, το μήκος του σκάφους και τον κινητήρα του. Η ικανότητα αλίευσης όμως εξαρτάται, για παράδειγμα, και από το, τα αλληλευτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται. Ως δεύτερο βήμα θα πρέπει να αξιολογήσουμε τους αλείς μας. Εκεί όπου υπάρχει μεγάλη πλεονάζουσα ικανότητα θα πρέπει να υπάρχει υποχρέωση μείωσής της. Σε πολλές περιπτώσεις ένα εύκολο μέσο γι' αυτό θα ήταν η εισαγωγή συστήματος TFC μεταβάσιμων αλληλευτικών εκχωρήσεων. Αν το κράτος μέλος αποδείξει ότι την μείωση της πλεονάζουσας ικανότητας την επιτυγχάνει χωρίς μεταβιβάσιμες εκχωρήσεις, πρέπει ε, ε, να λαμβάνεται αυτό υπόψη. Ε, θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να μην υποχρεωτικό το σύστημα μεταβάσιμων εκχωρήσεων, αλλά υπό την προϋπόθεση μόνο ότι θα αξιολογούνται οι ε, ικανότητες και όπου συνιστούν πρόβλημα θα πρέπει να γίνεται πραγματική μείωσή τους. Ένα άλλο πρόβλημα είναι η περιφερειοποίηση. Εδώ έχουμε πολιετή σχέδια. Για να επιτευχθούν οι στόχοι της κοινή αλληλευτικής πολιτικής χρειάζεται βελτιωμένη ε, ένταξη των εμπλεκομένων και των ενδιαφερομένων ε, στον τομέα. Πρέπει λοιπόν να πούμε ότι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να συμμετέχουν στην επεξεργασία μιας πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πολιετές σχέδιο τα πρώην ε, τα ΡΑΚ, τα Περιφερειακά Γνωμοδοτικά Συμβούλια πρέπει να παίξουν μεγαλύτερο ρόλο. Προϋπόθεση όμως είναι η σύνθεσή τους να γίνει πιο αντιπροσωπευτική. Ε, οι εργαζόμενοι, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, η παραγωγή πρέπει να συμμετέχουν. Η επιστημονική επικούρηση των γνωμοδοτικών συμβουλίων πρέπει να βελτιωθεί. Τα κράτη-μέλη πρέπει να υποχρεωθούν όταν εγκρίνουν εθνικά μέτρα, όταν θεσπίζουν εθνικά μέτρα θα πρέπει να συνεργάζονται με αυτά. Αυτή η συνεργασία μπορεί να συντονίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ως Επιτροπή θα ε, αναθέσουμε στη νομική μας υπηρεσία να εξετάσει πάλι πώς και αν μπορούμε να προχωρήσουμε στην περιφερειοποίηση. Γιατί πιστεύω ότι ε, πολλά μπορούν να αποφασίζονται επιτόπου στις παράκτιες ε, περιοχές μας. Δεν χρειάζεται να τα ρυθμίζουν όλα οι Βρυξέλλες. Το έγγραφο εργασίας έχει και ένα πρόσθετο κεφάλαιο για την Μεσόγειο και τον Εύξηνο Πόντο. Επειδή η κατάσταση εδώ διαφοροποιείται από ε, την υπόλοιπη Ευρώπη, τα αποθέματα ηχθείων σε μεγάλο βαθμό ε, ψαρεύονται με παράκτη αλία. Λίγα αποθέματα είναι αυτά τα οποία αλλιεύονται από πολλές χώρες ταυτόχρονα και η δομή του στόλου διαφέρει από εκείνη του Ατλαντικού και της Βόρειας Ευρώπης ε, γιατί είναι μικρότερης κλίμακας. Σαφώς. Η μεταρρυθμιστική πρόταση εδώ θα πρέπει να βελτιωθεί. Θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένα μέτρα πρόσθετα για τη Μεσόγειο. Για παράδειγμα, υποχρέωση να υπάρχει δίκτυο για τις κλειστές περιοχές για την αλληλεία. Επίσης χρειάζεται μια πιο φιλόδοξη πολιτική για ε, τη βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια και την πρόθεσή της. Τέλος θα ήθελα να πω ότι ε, συμφωνώ με τους προηγούμενους ομιλητές σχετικά με τη μικρή αλληλεία, τη μικρής κλίμακας. Θα πρέπει να την λάβουμε υπόψη μας περισσότερο. Γι' αυτό χρειάζεται νέος ορισμός. Τι είναι λοιπόν αυτή η μικρή κλίμακας αλληλεία. Στο έγγραφο εργασίας μου, ε, στην ε, πρόταση 22, λέω ότι ο ορισμός της μικρής κλίμακας αλληλείας πρέπει να βελτιωθεί και να συμπεριλάβει άλλα κριτήρια από το μήκος των σκαφών όπως για παράδειγμα το μέγεθος της επιχείρησης ή το τζίρο. Ε, ανασκάφος. Ε, τα βασικά κριτήρια θα πρέπει ε, να είναι τα ίδια για όλα τα κράτη-μέλη. Προσβλέπω με χαρά στις απόψεις σας και προφορικά εδώ και γραπτός γιατί θα με διευκολύνει στην περαιτέρω εργασία μου και βεβαίως θα σας συναντήσω και στο μέλλον. Πολλούς από εσάς τους καλωσόρισα και στο γραφείο μου και θα χαρώ να δω και περισσότερους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ρόντουστ και να περάσουμε τώρα στις ερωταπαντήσεις. Και σας επαναλαμβάνω θα είμαι πολύ αυστηρός με το χρόνο. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Λάρσον από το Σουηδικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν να πω ότι υποστηρίζουμε την Επίτροπο και την πρότασή της Έχουμε πάνω από 80 από θέματα τα οποία είναι αντικείμενο υπερελίευση και πρέπει να το αλλάξουμε αυτό. Κανεί δεν μπορεί να στέκεται σε τρία πόδια ταυτόχρονα. Έτσι λοιπόν πρέπει να θέσουμε κάποιε προτεραιότητε. Καταρχήν λοιπόν πρέπει να δούμε τι οικολογικέ, τι βιολογικέ πτυχέ και κατόπιν πρέπει να δούμε ε, και το κοινωνικό και οικονομικό κομμάτι. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να το δούμε αν δεν υπάρχουν ε, ψάρια στη θάλασσα. Καταρχήν πρέπει να δούμε λοιπόν το θέμα τη οικολογική ηλικίας μέχρι το 2015 ε, θα ήταν ε, καλό να έχουμε βιώσιμα αποθέματα τα οποία θα είναι ένας ε, καλός τρόπος υλοποίησης της αλίας. Δεν μπορούμε βέβαια απλώς να, να κάνουμε ευχολόγια εδώ, πρέπει να είμαστε σαφείς. Και Νομίζουμε ότι ορισμένα θέματα είναι εθνικά ζητήματα και συμφωνώ με την κυρία Ρόντουστ και με τον τρόπο που προτίμασε ε, το έγγραφο της. Νομίζω ότι το... η απαγόρευση των ε, απορρίψεων ε, είναι κάτι θετικό. Δεν θα πρέπει να έχουμε παρεμπιπτόντα αλλιεύματα και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις για τα παρεμπιπτόντα αλλιεύματα που εκφορτώνονται. Σας ευχαριστώ ο κύριος Πίρκερ Χουβά από την Αυστριακή Βουλή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, κυρία συνάδελφε Ρόντουστ, σας ευχαριστώ θερμά και σας συγχαίρω για το έγγραφο εργασίας. Ως ε, περίκλειστη χώρα που καταναλώνει όμως ψάρια, θεωρούμε ότι είναι σημαντική μια κοινή προσέγγιση ιδιαίτερα εις ό,τι αφορά τη διατήρηση της βιομάζας μέχρι το 2015. Είμαστε πεπισμένοι, όπως, και, όπως είπε και η Επίτροπος Δαμανάκη, μήπως δεν με ακούτε. Ε, ναι, ε, πρέπει να επιτύχουμε και να διατηρήσουμε αυτούς τους στόχους. Πιστεύω ότι θα ήταν όμως έξυπνο ε, αυτό το biologically possible ε, αυτό το βιολογικά εφικτό να μην σημαίνει ότι οι στόχοι μας θα υπονομευθούν. Θα πρέπει να έχουμε σχέδια διαχείρισης για κάθε είδος, αλλά να διατηρήσουμε το στόχο του 2015. Αυτό είναι σημαντικό. Επίσης συμφωνούμε με τη μείωση της ε, πλεονάζουσας ικανότητας και εδώ προτείνουμε στο μέτρο 18 να προσθέσουμε μια, ε, ένα χρονοδιάγραμμα, μια καταληκτική ημερομηνία για, τον, για την προσαρμογή των στόλων. Είναι σημαντικό να έχουμε χρονοδιαγράμματα, ούτω ώστε να επιτευχθούν αυτή τη φορά όντω οι στόχοι μα. Για τι παρατηρήσει σα τώρα, για τη μικρή κλίμακα αλληλεία, ε, ναι, συμφωνώ, γιατί αυτοί παράγουν ποιοτικό προϊόν στις μικρές επιχειρήσεις τους και στην Αυστρία ως καταναλωτές. Θέλουμε να εξακολουθήσουμε να έχουμε αυτά τα προϊόντα ποιότητα στα υποδειγματικά στην ε, κατανάλωση. Τέλος, για την οδηγία για, την συνεπή, για τα συνεπή διαφανή αποτελεσματικά κριτήρια για την υδατοκαλλιέργεια είναι πολύ σημαντικά και τα στηρίζομαι γιατί παίζουν σημαντικό ρόλο και θα είναι ακρογωνιαίος λίθος πραγματικά τα μέτρα αυτά για το μέλλον της Αλίας. Ευχαριστώ κύριο Μιλάν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δύο λεπτά. Έχω δύο πράγματα θα πω κάτι που δεν υπάρχει κατά την άποψή μου και κάτι που δεν λειτουργεί. Αυτό που δεν υπάρχει σε αυτή τη μεταρρύθμιση λείπει θάλασσα. Μιλάμε για τους αλείς, για τα ψάρια, για τα μέσα, για τους στόχους, αλλά δεν μιλάμε για τη θάλασσα. Εγώ πιστεύω ότι δεν ε, πρέπει να βάλουμε το χέρι στη θάλασσα, δηλαδή πρέπει να εγγυηθούμε ε, ότι η θάλασσα παράγει περισσότερο. Αυτή είναι μια οικοσυστημική προσέγγιση και όχι ε, αποκλειστικά μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Δεν υπάρχει ούτε μία λέξη και νομίζω ότι πρέπει το Κοινοβούλιο να κάνει κάτι γι' αυτό. Δηλαδή να πούμε κάτι έτσι ώστε να δημιουργήσουμε συνθήκες να παράγει περισσότερο η θάλασσα. Παραδείγματο χάρη, μπορούμε το χρόνο που δεν γίνεται ελεία να τον μεταφράσουμε σε χώρο όπου δεν υπάρχει αλεία. Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο ε, επόμενο περιοχών σε όλες ε, τις ευρωπαϊκές ακτές και μπορούμε με έναν τέτοιο τρόπο όπως ο Κοπέρνικος να αλλάξουμε τη φιλοσοφία μας. Ε, θεωρώ ότι αυτό λείπει σήμερα σε αυτή τη μεταρρύθμιση. Τώρα αυτό που δεν λειτουργεί και είναι το δεύτερο θέμα που θέλω να αναφέρω ε, είναι κάτι που δεν αποδεικνύεται σε καμία περίπτωση ότι το να εισαγάγουμε την αγορά ε, των μεταβιβάσιμων παραχωρήσεων οδηγεί σε μείωση της ελευτικής προσπάθειας. Βλέπετε, είναι μια απόπειρα αυτή. Αλλά αυτή η απόπειρα, έτσι όπως αναφέρεται, εκεί όπου έγινε, είχε δραματικά αποτελέσματα και μάλιστα υπήρξε μεγαλύτερη αύξηση με τη συγκέντρωση και δημιουργήθηκε μία άρνηση της ιστορίας, του πολιτισμού, της παράδοσης, του κοινωνικού αντικτύπου ε, στα πλαίσια της Ελίας. Ε, και έτσι λοιπόν κανένας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας δίνει απάντηση εδώ και μήνες. Ε, αν μπορούμε να δούμε αν θα υπάρχει πραγματικά όφελος από αυτές τις μεταβάσιμες ηλεκτρικές παραχωρήσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ο κύριος Γκαρσία και τρεις ε, ερωτήσεις κύριε Ρόντους. Για το πρώτο θέμα, για τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, θα επιμείνω ε, για μια ακόμα περισσότερο σε όσα υπόθηκαν και από άλλους ομιλητές. Μας φαίνεται ότι να θέσουμε τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση στο 2015 είναι κάτι αδύνατο να γίνει αν δεν υπάρχει δραστική ε, θυσία όλων των κοινωνικο-οικονομικών στοιχείων στην Ευρώπη. Έτσι λοιπόν μα λοιπόν, μας ε, φαίνεται ότι δεν θα έπρεπε να θέσουμε το στόχο αυτό νωρίτερα από το 2020 όπω έχουμε και στη συμφωνία του Johannesburg. Και στη δική μα κοινοβουλευτική ομάδα τράβηξε την προσοχή η πρόταση κανονισμού γιατί δεν αναφέρεται σε κανένα άρθρο ή δυνατότητα τη διαχείριση τη ελευτική προσπάθεια. Αν θέλουμε να πετύχουμε συγκεκριμένου στόχου, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, αυτό δεν θα επιτευχθεί με τη συμπερίληψη ενό συστήματο. Ε, μεταβιβάσιμων ελευτικών δικαιωμάτων. Κάτι τέτοιο μπορεί να ισχύει μακροπρόθεσμα, όχι βραχυπρόθεσμα. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό όμω να συμπεριλάβουμε την έννοια τη ελευτική προσπάθεια. Και θεωρείτε λοιπόν, πρώτη μου ερώτηση, ότι είναι απαραίτητο να βάλουμε τον έλεγχο τη ελευτικής προσπάθεια μέσα στα μέτρα του άρθρου 7 της πρώτης κανονισμού. Σε ό,τι αφορά τις απορρίψεις ε, δεν θα πω κάτι παραπάνω γιατί ήδη υπόθηκαν αρκετά. Χαίρομαι που είναι σταδιακή η εφαρμογή, ελπίζουμε να γίνει και στην πράξη και τέλος ε, για τα ITQs, ε, για τις ατομικές μεταβιβάσιμες ποσοστώσεις. Δεν συμφωνούμε με την πρόταση της Κομισιόν να περιορίσει την μεταβίβαση μεταξύ κρατών μελών. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να σεβόμαστε τους ε, κανόνες της ενίας αγοράς. Δεν μπορούμε να διατηρήσουμε ε, αυτές τις διακρίσεις ε, που υφίσταται ο τομέα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην υπάρχει δηλαδή ελευθερία της εγκατάστασης λόγω της εθνικότητας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Γκαρσία. Κυρία Έρμπιου από το Γαλλικό Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούν ε, για τα περιβιώσιμη ε, αλίας, αλλά υπάρχει και η κοινωνική και η οικονομική διάσταση, το οποίο δεν μπορούμε να παραγνωρίζουμε. Για να επιτύχουμε την ε, βιώσιμη αλία χρειαζόμαστε καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στους πολιτικούς, δηλαδή τους επιστήμονες και τον κλάδο κάθε χώρα. Θα συμφωνήσω με αυτά που έλεγε ο συνάδελφος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι χρειαζόμαστε μια πιο οικοσυστημική προσέγγιση, δηλαδή χρειαζόμαστε ένα νέο πρότυπο οικοδόμησης τεχνογνωσίας που θα βασίζεται σε στενή διαβούλευση ανάμεσα στον κλάδο και στους ερευνητές. Ξέρουμε ότι πολλές περιοχές της Ένωσης έχουν ήδη συμμετάσχει στη συλλογή ε, των στατιστικών στοιχείων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλουμε λοιπόν να προωθήσει αυτήν την κοινή τεχνογνωσία ούτως ώστε ε, να συλλέγονται συστηματικά και τακτικά τα στατιστικά δεδομένα και να αναπτυχθεί επαγγελματική συνείδηση στον κλάδο. Ω προ ε, του ερευνητικού στόχου έχει ήδη σημειωθεί πρόοδο σε τοπικό επίπεδο, όπω στη χώρα μου παραδείγματο χάρη. Οι επιστήμονε ε, που είναι δίπλα ή και ακόμη και εν πλώ συμβουλεύουν, ε, συμβουλεύουν συγγνώμη, του αλληλεί και είναι αξιόπιστα τα επιστημονικά δεδομένα που προκύπτουν από αυτό. Ε, τώρα, οι διάφορε πρωτοβουλίε που έχουν αναλυθεί έχουν επιδρέψει μια μετριοπαθή προόδο, η οποία όμως είναι χαρακτηριστική ε, για κάποιες περιοχές και για κάποια αποθέματα. Ζητάμε μείωση των απορρίψεων, βεβαίω, αλλά δεν θα πρέπει να είναι ε, μηδενική απόρριψη. Σίγουρα δεν πρέπει ε, ε, η λύση αυτή να υλοποιηθεί νυχθημερών. Θα πρέπει να είναι και σταδιακή και στοχευμένη η προσέγγιση μας. Οπότε θα ήθελα να ρωτήσω, προβλέπετε μία εις βάθος ανάλυση αντικτύπου, γιατί θεωρώ ότι είναι απαραίτητο. Επίσης θα πρέπει να μελετήσουμε τα περί επιλεκτικού εξοπλισμού, επίσης της χωροταξίγης προσέγγισης αλίας, δηλαδή ανά και ε, ε, ε, θα πρέπει να έχουμε ομοιόμορφα κριτήρια για να ταξινομούμε τα σκάφη και όπως λένε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε κυρία Λοβίν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα τώρα να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών σε σχέση με αυτήν την μεταρρύθμιση. Τι περιμένουν, λοιπόν, ε, θέλουν υγιή ψάρια που δεν πάσχουν από τον ευτροφισμό των ε, υδάτων ε, γιατί έχουμε, έχουν πληγεί τα οικοσυστήματα. Χρειαζόμαστε λοιπόν υγιείς θάλασσες για να έχουμε υγιή ψάρια. Μιλάμε για αυτάρκεια που ζητούν οι καταναλωτές. Μα, συγγνώμη, εισάγουμε πάνω από 60% των ψαριών που καταναλώνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ευρωπαϊκό στόλο αλλιεύει ανά τον κόσμο για να προμηθεύει την αγορά. Μπορούμε να επιτύχουμε πολύ μεγαλύτερη αυτάρκεια. Επίσης, ε, θέλουμε έναν οικονομικά βιώσιμο κλάδο. Ε, και δεν θα συμβεί αυτό μόνο αν ε, ανακτήσουμε τα αποθέματα. Θα πρέπει για να επιτύχουμε αυτού του τρει στόχους να κάνουμε μία ε, εκβάρθων αναθεώρηση της ε, πολιτικής. Θα πρέπει να εμείνουμε σε αυτό το στόχο της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης για το 2015 γιατί είναι ο καλύτερος τρόπος που έχουμε στη διάθεσή μας. Ε, ισχυρίζονται κάποιοι ότι δεν είναι δυνατό, δεν είναι εφικτό αυτό μέχρι το 2015. Μα δεν αληθεύει αυτό. Μπορούμε να έχουμε στόχου ω προ ε, την ε, θνησιμότητα, θνησιμότητα των ψαριών και να έχουμε την FMSY, την περίφημη, δηλαδή μέχρι τη βιώσιμη απόδοση που βασίζεται στη θνησιμότητα των ψαριών. Αυτό μέχρι αύριο μπορούμε να το επιτύχουμε. αλλά Καταλαβαίνετε ότι άμα παίρνουμε 80% των γεννητόρων ε, από την βιομάζα, ε, δεν μπορούμε να επιτύχουμε το στόχο. Αύριο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη θνησιμότητα των ψαριών κριτηρίων, να ρίξουμε αυτό το ποσοστό στο 25%. Χρειαζόμαστε ένα υγιή κλάδο, υγιή θάλασσε και ε, έτσι οι καταναλωτέ θα έχουν υγιή και σήμερα και στο μέλλον. Το χρωστάμε αυτό στι μελλοντικέ γενιέ. Α μην αποκλίνουμε από τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Σα παρακαλώ, σα ευχαριστούμε κυρία Κύριε από το Ιταλικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Θέλω όμως να κάνω μια σημαντική εισαγωγή. Θεωρώ ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για περιβαλλοντική εφορία αν ε, δεν ε, συμβαδίζει ο σεβασμός του περιβάλλοντος με το σεβασμό των αλλιέων. Ε, νομίζω ότι πρέπει να σεβόμαστε και τους αλλιείς και τις οικογένειές τους που ζουν από αυτή τη δουλειά. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ σε κάποια ουσιαστικά σημεία. Εμείς είμαστε εντελώ αντίθετοι στο σημείο των μεταβιβάσιμων παραχωρήσεων γιατί θεωρούμε ότι στη Μεσόγειο αυτό το σύστημα δεν μπορεί να εφαρμοστεί και επίσης ε, θα πρέπει ε, να σχετίζεται με μια ε, ποσότητα αλίας που θα πρέπει να προσθεί έτσι λοιπόν επειδή στη Μεσόγειο ισχύουν ιδιαίτερες προϋποθέσεις θα πρέπει το κράτος μέλος να μπορεί να υιοθετεί το σύστημα κατά τη δική του διακριτική ευχέρεια και να αναφερθώ και στην αλία μικρής κλίμακας που είναι νομίζω το δύνατο σημείο χίλιο πτέρνα όλης της μεταρρύθμισης γιατί δεν μπορούμε να αναφερόμαστε είμαστε στην ε, μικρή αλία και αναφερόμαστε μόνο στα 12 μέτρα μήκους του σκάφους. Πρέπει να λαμβανούμε υπόψη και άλλες παραμέτρους και πρέπει να επιτρέψουμε στα εθνικά κράτη να εφαρμόσουν μέτρα κοινωνικής επόσβεσης σε περιόδους κρίσης. Έτσι λοιπόν δεν θα πρέπει να επιδεινώσουμε ακόμη περισσότερο την κατάσταση του κλάδου από επαγγελματική σκοπιά. Και επομένω θέλω να υπερασπίσω να μην διακόψουμε την δημόσια στήριξη στον τομέα ε, κυρίως αναφέρομαι στη συνεισφορά ε, των παροπλισμών ε, Εμεί θεωρούμε ότι θα έπρεπε να έχουμε κάποια πολιετή σχέδια διαχείριση όπω προβλέπεται από την ΚΑΛΠ. Πρέπει λοιπόν με χρήματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίζουμε την χρηματοδότηση στα πλαίσια εθνικών προγραμμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος ε, Γκάμπριελ ε, Γαβρίλ από την Κύπρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για την Κύπρο η στήριξη της αλίας μικρής κλίμακας είναι ουσιώδες ζήτημα. Για την επίτευξη των στόχων της νέας κοινή αλληλευτικής πολιτικής είναι απαραίτητη η ανάληψη παρόμοιων μακροπρόθεσμων δεσμεύσεων και από τα γειτονικά κράτη και τους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περίπτωση της Μεσογείου, πώς θα εξασφαλίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την ανάληψη παρόμοιων μακροπρόθεσμων δεσμεύσεων από τους μεσογειακούς εταίρους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Γκάλαγκερ από το Κοινοβούλιο. Uh, uh, Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα μακρηγορήσω. Είναι πολλές οι ερωτήσεις και λίγος ο χρόνος με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Κάποια θέματα θα θέσω. Η Επιτροπός δεν είναι εδώ. Ίσως η κυρία Ρόντους θα το σκεφτούν. Ε, ε, υπάρχουν κάποια προβλήματα με την μεταρρύθμιση. Γιατί πρέπει να βοηθήσουμε αυτούς που θα χάσουν θέσεις εργασίας. Όπως όλοι στην Ιρλανδία, είμαι κι εγώ εντελώς κατά των μεταβιβάσιμων ποσοστώσεων. Είναι εθνικός πόρος και επουδενή δεν μπορούμε να τον πουλάμε ή να τον μισθώνουμε ε, για 15 χρόνια. Μπορεί να το μην το πάρουμε πίσω ποτέ θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι αν συμβεί αυτό, και πάλι ελπίζω να μην συμβεί, τι προστασία θα έχουν τα πληρώματα. Παλιά στην Ιρλανδία είχαμε κάνει παροπλισμό και έχασαν τα πληρώματα, τη δουλειά τους, απολύθηκαν και τέρμα τέλος. Θα πρέπει λοιπόν να το λάβουμε αυτό υπόψη μας στον κλάδο. Επίσης τα τελευταία χρόνια σε όλα τα κράτη-μέλη μας είδαμε τον αριθμό μικρών λιμανιών που έχουν αποδεκατιστεί, το, ε, ε, ε, το, είδαμε τα μικρά λιμάνια να αποδεκατίζονται. και αυτή ίσως είναι ερώτηση στον κύριο Πιστεύω ότι θα πρέπει να περιχαρακώσουμε τα μικρά λιμάνια που αλλιώς δεν θα επιβιώσουν και όσους δραστηριοποιούνται εκεί. Ε, μπορεί να υπάρξουν κάποια σχέδια που να αφορούν τη θάλασσα, τους ε, ε, ναυτικούς, αλλιώς θα χαθούν. Τέλος, πολλές φορές διστάζομαι να μιλήσουμε για την καταστροφή από τις φώκες που καταναλώνουν 20-40 κιλά ψάρια την ημέρα. Μιλάμε για βιώσιμη αλία και φοβόμαστε να μιλήσουμε για το ζήτημα αυτό. μιλάμε για τις απορρίψεις ε, που βεβαίως βρίσκουν αντίθετους ε, πολλούς αλλά ας δείξουμε το θάρρος να μιλήσουμε και για τις φώκες που θα επηρεάσουν την ε, μέγιστη βιώσιμη απόδοση εάν αντιμετωπιστούν με μέτρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Δαμανάκη και, την κυρία Ρόντους για την ειλικρίνειά τους. Στο Φλαμανδικό Κοινοβούλιο είμαστε υπέρ της βιώσιμης αλίας και θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχουν δυνατότητες εξαιρέσεων βέβαια ε, στα πλαίσια της, πολιτικής, της κοινής πολιτικής αλίας. Τώρα για την καταληκτική του 2015 δεν υπάρχουν αρκετά επιστημονικά δεδομένα και επίσης πρέπει να βεβαιωθούμε ότι θα έχουμε τα απαραίτητα επιστημονικά στοιχεία στη διάθεσή μας που θα αφορούν την ποσότητα της αλίευσης. Οι απορρίψεις, ναι, πρέπει να μειωθούν και το σύστημα των ποσοστώσεων θα πρέπει να προβλέπει κάτι για τη μεικτή αλληλεία. Γιατί αλλιώς στο Βέλγιο αυτή η αλληλεία δύσκολα θα διατηρηθεί. Τώρα, για την ανασύσταση των αποθεμάτων ψαριών. Δεν συμφωνούμε με τις μεταβιβάσιμες αλλιευτικές παραχωρήσεις, γιατί δεν νομίζουμε ότι έτσι θα αντιμετωπιστεί η πλεονάζουσα ικανότητα του αλλιευτικού στόλου με τον καλύτερο τρόπο, γιατί είναι μεγαλύτερο το κόστος ε, ε, και δυσκολεύονται οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά οι παραχωρήσεις αυτές θα καταλήξουν σε ελάχιστα χέρια σε τελευταία ανάλυση. Εμείς έχουμε μικρό αλλά δραστήριο στόλο στο Βέλγιο και υπάρχουν τρία περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια. Ε, οπωσδήποτε αν ισχύουν διαφορετικοί κανόνες ε, δεν θα υπάρξει απλούστευση Πώς θα δημιουργήσουμε ίσους κανόνες ε, συμμετοχής αν έχουμε διαφορετικούς κανόνες. Και ε, σε ό,τι αφορά την εξωτερική διάσταση, συμφωνούμε με την άποψη της Επιτρόπου σε αυτό το θέμα. Η κυρία από το Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την εισηγήτρια κυρία Ρόντους για το έγγραφο εργασίας της. Ε, με το οποίο συμφωνώ σε πολλά σημεία, ιδιαίτερα εις ό,τι αφορά τη μείωση της πλεονάζουσας ικανότητας και την εισαγωγή των μεταβιβάσιμων αλλιευτικών ε, δικαιωμάτων. Τώρα, για την απαγόρευση της απόρριψης, αντί για την προσέγγιση της Κομισιόν με βάση τα είδη, πιστεύω και εγώ ότι πρέπει να προχωρήσουμε με βάση τον τύπο της αλληλείας. Θα πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσεις για την αλληλεία ε, όπου επιβιώνουν ε, πολλές απορρίψεις όπως στα καβούρια, σε μας ε, ή σε άλλα είδη στη Βαλτική. Τώρα, για την πρακτική εφαρμογή, η απαγόρευση της απόρριψης δεν πρέπει να σημαίνει ότι θα εξαλειφθούν κάποια είδη αλληλεία στη Βαλτική, για παράδειγμα, σε σχέση με τις και στα πλαίσια των μειωμένων ποσοστώσεων. Τώρα, γιατί πρέπει ε, ε, γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσεις. Επίσης, η μικρή κλίμακα αλληλεία, αυτό το θέμα δεν λαμβάνεται παρκώς υπόψη στην πρόταση. Ε, ιδιαίτερα ε, όταν πρόκειται για σκάφη κάτω από 12 μέτρα και ε, συγκεκριμένο αλλιευτικό εξοπλισμό. Σε ό,τι αφορά τη διατήρηση της παράκτειας αλίας, εδώ χρειάζονται καλύτερες προτάσεις αλλά και μέτρα προώθησης. Σημαντικό είναι για μας και το θέμα το τελευταίο της περιφερειοποίησης. Το one fits all, ένα μέτρο για όλους δεν μπορεί να ισχύσει. Εμείς ε, θα συμμετέχουμε και στις μελλοντικέ συζητήσεις με επικοδομητικές προτάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Καντέκ από το, Γαλλικό Ευρω... από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με συγχωρείτε. Ευχαριστώ. Ε, κυρία συνάδελφε από την Ομοσπονδιακή Γερμανική Βουλή, θα διαφωνήσω μαζί σας. Δεν θέλω να εφαρμοστεί το σύστημα των μεταβιβάσεων, μεταβιβάσιμων παραχωρήσεων, διότι θεωρώ ότι έτσι νομισματοποιείται το σύστημα και θα αποφασίζει η αγορά τελικά. Βλέπουμε όμως και σε άλλους τομείς που μας έχει οδηγήσει η αγορά όταν οδηγεί εκείνη. Ε, αναπόφευκτα θα συγκεντρωθούν κεντρικά όλα τα δικαιώματα και όχι μόνο αυτό, αλλά θα υπάρξει και κατάχρηση δεσπόζουσα θέση σε πολλέ περιπτώσει και σα πενθυμίζω ότι αυτό αντιβαίνει στου κανόνε τη νέα αγορά και τη συνθήκη. Ε, αυτή η ομαδοποίηση των δικαιωμάτων θα οδηγήσει σε δραστική μείωση του αριθμού ε, των σκαφών Οπότε θα αλλάξει όλη η ε, χορτακτική διευθέτηση, αν θέλετε, των ε, επιμέρους περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας λέει η κυρία Δαμανάκη ότι προτείνονται δικλείδες ασφαλείας. Ναι, προτείνονται, αλλά αντιβαίνουν στην ε, συνθήκη και συγκεκριμένα στις διατάξεις περί ενιαίας αγοράς. Λοιπόν, Ίσως δεν σας κατάλαβα κιόλας. είχα καταλάβει ότι είστε υπέρ του συστήματος των μεταβάσιμων παραχωρήσεων. Γι' αυτό τα λέω αυτά. Ε, συγκεκριμένα θα πρέπει να ανανεωθεί ο στόλος. Σας υπενθυμίζω ότι κατά μέσο όρο είναι 27 χρονών περίπου τα σκάφη και υπάρχουν καταστροφές κάθε χρόνο γιατί είναι απαρχαιωμένα τα σκάφη. Και στη Γαλλία ε, είχαμε νεκρούς πρόσφατα ε, λόγω, του, λόγω αυτού θα πρέπει με ευφιέστερο τρόπο να αλλιεύουμε με ασφαλέστερα ε, σκάφη και πιο ε, επιλεκτικούς εξοπλισμούς. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας ούτω ή άλλω, ε, αν δεν έχουμε ψάρια, δεν θα έχουμε και ψαράδε. Οπότε, πρωταρχικό στόχο ε, είναι να προστατεύσουμε τα αποθέματα. Φυσικά, για τι παράκτιε περιοχέ είναι σημαντικό να ε, προστα... λάβουμε υπόψη την οικονομική και την κοινωνική πτυχή. Σχετικά με την απαγόρευση των απορρίψεων, νομίζω προσυπογράφουμε όλοι αυτό το στόχο. για τι απορρίψει, φυσικά δεν μπορούμε να πετούμε τα ηχθίδια επειδή δεν έχουν εμπορική αξία, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορέσουμε ούτε να εκφορτώσουμε ούτε να χρησιμοποιήσουμε τις ε, απορρίψει με το νέο σύστημα. Σα ευχαριστούμε κύριε Καντέκα. Ο κύριο Χάρινγκτον ε, τώρα από την Ιρλανδία. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ πρόεδρε. Λίγε ερωτήσει προ το πάνελ. Η Ιρλανδία είναι κατά των παραχωρήσεων, των μεταβιβάσιμων γιατί έχουμε αντίφαση μεταξύ των ε, ιδιοκτήτων και των ε, κοινών ε, παραχωρήσεων. Ο στόλος μας συμμετέχει στα εθνικά ιδρύματα μαζί με άλλους στόλους και δεν θα υπήρχαν διασφαλίσεις έτσι. Επίσης, η... πολλές φορές η ικανότητα μπορεί να φύγει από τη χώρα. Δεν υπάρχουν ε, εγγύηση σε αυτό το τομέα και αυτό μας ανησυχεί. Επίσης ε, θα ε, υπήρχαν έτσι στόλοι, θα δημιουργούνταν στόλοι που δεν θα λειτουργούσαν με βάση το κριτήριο της βιωσιμότητας. Όταν μειώνονται οι στόλοι και ο αριθμός των σκαφών σε ένα τύπο αλίας, πολλοί αυξάνουν το μέγεθος των σκαφών, μήκος κινητήρα και έτσι αυξάνεται η ικανότητα. Παρά τα μέτρα μείωσης, θα πρέπει τα κράτη-μέλη να αποφασίζουν τις παραχωρήσεις και την ευελιξία που θα προβλέπεται εκεί. Εκεί εδώ επιμένουμε. Τώρα, για τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, ναι να επιτευχθεί, αλλά όχι μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπει η Κομισιόν. Σε, κάποιες, σε κάποιους τύπους αλληλείας μπορεί να γίνει αυτό, αλλά μόνο με σύμφωνη γνώμη των αλλιέων και με τοπικά σχέδια διαχείρισης. Και αυτό θα είναι δύσκολο να επιτευχθεί μέχρι ε, το 2015. Για τις απορρίψεις, αυτό ε, μας βρίσκει σύμφωνος, αλλά δύσκολα θα επιτευχθεί. Μπορεί να γίνει σε κάποιους τύπους αλίας βραχυπρόθεσμα. Ε, στη μεικτή αλία δεν μπορεί να γίνει. Και καλό την Κομισιόν να ζητήσει από τα κράτη-μέλη να ε, δώσουν στοιχεία ε, και για βενθικά είδη και για μεικτή αλία, ώστε να ξέρουμε καλύτερα το αντικείμενο πριν λάβουμε αποφάσεις. Ο κύριος Κοκκίνης από τη Λιθουανία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντική η συζήτηση αυτή γιατί υπάρχουν ε, πολλές και διαφορετικές απόψεις. Βεβαίως η μεταρρύθμιση είναι σωστή, αλλά τα χρονοδιαγράμματα μας ε, φοβίζουν. Δηλαδή θα έχουμε προβλήματα, δεν θα μπορέσουμε να τα τηρήσουμε διότι πίσω από κάθε κανονισμό βρίσκονται άνθρωποι όπως ε, ακούσαμε και κλάδοι ολόκληροι. Σημαντικό να επιδιώκουμε στόχους αλλά με ευελιξία στα χρονοδιαγράμματα. Αν είναι αυστηρά τα χρονοδιαγράμματα θα κερδίσουν οι χώρες που ε, θα παρουσιάσουν καθυστερήσεις ε, και που θα καθυστερήσουν να μεταβιβάσουν αρμοδιότητες. Αν ε, μια χώρα δεν μπορεί να αξιοποιήσει τις ποσοστώσεις, θα πρέπει να μπορεί να τις ε, μεταβιβάζει. Αλλά όταν πρόκειται για μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ χωρών, αυτό δεν είναι καλό, διότι οι ισχυρότερες χώρες ε, με ισχυρότερο τομέα αλληλείας θα υπερισχύσουν πάνω στις χώρες ε, όπου ο τομέας αυτός είναι πιο αδύναμος. Βεβαίως όλοι θα πρέπει να αποκομίζουν κέρδη ε, στον τομέα αυτών. Δεν πρέπει λοιπόν να σπεύσουμε, μη βιαστούμε. Προβλέπεται μεταφορά ε, κονδυλίων από το Ειδικό Ταμείο μετά το 2014 όμως. Γι' αυτό δεν πρέπει να βιαστούμε. Ευχαριστώ. από τις κατοχώρες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κοιτάξτε, αν αδειάσουν οι θάλασσε, ε, κανεί ε, δεν θα βγει κερδισμένο. Συμφωνούμε με την Επίτροπο, λοιπόν. Πρέπει λοιπόν να δούμε πρώτα τι παράγει η θάλασσα. Αλλά πώς ε, μπορούμε να το πράξουμε αυτό, να βελτιώσουμε την παραγωγή τη θάλασσα με ποιε μεθόδους. Σε ό,τι φορά τώρα τη βιώσιμη αλία, η Κομισιόν ε, μας είπε ότι πρέπει να αναπτυχθεί και απασχόληση, αλλά σε ποια βάση μπορούμε να κάνουμε ε, μια τέτοια δήλωση. Ευχαριστώ. Καπακ Κασένα από τον Στακ Ευχαριστώ κυρία Ρόντους για την έκθεση και ευχαριστώ και την ε, κυρία Δαμανάκη. Χρειάζονται τολμηρές μεταρρυθμίσεις, αυτό είναι σωστό. Ξέρουμε ότι οι ποσοστώσεις κατανέμονται σήμερα με βάση το, την αρχή της ε, σχετικής σταθερότητας και αναρωτιέμαι πώς ε, με, τη, το σύστημα με τις μεταβιβάσεις ε, με τις μεταβιβάσιμες παραχωρήσεις θα διατηρηθεί το σύστημα της σχετικής σταθερότητας ιδιαίτερα ε, όταν γίνεται μεταξύ κρατών μια τέτοια παραχώρηση. Αποδυναμώνεται η δυνατότητα των κρατών μελών να ασκούν περιφερειακή πολιτική. Εγώ είμαι από το Σλέσβι Χόλσταϊν ε, που ε, για αυτό το κρατήδιο και η Βαλτική και η Βορεια Θάλασσα είναι σημαντική. Μέχρι τώρα δεν καταφέραμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσουμε την πλεονάζουσα ικανότητα. Ίσως επειδή εκεί όπου έχουμε ε, πλεονάζουσα ικανότητα υπάρχουν εναλλακτικές, δεν υπάρχουν εναλλακτικές δυνατότητες δημιουργίας εισοδήματος. Αυτό το πρόβλημα ξεπερνάει την ε, ε, εθνική αλληλεία. Ε, είναι θέμα κοινή αλληλευτική πολιτικής. Θα πρέπει λοιπόν παντού να προβλέψουμε σωστά μέτρα για τη μείωση της πλεονάζουσας ικανότητας. Βέβαια, δεν μιλάμε μόνο για βιώσιμη αλληλεία, ε, λαμβάνοντας υπόψη τα ψάρια, θέλουμε βιώσιμη αλληλεία και για τους ίδιους τους αλληλείς. δύο λόγια για την απαγόρευση των απορρίψεων θέλω αυτό να γίνει με βάση τον τύπο της αλίας και όχι με βάση τα είδη των ηχθείων. Θα πρέπει ψάρια που έχουν δυνατότητα επιβίωσης όταν ε, απορριφθούν να λαμβάνονται υπόψη. Ε, δεν ε, θα πρέπει να εκφορτώνονται αυτά σε κάθε περίπτωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σκεντεμόν από το Καλλικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η μελλοντική αλλιευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης εστιάζεται γύρω από αυτή τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Ε, κοιτάξτε, δεν νομίζουμε ότι προλαβαίνουμε να το κάνουμε αυτό μέχρι το 2015. Μέχρι το 2020 χρειαζόμαστε χρόνο, διότι πρέπει να διατηρηθούν τα αποθέματα. Ε, υπάρχει, υπήρχε στο παρελθόν η Τεχνική, Οικονομική και Επιστημονική Επιτροπή. Θέλουμε να επανασυσταθεί διότι ε, παρατηρούσε καθημερινά την κατάσταση επιτόπου και έτσι μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε οποιαδήποτε δράση. Ζητούμε επίσης κοινωνική προστασία ε, του ΑΛΙΕ. Χρειαζόμαστε επίσης ένα έλεγχο ω προς την εφαρμογή της νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό γιατί ότι το μισθολογικό και το κόστος και το κόστος παραγωγής διαφέρει από χώρα σε χώρα. Ε, δεν είναι ρεαλιστική η πρόταση γιατί υπάρχουν ε, ε, μη προσαρμοσμένα τεχνικά μέτρα. Έχουμε διάφορα προβλήματα βάσει του ισχύοντος συστήματος, αλλά δεν ξέρω αν μπορούμε να δεχτούμε τις νέες προτάσεις. Είμαστε κάθετα αντίθετοι σε αυτό το σύστημα των μεταβιβάσιμων παραχωρήσεων. Θα σημάνει το θάνατο της ερασιτεχνικής βιομηχανικής ε, αλληλεία, ε, ε, αυτά τα δικαιώματα, αυτέ οι παραχωρήσει θα πρέπει να διέπονται από διαφάνεια και να υπάρξει ισότιμη κατανομή. Άρα θα πρέπει να τα διαχειρίζονται οι εμπορικοί εργασία των αλλήλ, ασφάλεια των πλοίων και ούτω καθεσή. Εμεί είμαστε υπέρε τη περιφερειακή διακυβέρνηση του κλάδου. επιση το ίδιο ισχύει για τι συνθηκε ασφαλεια κατά την εργασία των αλλήλων, ασφάλεια των πλοίων και ούτω καθεξή. εμει είμαστε υπέρ τη περιφερειακη διακυβερνηση του κλάδου. τελο η μεταρρύθμιση τη ΚΟΑ στο στον κλάδο της αλίας θα πρέπει να επιτρέψει πιο ευέλικτε σχέσεις ανάμεσα σε επαγγελματικέ οργανώσεις. Χρειαζόμαστε δηλαδή ένα πιο ευέλικτο όργανο για να ρυθμίσουμε την αγορά. Επίση. θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις περιβαλλοντικές ανησυχίες ε, ε, και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά τι εισαγωγέ. Ευχαριστούμε τώρα από τη Λετωνία ο κύριο Μπλούφελντ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ρόντουστ. Εμεί μπορούμε να υποστηρίξουμε την προσέγγιση μέγιστη βιώσιμη απόδοση, ε, αυτή τη στεδιακή προσέγγιση, αλλά είναι σημαντικό να πετύχουμε σε σταδιακούς ρυθμούς αυτά τα επίπεδα. Πιστεύουμε ότι μια τέτοια προσέγγιση θα πρέπει να εφαρμοστεί στη Σαρδελόρεγκα, στο ΣΠΡΑΤ, και στα πελαγικά είδη στη Βαλτική και δεν πιστεύουμε ότι είναι αποδεκτή η προθεσμία του 2015 καθώς σήμερα οι διορθώσεις σε ό,τι αφορά τα αποθέματα δεν εφαρμόζονται και θα έπρεπε να μιλήσουμε ε, εδώ για το γάδο και νομίζουμε ότι θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε ε, για την απαγόρευση των απορρίψεων αν συμπεριληφθεί στις ποσοστώσεις παράλληλα με την απαγόρευση θα πρέπει να εξετάσουμε και τα πρότυπα που ισχύουν στη διατροφικό τομέα, στον τομέα των τροφίμων, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι οι σημερινοί πόροι δεν θα χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους πέραν της διατροφής. Ε, σε ό,τι αφορά τώρα τις απαγορεύσεις των απορρίψεων, θεωρούμε ότι δεν ε, πρέπει ε, να δημιουργούμε μεγαλύτερο άχθο για τους αλείς και για τους φορείς ελέγχους, ελέγχου Παραδείγματο χάρη θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ε, το θέμα ε, των καμερών παρακολούθησης ε, στα σκάφη. Δεν θεωρούμε ότι είναι εύλογο να υπάρχει κάτι τέτοιο. Θα συνεργαστούμε με την Κομισιόν για να βρούμε λύσεις επωφελείς για όλους και αυτό σημαίνει ότι είμαστε έτοιμοι να ε, προχωρήσουμε προς τη μεταρρύθμιση, αλλά θα πρέπει να διορθώσουμε ορισμένα στοιχεία. Κυρία Μπέκτα από το Bundestag. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και εσάς κυρία Ρόντους για την έκθεση. Συμφωνούμε και είναι και έξυπνη ιδέα η απαγόρευση απορρίψεων να γίνει σταδιακά και ανάλογα με το ε, ποσοστό Επιβίωση των μικρών των ψαριών στο κάθε είδος. Δεν έχει νόημα όμως από άποψη πόρων τα μικρά ψάρια να μην χρησιμοποιούνται ως ηχθιάλευρα αλλά ε, με καλύτερο τρόπο και να είναι αυτό ένα κίνητρο ώστε να ε, ένα σημαντικό ε, ε, ποσοστό των πόρων να ε, επαναρρίπτονται. Επίσης, για την μείωση της πλεονάζουσας ικανότητας, πότε θα υπάρχει ένα, μια διαδικασία που να μας δείχνει σε ποιο βαθμό οι εθνικές ικανότητες θα ευθυγραμμίζονται με τις αλλιευτικές δυνατότητες. Δεν θα πρέπει πάνω σε αυτή τη βάση να υπάρξουν μετά μέτρα για στοχευμένη μείωση της πλεονάζουσας ικανότητας και όχι γενικά μέτρα που θα ισχύουν ε, γενικά για όλους τους στόλους. Μια άλλη πρόταση. Ε, μήπως ε, μπορούμε να καταργήσουμε την αρχή της αλλιευτικής προσπάθειας. Δηλαδή, αν, ε, υπάρχουν, αν υπάρχει ε, βάλουσα, ε, πλεονάζουσα ε, ικανότητα να συνυπολογίζεται στα συνολικά επιτρεπόμενα αλλιεύματα. Επίσης, οι προθεσμίες υπάρχουν προβλήματα σε σχέση με τη στρέβλωση του ανταγωνισμού και κάποια μέτρα, εάν παραμείνουν ε, προαιρετικά, δεν θα εφαρμοστούν από κάποια κράτη-μέλη. Ίσως λοιπόν θα έπρεπε να είναι ε, υποχρεωτικά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος από τη Γερουσία της Ισπανίας. Ευχαριστώ. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή για αυτή την ε, συνεδρίαση, γιατί για μας, ε, για την Ισπανία και την Γαλλική είναι καθοριστική μεταρρυθμίση αυτή. Καταρχήν θα ήθελα να πω και γι' αυτό θα επαναλάβω κάποια ζητήματα με τα οποία συμφωνούμε όλε οι πολιτικέ ομάδε τη Ισπανίας ότι η βιωσιμότητα τη αλίας είναι ένα κοινό στόχο. Ε, αλλά αυτό που ε, ε, απασχολεί κυρίω είναι το ότι πρέπει να υπάρχει και οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα. Πρέπει να προστατεύσουμε και του αλίες προστατεύοντα την αλία και να λαμβάνουμε υπόψη ότι η απασχόληση είναι η κύρια ανησυχία των κοινωνιών μας αυτή τη χρονική στιγμή και έτσι θα πρέπει να προβλέπεται και η διαφοροποίηση της οικονομική δραστηριότητα ε, στον κλάδο. Δεύτερον, ε, σε σχέση με το πρέπει ε, η μέγιστη βιώσιμη απόδοση που προβλέπεται για όλα τα είδη, αν και έχει καλές προθέσεις, θεωρούμε ότι δεν είναι ρεαλιστικό στόχο. Έτσι λοιπόν θα ήταν πιο χρήσιμο να έχουμε την άμεση βιολογική ασφάλεια για τα κινδύνα που είναι σε κίνδυνο και να διευρύνουμε σε συγκεκριμένα αποθέματα το στόχο της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης με μεγαλύτερη προθεσμία επίση η αρχή τη πρόληψη δεν μπορεί τυφλά να εφαρμοστεί ούτε να οδηγήσει σε δραστικέ περικοπέ. Ό,τι αφορά τι απορρίψει, να πούμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε στην εξάλληψη, αλλά πρέπει να γίνει σταδιακά, με σχεδιασμένο τρόπο και να έχουμε ε, ε, ε, επαρκή χρόνο για να γίνει αποδεκτό από τον κλάδο. Το να γίνει άμεσα θα μα δημιουργήσει δυσεπίλητα προβλήματα. Και συμφωνώντας ε, με τις μεταβάσιμε ελευθερικές παραχωρήσει μπορεί να είναι ένα κατάλληλο προσανατολισμό. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να εισαχθεί ευελιξία ε, που να επιτρέπει την εφορία και την αντιγωνιστικότητα του τομέα. Την πρώτη απέτηση ε, είναι να γίνονται αλλιεύσει σε αλλιεύματα για τα οποία υπάρχουν ποσοστώσεις. επίση θέλουμε να εξαιρείται και η αλλία μικρή κλίμακα. Δεύτερον, πρέπει να διαφοροποιηθεί η βιομηχανική αλία από την αλία μικρή κλίμακα και πρέπει να διαφοροποιηθεί η βιομηχανική υδατοκαλλιέργεια από την παραδοσιακή υδατοκαλλιέργεια, η οποία σέβεται το περιβάλλον και επίση πρέπει να συμπεριληφθεί και η εκτροφή ε, των μαλακίων ε, και εκεί να λαμβάνουμε υπόψη και το ρόλο των γυναικών ε, που έχουν τεθεί σε περιθωριοποίηση στο παρελθόν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σορτέλ από την Bundestag. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, οι δύο συνάδελφοί μου από τον Bundestag και τον Bundesrat, άνω κάτω βουλή, ε, μίλησαν για όλα τα θέματα και έλαβαν θέση. Ε, δεν θα τα επαναλάβω. Μία παρατήρηση μόνο θα προσθέσω. Μέχρι τώρα... Ε, λαμβάναμε τα κείμενα της Κομισιόν και ξέρω από πολλές συζητήσεις και από συναδέλφους ε, που βρίσκονται ε, εδώ σήμερα ότι και ε, πραγματικά τους τελευταίους μήνες απελπιστήκαμε με αυτά που μας πρότεινε η Κομισιόν. Πολλές φορές έχουμε την εντύπωση ότι δεν αντλούν διδάγματα από το παρελθόν. Βεβαίως ε, τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αναλάβει μεγάλο ρόλο ε, στο πρόσωπο της κυρίας Ρόντουστα και ε, στη δεκάλεπτη ομιλία της μίλησε πάρα πολύ συγκεκριμένα, γνωρίζει το θέμα πολύ καλά και βέβαια στο επίκεντρο της εργασίας της είναι η αλληλής. Καλό τα Εθνικά Κοινοβούλια να συμφωνήσουν με την κυρία Ρόντουστα και να προχωρήσουν προς αυτή την κατεύθυνση που προτείνει, γιατί έτσι θα προχωρήσουμε σωστά. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες να κάνουμε ε, εφικτές συμβιβαστικέ ε, τροπολογίες και να βρούμε εφικτές συμβιβαστικέ λύσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τέλος. Ο κύριος Κάρτινε ε, από το Ηνωμένο Βασιλείο. If the Commission's proposals are to αν, για να πετύχουν οι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής χρειαζόμαστε μια οικοσυστημική προσέγγιση. Οι συνάδελφοι σήμερα δικαίω μίλησαν και για την οικονομική και κοινωνική διάσταση. Δεν μπορούν να εκλείψουν οι σε μικρή ε, κλίμακα, όπω είπαν και οι συνάδελφοι από την Ιρλανδία παραδείγματο χάρη. Και όχι μόνο μπορούν όμω δυστυχώ, αλλά θα εκλείψουν. Δεν έχουν κινητήρε εδώ και 150, πριν από 150 χρόνια τα σκάφη μα. Δεν είχαμε δορυφόρου, τίποτα δεν είχαμε παρό όλα αυτά οι ε, δικοί μας ε, ε ψάρευαν 13 φορές περισσότερα ψάρια σε σχέση ε, με σήμερα από, σε διάφορες περιοχές του του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν δημιουργηθεί μεγάλες κοινότητες αλλιών, αλλά ε, ε, εξαφανίζονται διότι αγνοούμε αυτή την ανάγκη για υιοθέτηση οικοσυστημικής προσέγγισης. Χρειάζεται όμως και μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου. Όπως μας υπενθύμισε η κυρία Ρότους, δεν έχουν διαβατήρια τα ψάρια. Καταλαβαίνετε, μετακινούνται και χρειαζόμαστε ε, οπωσδήποτε να αποφύγουμε τα εθνικά σύνορα και την ε, οριοθέτηση συγκεκριμένων περιοχών. Χρειαζόμαστε συνολική προσέγγιση. Κυρίω στο Βυσκαϊκό κόλπο μα μίλησε η κυρία Ρόντου ε, για το 2015 και το στόχο τη ε, ε, μέγιστη βιώσιμη απόδοση και είπε να βασιστούμε στα ψάρια. Αυτό είναι σωστό. Ε, γιατί μόνο αυτή η μέγιστη βιώσιμη απόδοση μπορεί να επιτευχθεί, αυτή που βασίζεται στην εθνισμότητα των ψαριών. Ναι, χρειαζόμαστε όντω καλύτερη διαχείριση, αλλά για να έχουμε καλύτερη διαχείριση θα πρέπει να έχουμε και πιο αξιόπιστα επιστημονικά δεδομένα. Μόνο έτσι θα επιτύχουμε τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Καταλαβαίνετε ότι αν δεν μπορούν να εκφορτώσουν οι αλείς δεν θα έχουμε ούτε τα επιστημονικά δεδομένα. Χρειαζόμαστε σωστέ επιστημονικέ συμβουλέ. Πώ θα γίνει αυτό χωρί εκφορτώσει, πώ θα υπολογίσουμε τη βιομάζα όλων των ψαριών όχι μόνο αυτών που έχουν εμπορική αξία. Μόνο έτσι μπορούμε να κάνουμε μια σφαιρική αξιολόγηση του συστήματο και να υιοθετήσουμε αυτή την οικοσυστημική προσέγγιση. Χρειαζόμαστε μια ε, συνεταιριστική ε, τοπική διαχείριση και όχι αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σα ευχαριστούμε. Μάλιστα, ολοκληρώσαμε λοιπόν το γύρω των ερωτήσεων. Να δώσουμε τώρα το λόγο στην κυρία Ρόντουστ για να προσπαθήσει να συνοψίσει. Γιατί πολλέ ε, από τι ερωτήσει ε, οδεύουν προ την ίδια κατεύθυνση. Παρακαλώ, προσπαθήστε να συνοψίσετε, κυρία Ρόντουστ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θερμό ευχαριστώ προς όλους τους συναδέλφους για τις παρεμβάσεις τους που με ωφελούν πολύ. Κατέγραψα πολλά πράγματα. Πολύ σύντομα να σχολιάσω κάποια πράγματα. Ο συνάδελφος από την Αυστρία. Ευχαριστώ ε, για την προσθήκη στην πρόταση 18. Θα το δω. Καλό θα ήταν όμως να μου το στείλετε και εγγράφος. Ε, ο Ισπανός συνάδελφος θεωρεί ότι δεν γίνεται μέγιστη βιώσιμη απόδοση να επιτευχθεί μέχρι το 2015. συμφωνώ. Γι' αυτό στην πρότασή μου μιλάω για το FMSY γιατί έμαθα τις τελευταίες εβδομάδες ότι για βιολογικούς λόγους εν μέρη δεν μπορεί η μέγιστη απόδοση να επιτευχθεί μέχρι το 2015 και θέλω να είναι ρεαλιστική η μεταρρύθμιση. Οπότε το είπα αρχικά. Τώρα, για τις μεταβιβάσιμες παραχωρήσεις. Δείτε τις προτάσεις μου 18 και 19 επ' αυτών, γιατί λέω ότι οι μεταβιβάσιμες ελευθερικές παραχωρήσεις θα εφαρμόζονται μόνο όταν αρνείται ένα κράτος μέλος ε, τη να, να, τη... μειώσει την σαφή πλεονάζουσα ικανότητα. Πως ε, ε όταν υπάρχει πλεονάζουσα ικανότητα θα πρέπει να μειώνεται. Αυτό δεν το κάναμε στο παρελθόν. Στην έκθεση θα υποβάλουμε κι άλλες προτάσεις και τονίζω πάλι ότι πιστεύω ότι τα TFCs, οι μεταβιβάσιμες ελευθερικές παραχωρήσεις, θα εφαρμόζονται όταν αρνείται ένα κράτος μέλος να μειώσει την ικανότητα. Τότε θα είναι δεσμευτικές. Ο πρώτος συνάδελφος από τη Γαλλία είπε ότι επιθυμεί καλύτερη συνεργασία μεταξύ επιστήμης και αλίας. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω μαζί του, αλλά αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινεί, στο παρελθόν πολύ συχνά υπήρχε μια, διαφορά μεταξύ απόψεων αλληλείας και επιστήμης. Οι αλληλείς ε, θεωρούσαν, οι επιστήμονες θεωρούσαν ότι οι αλληλείς δεν είναι αρκετά ενημερωμένοι και οι αλληλείς από την άλλη έλεγαν ότι είναι υπερόπτες οι επιστήμονες και δεν ξέρουν την καθημερινή πραγματικότητα. Και οι δύο έχουν τα δίκαια τους, αλλά εγώ νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να κάτσουν και οι δύο, τα δύο μέρη γύρω από ένα τραπέζι. Και εμείς ως Κοινοβούλιο πρέπει να φροντίσουμε να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί χρειαζόμαστε κατεπηγόντως στοιχεία. Απορρίψεις πρέπει να αποφεύγονται και πολλοί από εσά συμφώνησαν μαζί μου εδώ. Οι ιδέες από τη Γαλλία μου φαίνονται πολύ καλές και θα τις εξετάσω ε, λεπτομερέστερα. Εν πάση περιπτώσει οι απορρίψεις θα πρέπει να ε, αποτιμώνται με κάποιο τρόπο. Στο τέλος ο συνάδελφος από τη Μεγάλη Βρετανία είπε ότι... Ε, θα πρέπει να έχουμε καλύτερο σύστημα δεδομένων για να αποφεύγουμε τις υπερβολές της απορρίψης. Η συνάδελφος από την Ιταλία είπε ότι θα πρέπει να δείξουμε μεγαλύτερο σεβασμό στους αλληλείς. Βεβαίως και πρέπει. Αλλά πρέπει επίσης να πω ξεκάθαρα ότι... Ε, αν δεν φροντίσουμε για την βιωσιμότητα, μπορεί να σεβόμαστε τους αλληλείς, αλλά δεν θα έχουν αλλιεύματα. Ε, εγώ δείχνω το σεβασμό μου προς τους αλληλείς επιτρέποντας στα παιδιά τους να ε, συνεχίσουν ε, να δραστηριοποιούνται στον κλάδο αυτό. Το τελευταίο διάστημα ασχοληθήκαμε πάρα πολύ και με τους επαγγελματίες του κλάδου και με τους επιστήμονες για να καταλήξουμε σε ένα σωστό σύστημα. Τώρα, το σύστημα των μεταβιβάσιμων ποσοστώσεων η Ιταλίδα συνάδελφος δεν συμφωνεί γιατί ε, στη Μεσόγειο δεν ε, λειτουργούν οι ποσοστώσεις. Ναι, ε, πράγματι δεν έχουμε ακόμη ποσοστώσεις στη Μεσόγειο και ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα. Οι μεταβιβάσιμες παραχωρήσεις δεν μπορούν να διαπραγματεύονται. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Και είπα στην εισαγωγική μου ομιλία ότι χρειάζεται ένα χωριστό κεφάλαιο για τη Μεσόγειο και τον Εύξηνο Πόντο. Στη σοσιαλιστική μου ομάδα παρακάλεσα τους συναδέλφους από τη Μεσόγειο και από τον Εύξηνο Πόντο να συνεργαστούν για να επεξεργαστούν και να υποβάλουν προτάσεις. Για την αλληλεία μικρής κλίμακας, το είπε και η Επίτροπος Δαμανάκη και οι συνάδελφοι από την Ιταλία, ε, και τον ορισμό που πρέπει να ξεπερνάει τα 12 μέτρα. Είναι λάθος ο ορισμός ε, μπορεί κάποιος να έχει ισχυρότατο κινητήρα πάνω σε σκάφος 12 μέτρων και τόσο πολύ αποτελεσματικά αλλιευτικά εργαλεία που να είναι μεγάλης κλίμακας αλληλεία. Δεν με πείθει λοιπόν αυτό. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε τι κύκλο εργασιών έχει αυτό το σκάφος και πώς λειτουργεί και πώς είναι, ποια είναι η δομή της επιχείρησης. Ε, για την Φλάνδρα ε, το 2015 και τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Το είπα και εγώ ότι δεν προλαβαίνουμε, αλλά θα πρέπει να είναι δεσμευτική ε, για το 2015. Και υπάρχουν αρκετές πληροφορίες και δεδομένα από την επιστήμη ότι μπορούμε να στηριχτούμε σε, στη συνιστόσα που σας είπα. Τώρα, για τις μεταβιβάσιμες αλληλευτικές παραχωρήσεις, δείτε την πρότασή μου υπαριθμών 19 Πιστεύω ότι δεν διαφέρουν οι απόψεις μας. Ευχαριστώ για την κυρία Ρούφ για την υποστήριξή της. Ο ορισμός των μικρών, της μικρής κλίμακας αλλιέων πρέπει να τον δούμε. Εγώ έχω κάνει μια πρόταση. Τώρα, αν θα περάσει δεν το ξέρω ακόμα. Αλλά είμαι ευγνώμων για κάθε ιδέα που θα μου δώσετε. Πάντως το να λέμε ότι μικρός αλλιέας είναι με σκάφος 12 μέτρων, αυτό σήμερα δεν αρκεί. Ε, συνάδελφοι από, συνάδελφος από την ε, ε, Ιρλανδία, είστε κατά των μεταβιβάσιμων αλληλευτικών παραχωρήσεων, ενδεχομένως, αλλά σκεφτείτε τι θα κάνουμε με τις χώρες που έχουν πλεονάζουσα ικανότητα. Η κυρία Φράγκα είναι εδώ μαζί μας, που είναι σκιώδης δική μου στην έκθεσή μου και στη συνάντηση των σκιωδών η κυρία Φράγκα είπε κάτι το οποίο χαράχτηκε στο μυαλό μου. Πρέπει να εξηγήσω ότι η κυρία Φράγκα είναι θεσμός εδώ στο Κοινοβούλιο. Ασχολείται με την αλληλεία από τότε που ήρθε στο Κοινοβούλιο και είναι πολλά χρόνια ευρωβουλευτής. Ε, δεν υπάρχει χώρα που, δέχεται, που παραδέχεται ότι έχει πλεονάζουσα ικανότητα, λέει η κυρία Φράγκα. Νομίζω ότι ε, είναι λόγος αυτός για να σκύψουμε πάνω από το θέμα και να δούμε πού όντως υπάρχουν πλεονάζουσες ικανότητες, γιατί ξέρουμε, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινεί, ότι εξακολουθούμε να έχουμε πλεονάζουσα ικανότητα. Αλλιώς δεν θα καθόμαστε εδώ να συζητάμε. Θα μπορούσαμε να διαμορφώσουμε αλλιώς τον ελεύθερο χρόνο μας. Προς συναδέλφους από την Ιρλανδία πάλι για τις μεταβάσιμες παραχωρήσεις, ε, μίλησα γι' αυτό, φοβάστε τη διαπραγματευσιμότητα των ποσοστώσεων. Εγώ στο έγγραφο εργασίας μου και μάλιστα δεν το συζητούμε επί διαφορετικής βάσης στην Επιτροπή. Καθιστώ απόλυτα σαφές ότι η διαπραγματευσιμότητα θα γίνεται μόνο ε, στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να το δουν αυτό πολύ προσεκτικά και τη διαπραγματευσιμότητα να την οργανώσουν σωστά και με βάση το μέγεθος ενός τύπου αλίας. Γιατί όταν η διαπραγμάτευση ωφελεί μόνο τους μεγάλους, ε, τότε δεν θα υπάρχει πια μικρής κλίμακας αλία. Δείτε το λοιπόν και βοηθήστε τις κυβερνήσεις να, λάβουν σωστές να λάβει σωστές αποφάσεις. Εγώ δεν θα ήθελα η διαπραγματευσιμότητα να ξεπερνά τα εθνικά σύνορα και να προβλέπεται και εκεί. Σπέβδω να προσθέσω σε αυτούς που το περιμένουν ότι ήδη από τώρα υπάρχουν αρκετές δυνατότητες για κάτι τέτοιο, αλλά εγώ δεν θα το συμπεριλάβω στις προτάσεις μου, σίγουρα όχι. Ο συνάδελφος από τη Λιθουανία είπε ότι δεν προλαβαίνουμε με τα χρονοδιαγράμματα. Ε, απαντώ ότι εμείς μιλούμε για το 2015 ε, γιατί οι επιστήμονες όλα τα κράτη-μέλη επειδή κάναμε ακροάση με τους επιστήμονες, ότι το FMSY μπορεί να είναι εφικτό μέχρι το 2015 και ισότι ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες και τη μεταβιβασιμότητα, νομίζω ότι υπάρχει αρκετά ήδη. Η συνάδελφος από την ε, Ολλανδία είπε ε, πώς ε, αποδεικνύονται οι εξελίξεις και τα δεδομένα. Αυτό γίνεται σε συνεργασία με τους αλληλείς και τους επιστήμονες. Και από κοινού θα πρέπει να δούμε ε, τι αποθέματα έχουμε και τι είδη. Ε, για τις μεταβιβάσιμες ποσοστώσεις, ναι, αλλά μόνο ε, σε επίπεδο κράτους μέλους, όχι κάτι άλλο. Ναι, έχετε δίκιο, στο μέλλον θα έχουμε προβλήματα αν εφαρμόσουμε το φιλόδοξο σχέδιο της μεταρρύθμισης. Εγώ είμαι ευγνώμων διότι ολόκληρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησε ε, τα τρία μεγάλα ταμεία το Μεγάλο Ταμείο Γεωργίας, το Μεγάλο Ταμείο Συνοχής ε, και το Μεγάλο Ταμείο Αλίας ε, να τα βάλουν κάτω από μία αιγίδα. Θα ε, αποφασίζομαι σε σχέση, το κάθε ταμείο ε, θα αποφασίζει για τα κονδύλια του, αλλά η χρησιμοποίηση θα αποφασίζεται ε, από κοινού. Και θα γίνονται διαβουλεύσεις και με άλλες επιτροπές, Περιφερειακή Επιτροπή για παράδειγμα, ούτως ώστε να υπάρχουν εναλλακτικέ προσφορές προς τους αλληλείς. Τώρα, για το 2020 ε, και αυτά που είπαμε το MSY, δεν θα το επαναλάβω, σταδιακή εφαρμογή του MSY για το, θα αρχίσουμε με το FMSY και αργότερα θα μιλήσουμε για το υπόλοιπο όταν έρθουν και άλλα δεδομένα, ε, ούτως ώστε να είναι σωστή και η πρόταση. Έλεγχος των αλλιέων. Αυστηρό, είναι υπερβολικά αυστηρός αναφέρθηκε. Εκεί πρέπει να πω πρέπει να προσέξουμε ε, να μην το παρακάνουμε. Τα προηγούμενα χρόνια μάθαμε ότι οι έλεγχοι δεν διεξάγονταν σωστά σε κάποια κράτη-μέλη. Και αν συνεχιστεί αυτό, αν δεν, γίνεται σωστά η, δεν γίνονται σωστά οι έλεγχοι, τότε μπορούμε να αποφασίζουμε ό,τι θέλουμε στα κοινοβούλια μας, αλλά δεν θα έχουμε αποτέλεσμα. Ε, ε μπορώ να φανταστώ, ε, και εγώ του κόσμου αυτού είμαι, μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί κανείς να παρακάμπτει την νομοθεσία. Ε, πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε με σωστά μέτρα τους έντιμους αλείς που υπάρχουν πολλοί από αυτούς. Ε, τώρα για τα μικρά ε, ψάρια και την αξιολόγησή τους ε, δεν, η συζήτηση συνεχίζεται δεν θέλω να πω κάτι οριστικό τα νεαρά Όποιος αλλιεύει νεαρά ψάρια πρέπει να τιμωρείται με κάποιο τρόπο. Αυτό θα το δούμε καλύτερα. Πάντως έχω εμπιστοσύνη στους αλληλείς που έχουν μάθει ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η δραστηριότητα και στις επόμενες γενιές. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Για τα τέλη διαχείρισης της αλληλείας, ε, αυτό δεν έχει ακόμα συζητηθεί, ε, οπότε δεν θα το σχολιάσω καθόλου. Για τη Γαλλικία, ε, έχω πρόθεση να επισκεφθώ σύντομα τη Γαλλικία, θα συναντηθούμε και εκεί και θα συσκεφθούμε για ε, συστήματα ε, κοινωνικά δίκαια. Έχω υπόψη μου και τη λειτουργία των υπόλοιπων ταμείων και είπε και η κυρία Δαμανάκη ότι το καινούριο ταμείο, το ΕΤΘΑ, θα έχει κονδύλια στη διάθεσή του που πρέπει σωστά να διαχειριστούμε. Βεβαίως δεν πρέπει να ερμηνεύομαι περιοριστικά την αρχή της ε, προφύλαξης, όλοι κάνουμε σκέψεις σχετικά με τη σωστή ε, χρησιμοποίησή του. Βεβαίως, διαφοροποίηση χρειάζεται μεταξύ παράκτιας αλίας και βιομηχανικής αλίας. Ε, αυτό επίσης όπως ε, είδατε μας απασχολεί πολύ. Ε, επίσης ε, ευχαριστώ τον πρόεδρο της Γερμανικής Ένωσης Αλλιέων και όταν είναι τόσο φιλικά διακείμενοι οι αλλιείς τότε θεωρώ και εγώ ότι δεν έχω κάνει πάρα πολλά λάθη. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας και που απαντήσατε στις ερωτήσεις. Λοιπόν, έχουμε καθυστερήσει όπως πάντα, επομένως θα περάσουμε στο επόμενο πάνελ που έχει να κάνει με την κοινή οργάνωση αγορά και τι οργανώσει παραγωγών. Και θα δώσουμε για 10 λεπτά το λόγο στον κύριο Στίβενσον για την παρουσίαση. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Εξότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, καταρχήν, να αναφερθώ στο θέμα των οργανώσεων παραγωγών. Έχουμε 214 οργανώσεις παραγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν σημαντικό ρόλο διαδραματίσουν ε, όχι μόνο ως αντιστάθμισμα ε, στους λιανιμπόρους αλλά και στην καθημερινή διαχείριση των ελευτικών δραστηριοτήτων ε, υπέρ των μελών τους. Ορισμένε από αυτές το κάνουν πιο αποτελεσματικά από άλλους και ο κύριος στόχος της εκθεσής μου θα είναι να πετύχουμε ένα streamlining των οργανώσεων παραγωγών για να μπορούν να γίνουν πιο αποτελεσματικέ και να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ε, στην επιτεύξη της βιώσιμη Τα κριτήρια πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια για τον ελάχιστο αριθμό των μελών που θα πρέπει να ενθαρρύνεται να έχει μια οργάνωση παραγωγών, νομίζω θα πρέπει να συγχωνευτούν οι μικρότερε οργανώσει και οι διεθνικέ οργανώσει θα πρέπει ε, να ενθαρρύνονται στι ε, θαλάσσιε λεκάνε, έτσι ώστε να δεσμεύονται από κοινού και δεσμευτικού κανόνε. Ε, το θέμα τη διεθνοποίηση των οργανώσεων παραγωγών θα βοηθήσει τι εταιρείε να γίνουν πιο ανταγωνιστικέ σε διεθνέ επίπεδο για να πετύχουν του στόχου τη στρατηγική του 2020 και να δημιουργήσουν αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά στην ε, έκθεση μου υπάρχει επικάλυψη με την ε, έκθεση της κυρίας Ρόντεστ ε, για το βασικό κανονισμό, όμως ε, η απόλυτη επιτεκτική ανάγκη για την περιφερειοποίηση είναι πάρα πολύ σημαντική και τις οργανώσεις ε, παραγωγών ε, και για τους ελέγχους και για να γίνει αυτό ε, με κατάλληλο τρόπο θα πρέπει η Κομισιόν να παρουσιάσει μια δυνατότητα, μια σειρά μέτρων από τα οποία τα κράτη-μέλη θα μπορούν να επιλέγουν τα πιο κατάλληλα για τη δική του ελεία. Το να έχουμε μια βιώσιμη ελεία είναι πολύ πιο σημαντικό από το να διατηρήσουμε την ακαιρεότητα των συνθήκων. Και επίση οι οργανώσει παραγωγών θα έχουν σημαντικό να διαπραγματεύσουν στην ε, διαχείριση των ε, μεταβιβάσιμων παραχωρήσεων, που πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι κούσιο χαρακτήρα παρά υποχρεωτικέ και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν την ευελιξία να κατανέμουν δικαιώματα σε μία περίοδο 7-8 ετών και όχι 15 ετών όπως προτείνει η Κομισιόν. Τα κράτη-μέλη επίσης πρέπει να έχουν την τελική απόφαση για το αν μπορούν να είναι εμπορεύσιμα αυτά τα δικαιώματα. Θα πρέπει να φροντίσουμε να αποφύγουμε τη συγκέντρωση των TFC σε αυτών των παραχωρήσεων σε λίγες μεγάλες αλευτικές εταιρείες. Αυτό θα είναι παραγωγικό και θα έχουμε σοβαρές επιπτώσεις όπως όπως ακούσαμε, για τις θέσεις εργασίας στον τομέα και επίση. Οι οργανώσεις παραγωγών θα έχουν σημαντικό ρόλο και τα σχέδια διαπραγμάτευσης, στον καθαρισμό σχεδίων διαπραγμάτευσης και στην απαγόρευση αλίας Επίση, και θα μπορούν να δίνονται και ε, ψάρια σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, ψάρια που θα πήγαιναν για απόρριψη επανάληψη. Αν γίνει κάτι τέτοιο όμω, αυτό θα είναι καταστροφικό και οι τιμέ θα πέσουν ακόμη περισσότερο. Αυτά τα ψάρια θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για δόλωμα ή για ηχθιάλευρα όπου αυτό είναι δυνατό και να δίνεται επαρκή αποζημίωση στου αλείς για την εκφόρτωση αυτών των περιττών ψαριών και επίση θα πρέπει να υπάρχει και ε, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλεία ε, και Θάλασσα. Ε, και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη μοντέρνα τεχνολογία, τη σύγχρονη τεχνολογία υπέρ του τομέα έχουμε ηλεκτρονικέ αγορέ που λειτουργούν επιτυχώ σε διάφορα μέρη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. υπάρχει επίση δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί τεχνολογία για να βελτιώσουμε την ευβία των αγορών αναπτύσσοντα τι ηλεκτρονικέ αγορέ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και σχετίζοντά τι με ηλεκτρονικά ημερολόγια και συστήματα VMS. Έτσι λοιπόν θα αξιομολυθούν οι αγορέ για ορισμένα είδη και θα αποφευχθούν συμφορήσει ή λήψει και θα βελτιωθούν οι τιμές για όλου του ενδιαφερομένους. Επίση, θα πρέπει να έχουμε αρρωγή από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσα και σε αυτό το τομέα. Σε ό,τι αφορά τώρα την παρέμβαση τη αγορά, εδώ έχουμε ε, ένα σημαντικό επίμαχο σημείο στις ε, εκτεταμένε συζητήσει που είχα για την ε, πρόταση τη Κομισιόν, οποιαδήποτε σύστημα παρέμβαση με την ελεύθερη αγορά, όπω ο προτινόμενο σύστημα ε, μηχανισμού αποθήκευση ή ε, μηχανισμοί ε, ε, θα πρέπει να τα δούμε πάρα πολύ προσεκτικά. 45 εκατομμύρια ευρώ έχουν κατανεμηθεί στο EMFF για 5 χρόνια για να καταψύχονται τα ψάρια ενώ ε, το κόστος θα κατανεμόταν μεταξύ των οργανώσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ορισμένες ε, οργανώσεις ε, θεωρούν ότι πρέπει να παραμείνει η κατάσταση. Εγώ παραμένω ότι θα αναμένω ότι θα υπάρχουν ε, πολύ ουσιαστικές συζητήσεις στο θέμα αυτό κατά την υποβολή τροπολογιών όμως εγώ επιμένω ότι αν καταργηθεί η ελάχιστη τιμή παρέμβασης αυτό θα βοηθήσει τις οργανώσεις ε, για καλύτερες αγορές. Ε, ένα άλλο επίμαχο σημείο ε, ένα νόμφισιμο σημείο είναι το θέμα τη ετικετοθεσία. Το να δίνουμε στου καταναλωτέ σαφεί πληροφορίε, ευανάγνωστε για τα προϊόντα ελιάς και δατοκαλλιέργεια είναι κάτι ουσιώδε. Υπάρχει ανάγκη να καταργήσουμε τις διάφορες οικολογικές ετικέτες που εμφανίστηκαν με τα χρόνια ε, και αναφέρουν πόσο φιλικά είναι τα προϊόντα τους προς το περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να θέσει ίδια τους ελάχιστους κανόνες για ε, μια εθελούσια οικολογική ετικέτα θέτοντας τον πύχη πιο ψηλά από τους ε, υποχρεωτικούς κανόνες που διαπούν τώρα τον τομέα. Σε ό,τι αφορά τώρα τις πληροφορίες για τις ετικέτες πιστεύω ότι η ημερομηνία της εκφόρτωσης θα πρέπει να είναι υποχρεωτική και η ημερομηνία τη αλίευση ε, θα πρέπει να είναι κούσια. Η ποιότητα θα πρέπει να είναι ο κύριος παραγοντές για την ε, ετικετοθεσία και αυτό θα πρέπει να εξαρτάται και από τι τεχνολογικέ πτυχές όπως ο έλεγχο των περιβαλλοντικών συνθήκων, θερμοκρασία, υγρασία, μαζί και με μέτρα που αφορούν ε, τι διαδικασίε μεταποίηση και τα υλικά ε, πακεταρίσματος. Επίσης, ό,τι αφορά τα νοπά αλλά και τα καταψυγμένα ήδη χρησιμοποιείται, μάλλον απαιτείται νομοθεσία ε, και αναφέρεται ε, το αν ε, έχει ψυχθεί και αποψυχθεί ε, το προϊόν. Επίσης πρέπει να υπάρχει πλήρη συχνηλασιμότητα στο barcode. Σε ό,τι αφορά τώρα το προϊόντα του καλλιέργειας, η Κομισιόν έχει πει ότι σκοπεύει να παρουσιάσει ένα ξεχωριστό κανονισμό εν ευθέτω χρόνο, αλλά πάρα πολλοί από τον κλάδο είπαν ότι εξεπλάγησαν με αυτό, είπαν ότι οι σημερινοί κανόνες λειτουργούν ικανοποιητικά. Έτσι λοιπόν ε, ε, μια νέα νομική βάση θα πρέπει να αντικατοπτρίζει το status quo, τίποτα δεν πρέπει να γίνει που θα καταστήσει πιο δύσκολο ε, για τους μεταπιτές μας να έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα που χρειάζονται. Τώρα για την υδατοκαλλιέργεια υπάρχει καθολική ανάγκη να επεκτείνουμε την καλλιέργεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να καλύψουμε την μείωση των αποθεμάτων όπως ακούσαμε σήμερα 25% μόνο είμαστε αυτάρκης ε, σε ψάρια και προϊόντα και ε, καλλιέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι λοιπόν υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες ε, για επέκταση. Επαγγελματικέ οργανώσεις συμπεριλαμβανομένων και των οργανώσεων παραγωγών και των διαπαγγελματικών οργανώσεων και των ομοσπονδιών θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε δύο δεσμες μέτρων για να προωθήσουν τις δράσεις επικοινωνίας σε εθνικό και διεθνές πλαίσιο. Έτσι λοιπόν η δημιουργία να έχουμε ένα νέο Περιφερειακό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για την Δετοκαλλιέργεια πρέπει να υποστηριχθεί. Θα πρέπει να αποτελεί, πρέπει να έχουμε μία και μόνη οντότητα Ευρωπαϊκή Ένωση με έδρα και προσωπικό όπω υπάρχει για τα απελογικά ρακ, Περιφερειακά Γνωμοδοτικά Συμβούλια και θα πρέπει ε, να παγιώσουμε τα εφιστάμενα ρακ και να γίνουν πραγματικά γνωμοδοτικά συμβούλια για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Στίβενσον. Και ας περάσουμε τώρα στις ερωτήσεις, στο γύρο των ερωτήσεων. Καταρχήν τώρα Σκολομέρα από την Ισπανική Γερουσία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θα κάνω μία σύντομη εισαγωγή αναφερθώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Παππού Νέου για την ελεύθερη, ε, χωρίς δασμούς ε, εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, προϊόντων και σε εκείνη τη χώρα αλλιεύουν σκάφη Χωρί ε, χωρίς έλεγχο και ε, δεν υπάρχει σεβασμός των κανόνων προέλευσης. Ε, και εκεί στην Παππούα Γουινέκ φορτώνεται ψάρια από παντού και αυτά τα ψάρια μεταποιούνται σε κονσέρβες χωρίς να γίνονται σεβαστά και τα δικαιώματα εργασιακά. Πώ ε, λοιπόν στην ΕΑΚΟ ε, θα αντιμετωπιστεί ε, αθέμητο ανταγωνισμό προϊόντων τρίτων χωρών σε σχέση με το σεβασμό των περιβαλλοντικών συνδικών και των εργασιακών συνδικών και επίση για την ετικέτα που μιλήσατε εδώ, για του νέου κανόνε. Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω έχουμε προβλήματα ε, επιμελητία, ε, οργάνωση εδώ και έτσι λοιπόν ο υποχρεωτικό ε, χαρακτήρα τη ημερομηνία αλίευση. Γιατί έχουμε, παραδείγματο χάρη, κάποια σκάφη που αλλιεύουν και εκφορτώνουν την ίδια μέρα, ενώ κάποια άλλα που εκφορτώνουν μετά από τρει μέρε. Και αυτό θα σημαίνει ότι θα έχουμε πολλέ διαφορετικέ ημερομηνίε αλίευση και δεν νομίζω ότι είναι πρακτικό κάτι τέτοιο τέτοιο. Έτσι λοιπόν αυτό που προτείνεται είναι η ημερομηνία, να είναι η ημερομηνία της εκφόρτωσης. Αυτά Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τόρας. Επόμενη ερώτηση από τον κύριο Μπέν από τον Μπούντενστακ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λίγες παρατηρήσεις για το κεφάλαιο 4, ενημέρωση στους καταναλωτές. Είναι πολύ σημαντικό να είναι υποχρεωτικές οι ενδείξεις για το χρόνο αλίευσης, για να υπάρχει ανιχνευσιμότητα ε, του προϊόντος. Επίσης, ε, ε ψήξη, ε, και οι σχετικές διαδικασίες θα πρέπει να αναφέρεται αν υπάρχει επαν, επανειλημμένη ε, ψήξη και να είναι σαφές αν ένα προϊόν ε, μεταποιήθηκε νοπό ε, ή αποψυγμένο. Επίσης, η εμπορική ονομασία θα πρέπει να αναφέρεται όταν είναι μεταποιημένα τα προϊόντα. Είναι σημαντικό αυτό και επίσης η επιστημονική ονομασία θα αναφέρεται έτσι ε, ανεξάρτητα από, το, από, το, από τη μεταποίηση. Επίσης, ελάχιστα, με ελάχιστο μέγεθος εμπορίας. Αν έχουμε μία ρύθμιση σχετικά με την εκφόρτωση και αν υπάρχει απαγόρευση των απορρίψεων, τότε δεν έχει νόημα το ελάχιστο μέγεθος εμπορίας εν τη αυτή περίπτωση πρέπει να βρούμε μια λύση για το πώς θα ε, προβλέπονται κυρώσεις ε, ε, όταν εκφορτώνονται μικρά ψάρια. Αλλιώς δεν έχει νόημα η κοινή οργάνωση της αγοράς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Μιράντα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε διάφοροι εκπρόσωποι από τα Εθνικά Κοινοβουλία αλλά και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο έκαναν αναφορά σε μια αεροστεχνική αλία αλλά και σε, που να είναι βιώσιμη αλλά και σε βιώσιμη δεδοκολιέργεια. Εμείς στην Γαλλική έχουμε την εκτροφή ε, μηδιών σε φυσικές συνθήκες ε, και στο πλαίσιο της ε, ΚΟΑ η ποιότητα που διασφαλίζεται προέρχεται από τι γεωγραφικέ ενδείξει, προστατευμένε γεωγραφικέ ενδείξει και ονομασίες προέλευση ε, δεν ε, σημαίνει κάτι ιδιαίτερο. Έτσι λοιπόν πρέπει να υποστηρίξουμε αυτές τις ονομασίε προέλευση και αναγνώριση τη Ευρωπαϊκή παραγωγής με μέτρα που να εφαρμόζονται από τις οργανώσεις παραγωγών τροποποιώντα το άρθρο 11 Προ ε, την εξή κατεύθυνση. Να πούμε ότι η πρόθεση των προϊόντων τη ιδετοκαλλιέργεια, εκμεταλλευόμενη την ικανότητα πιστοποίηση, την δυνατότητα πιστοποίησης, ιδίω αυτών των ονομασιών προέλευση, όπω για τα μύδια, θα έπρεπε να υποστηριχθεί από τις διαπεγγελματικές οργανώσεις ε, που είχαν ε, μάλιστα προωθήσει αυτές τις προστατευόμενες ονομασίες. Ε, δεν, δεν γίνονται πάντοτε υποστήριξή τους ούτε σε περιφερειακό ούτε σε κρατικό επίπεδο και εμείς λυπούμαστε που υπάρχει πολιτική για περικοπές και Θέλουμε να αναφέρουμε αυτή τη δυνατότητα ότι η μεταποίηση και θέση εμπορία των προϊόντων αλίας και δατοκαλλιέργειας συμπεριλαμβάνεται μέσα ε, σε αυτή την έννοια της ευρωπαϊκής προστασίας. Δηλαδή να προστατεύσουμε αυτό που υπάρχει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πίνης από τη Λιθουανία. Ευχαριστώ. Ε, οι καταναλωτές πρέπει πάντα να γνωρίζουν τι αγοράζουν. Είναι υποχρεωτική η ενημέρωση, αλλά και εκεί δεν πρέπει να βιαστούμε. Δεν μπορεί να τα γράψουμε όλα σε μία ετικέτα. Ε, άλλωστε για όλα υπάρχει ένα τίμημα. Ο κανονισμός προβλέπει περισσότερες πληροφορίες, καλύτερη ενημέρωση. Ε, έχω κάποιες... Ε, αμφιβολίες σε σχέση με τις εξαιρέσεις. Γιατί αν, για παράδειγμα, πρέπει να αναφέρεται το είδος του ψαριού στα προϊόντα που, που έχουν συστατικό το ψάρι, τότε η παραγωγή θα έχουν μεγάλα προβλήματα. Θα τους δημιουργήσουμε πρόβλημα. Αν δηλαδή ζητάμε υπερβολικά πολλές πληροφορίες, τότε το γραφειοκρατικό βάρος, το φορτίο αυτό είναι πολύ μεγάλο και θα ε, δημιουργήσει και ε, αυξημένες δαπάνες. Και αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα σε πολλούς τομείς. Ευχαριστώ κύριο Γκαρσία. Ευχαριστώ πρόεδρε και πάλι. Για να μην επαναλάβω ορισμένα θέματα που τέθηκαν άκουσα και πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε με το πώς ε, θα κάνουμε πιο αποδοτική την αλευτική δραστηριότητα ε, τώρα, εγώ θα ήθελα να μου πει ο συζητητή αν συμφωνεί με τα εξή. Καταρχήν, για να αποφύγουμε η ελευτική δραστηριότητα να προσανατολιστεί στην αλία των Εκτιδίων, το άρθρο 8, ε, δάφιο Β, θα πρέπει να εμποδίζει να εκφορτώνονται πάνω από το 25% του συνόλου των ανεπιθύμητων ε, αλευμάτων από τα εμπορικά είδη. Ε, τώρα, σε ό,τι αφορά με το Ταμείο, το άρθρο 38, η δημιουργία του Ταμείου θα πρέπει να επιτρέψει τη συνεισφορά δημοσίων και ιδιωτικών κονδυλίων. Και τέλος, ε, στο άρθρο 45, όπου γίνεται λόγος για εκούσια πρόσθετη ενημέρωση, πέρα από τις υποχρεωτικές πληροφορίες, εμείς θεωρούμε ότι τόσο οι περιβαλλοντικές πληροφορίες ε, όπως και η ηθική ε, θα πρέπει να καταρτίζονται βάσει κάποιων ελάχιστων προτύπων που θα καταρτίζονται στην ε, νομοθεσία της Ένωσης και δεν θα πρέπει να παρουσιάζονται κούσεις πληροφορίες που να μην μπορούν να επαληθευτούν. Θα ήθελα να μου πείτε αν τις προτάσεις αυτές τις θεωρείτε ότι βελτιώνουν την ε, αποδοτικότητα των ε, λευτικών επιχειρήσεων ε, και θα ήθελα να μου πείτε, κύριε Σιγητά, αν θεωρείτε σκόπιμο αυτό που δεν επιτρέπεται να θέσει στην εμπορία ένας Ευρωπαίος ψαράς να μην επιτρέπεται να το θέσουν σε εμπορία και οι αλείς των τρίτων χωρών και αναφέρομαι και σε προϊόντα που έρχονται στη δική μας κοινοτική αγορά χωρίς να γίνονται σεβαστές οι περιβαλλοντικές και εργασιακές προϋποθέσεις και συνθήκες που απαιτούμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριο Παπαγεωργίου. Θέλω να αναφερθώ σε τρία θέματα. Το πρώτο αφορά την πρόβλεψη για σήμαση των εμπορικών ε, σημάσεων προϊόντων ιδιωτοκαλλιέργειας από τρίτες χώρες, όπου επιβάλλεται η χώρα αναφοράς, να αναφέρει τη χώρα αναφοράς για το τελευταίο τρίμηνο εκτροφής. Θεωρώ όμως ότι αυτές οι πληροφορίες είναι εθελοντικές, εισάγονται πάρα πολλά ψάρια από τρίτες χώρες, Παγκάσους, Βιετνάμ κλπ. Τα οποία, ε, για τα οποία ο κοινωνικός κανονισμός δεν αναφέρει τίποτα. Στην ουσία ο έλεγχος γίνεται μόνο στο συσκευαστήριο. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες για τις συνθήκες που παράγονται αυτά τα ψάρια. Το δεύτερο που θέλω να πω, το ανέφερε η συνάδελφος από την Ιταλία και αφορά τα μύδια, ιδιαίτερα τα, ιδιαίτερα τα μύδια. Υπάρχει μια στάση των ε, εμπόρων, των εισαγωγέων, εξαγωγικού προϊόντα από τη χώρα μου τουλάχιστον είναι, όπου ό, κατά, το, κατά την αντίληψή τους σε πολλέ των περιπτώσεων χαρακτηρίζουν ότι έχουν επιβαρθεί από μια ασθένεια όταν θέλουν δηλαδή να ρίξουν τι τιμέ ή να εκμεταλλευτούν του παραγωγού έτσι, ε, χαρακτηρίζουν ας πούμε, επιβαρημένη την κατάσταση των μηδιών, επιστρέφουν παραγγελίες, καταστρέφονται επιχειρήσεις. Τουλάχιστον 100 επιχειρήσεις στη χώρα μας έχουν καταστραφεί εξαιτίας αυτών των λόγων από εξαγωγές σε χώρες, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όντως εκεί πρέπει να δοθεί μεγαλύτερο βάρος στις ομάδες παραγωγών και στις υποδομές και στη χρηματοδότηση για τον έλεγχο για να μπορούν αυτοί οι παραγωγοί να προστατεύσουν το προϊόν από τις εμπορικέ λογικέ που καθυλώνουν αυτά τα προϊόντα. Και το τρίτο που θέλω να πω αφορά και αφορά και το τέταρτο θέμα, η θαλάσσια στρατηγική που θα συζητήσουμε, αφορά α, ε, στάση μεγάλων χωρών, ιδιαίτερα στη Μεσόγειο. Για παράδειγμα, η Τουρκία έχει πάρα πολλέ επιδοτήσει εξαγωγές ψαριών και έχει και πάρα πολύ ισχυρού δασμού. Ψαρεύουμε στην ίδια θάλασσα, δίπλα-δίπλα τα καίκια. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι πρέπει να κάνει με αυτή την, με αυτή την κατάσταση. Δεν μπορεί να συνεχιστεί δηλαδή να έρχονται ψάρια στη χώρα να δημιουργούν αθέμητο ανταγωνισμό στη χώρα μας, να καταστρέφονται ε, αλληλείς και από την άλλη μεριά όταν πάμε να εξάγουμε εμείς θέτουν πάρα πολλοί ισχυρού φραγμού, Γίνεται κύρια με την Τουρκία αλλά και άλλε χώρε. Νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί όπως και ε, δεν μπαίνω στο άλλο θέμα αφορά και τη θαλάσσια στρατηγική. Τι πολιτική αηφορία θα εφαρμόσουμε στη θαλάσσια στρατηγική όταν οι άλλες χώρες για παράδειγμα εμείς σαν ευρωπαϊκή πολιτική σαν κοινή οργάνωση αλληλευτικής πολιτικής έχουμε στάνταρς και προοπτικές αλλά η θάλασσα είναι ενιαία μολύνεται ή δεν μολύνεται, προστατεύεται ή προστατεύεται όχι σε μια ενότητά της έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η προσέγγιση και πρέπει να τη δούμε και στο άλλο θέμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Στιβένσον έχει το λόγο για να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να συνοψίσω κάποιες ε, απαντήσεις ε, μαζί. Ετικετοθεσία. Είχαμε ένα μεγάλο κανονισμό σχετικά με την ενημέρωση των καταναλωτών που πέρασε από τη δεύτερη ανάγνωση και είχε μια δύσκολη διαδικασία στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου όπου κοντέψαμε να αποτύχουμε όπως ε, ο κανονισμός για τα καινούργια ε, τρόφιμα που απέτυχε και ξαναγυρίσαμε στον κανονισμό τον παλιό του 99 και δεν θέλαμε να πετάξουμε στα σκουπίδια τριών χρόνων δουλειά για την ενημέρωση των καταναλωτών, βρήκαμε μια συμβιβαστική λύση στο τέλος που ε, προβλέπει ότι θα ε, ζητήσουμε αξιολόγηση αντίκτυπου από την ε, Κομισιόν για τις τικέτες για την προέλευση, για τα αμυκτά προϊόντα, τα επεξεργασμένα, τα κονσερβοποιημένα, τα κατεψυγμένα, εκεί όπου για παράδειγμα έχουμε μια πίτσα με διαφορετικά είδη κρέατος, είναι δύσκολο να βάλουν στην ετικέτα τη χώρα προέλευσης όλων των διαφορετικών κρεάτων, γιατί αλλάζουν τα προϊόντα πολύ γρήγορα. Και έτσι είναι δύσκολο να ζητήσουμε από το εργοστάσιο να αλλάξει την ετικέτα για να αντικατοπτρίσει αυτές τις αλλαγές. Και πολλοί ήρθαν και μου είπαν ότι μετά από όλα αυτά και έχοντας ζητήσει από την Κομισιό να κάνει αντίκτυπο αξιολόγηση, αξιολόγηση αντίκτυπου, τώρα ε, υποβάλλεται νέες προτάσεις για την ετικετοθεσία και θα ζητήσετε από τους ε, παραγωγούς ε, με ε, τροφίμων, κονσεργοποιημένων κλπ, να ζητήσουν ε, ε, ε, στην ετικετοθεσία τη χώρα προέλευσης. αυτό δεν μπορεί να γίνει. Και κάποιοι μεταποιητές και κάποιες οργανώσεις παραγωγών μου είπαν ότι θα πρέπει να το διαγράψετε όλο αυτό το εδάφιο. Έκανα σήμερα το πρωί μια μεγάλη συζήτηση με την Κομισιόν για τα θέματα αυτά. Πάντως κάποια ζητήματα που αφορούν την ετικετοθεσία, τα άρθρα δηλαδή ε, για την ε, ετικετοθεσία, την επισήμανση την έκθεση για την κοινή οργάνωση της αγοράς, είναι σημαντικά, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την οικοσήμανση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό με ενδιαφέρει πολύ, και το συζήτησε και με την Επίτροπο Δαμανάκη. Καλύπτει κάποια ε, θέματα που έθεσαν οι ερωτώντες σχετικά με τους ίσους κανόνες του παιχνιδιού, ε, μεταξύ εισαγωμένων προϊόντων αλίας και υδατοκαλλιέργειας και εκείνων που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, οι παραγωγοί μας θα πρέπει να πληρούν πολύ αυστηρά κριτήρια και πολλοί λένε ότι παρόλο που ε, στηριζόμαστε στο 60% των καταναλωμένων προϊόντων από εισαγωγές δεν ισχύουν τα ίδια πρότυπα για αυτές τις εισαγωγές. Και βεβαίως ο κύριος Παπαγεωργίου είπε και το καταλαβαίνω ότι χρειάζονται μέτρα για να σταματήσουμε τις εισαγωγές κάποιων τέτοιων προϊόντων αν δεν πληρούν τα κριτήριά μας. Αλλά κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει ε, χωρίς να παρέμβει ο ΠΟΕ. Θα μπορούσε να γίνει αυτό αν είχαμε ε, προαιρετική σήμανση, ε, οικοσήμανση, ε, δηλαδή να φαίνεται ότι είναι ένα βιώσιμο προϊόν από βιώσιμα αλλιεύματα με, μεγάλη, με υψηλή κοινωνικο-οικονομική σημασία ε, και ορισμένα από αυτά τα θέματα δεν καλύπτονται από τη σημερινή ετικετοθεσία. Θα μπορούσαμε με την οικοσήμανση να, έχουμε να προσφέρουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους ε, καταναλωτές και εκείνοι που θα ήθελαν να κάνουν εξαγωγές ε, τρίτη θα έπρεπε να ζητήσουν το, την οικοσήμανση και τότε θα έπρεπε να πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις, τα ίδια πρότυπα όπως εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορούσε λοιπόν να γίνει με αυτόν τον τρόπο ε, αυτό στα πλαίσια της έκθεσης της ΚΟΑ, για την ΚΟΑ. Τώρα, άλλα θέματα που αφορούν, ε, ας πούμε, την ημερομηνία της εκφόρτωσης σε σχέση με την ημερομηνία αλίευσης. Η Κομισιόν στην πρόταση προτείνει η ημερομηνία αλίευσης να είναι υποχρεωτική. Εγώ ε, ήμουν πολύ ευγνώμων στους συναδέλφους από τη Γαλλικία που μου έδωσαν πολλά στοιχεία, γιατί για πρώτη φορά πήγα, ε, πήγα στη Γαλλικία και σε άλλα μέρη. Και ε, μου είπαν ότι οι μικροί αλείς που βγαίνουν στη θάλασσα και επιστρέφουν με νοπά αλλιευμένα ψάρια την ίδια μέρα, εκφορτώνουν ψάρια με την, που είναι το ίδιο φρέσκα, όπως μια τράτα η οποία βγαίνει και βάζει στον πάγο και γυρίζει μετά από μια ή δύο εβδομάδες ε, με τα ψάρια. Δεν υπάρχει διαφορά στην φρεσκάδα των ψαριών. Ο μικρός ψαράς μπορεί να μην έχει καθόλου πάγο στο σκάφος και τα αλλιεύματά του καμιά φορά μπορεί να μην είναι τόσο φρέσκα. Άρα η ημερομηνία της εκφόρτωσης πρέπει να είναι υποχρεωτική και της αλλιεύσης προαιρετική. Ε, Μπορεί ε, να θέλει ο μικρός αλλιέας να βάλει την ημερομηνία αλλιεύση γιατί του δίνει πλεονέκτημα στην αγορά, αλλά είναι, δημιουργεί σύγχυση στον καταναλωτή να λέει «Ε, εδώ είναι ένα ψάρι που είναι ηλικία μια ημέρα, έχει αληθεί πριν από μία έρα μία μέρα, ενώ το άλλο πριν από δύο εβδομάδες και ε, βγάζει το συμπέρασμα ότι τη μια μέρα μπορεί να είναι πιο φρέσκο ψάρι, ενώ κάτι τέτοιο μπορεί να μην συμβαίνει. Άρα λοιπόν ε, της εκφόρτωσης ημερομηνία πρέπει να είναι υποχρεωτική. Επίσης, για τα κατεψυγμένα και τα μεταποιημένα προϊόντα, το να έχουμε τρεις διαφορετικέ ημερομηνίε, ε, γιατί ήδη επιμένουμε να υπάρχει ημερομηνία της ψήξης, ε, το best before, ε, καταναλωθεί μέχρι και τώρα θέλουμε και την ημερομηνία εκφόρτωση και τη αλλίευση. Τι θα τα κάνει όλα αυτά ο καταναλωτή, τρει διαφορετικέ ημερομηνίε. Δηλαδή θα σκεφτεί ότι αυτό το κατεψυγμένο προϊόν, εδώ η ημερομηνία αλλίευση ήταν πριν από δύο χρόνια και δεν πρόκειται να αγοράσουν ψάρια, θα απορθαρρυνθούν και έτσι θα καταρρεύσει η αγορά. Οπότε χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή στο πώς θα προσεγγίσουμε όλο το θέμα της ε, επισήμανσης στα προϊόντα της ετικετοθεσίας. Και χαίρομαι και ευχαριστώ όλους όσους παρενέβησαν. Τώρα, ο συνάδελφος από την Ισπανική Γερουσία που νομίζω ότι έφυγε τώρα, ε, ρώτησε για το FTA της Νέας Ουινέας. Ε, έχουμε με τα προβλήματα αυτά της εμπορικής, Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου, τη συμφωνία. Εδώ ο κύριος Καντέκ είπε ότι ελπίζουμε ότι ε, οι μικροί βιοτέχνες αλληλείς στην Παππούα Νέου Γουινέα θα έχουν την ευκαιρία έτσι να ε, βελτιώσουν τα εισοδήματά τους. Όταν υπογράψαμε τη συμφωνία βέβαια, ήρθαν οι Κινέζοι, έφτιαξαν ένα τεράστιο εργοστάσιο μεταποίησης με Κινέζους εργαζόμενους, όχι ντόπιου, και άρχισαν να εκφορτώνουν ε, κινέζικα ψάρια που θα τα μεταποιούσαν στην Παπουασία Νέα Γουινέα και θα τα εισήγαγαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, με βάση τους κανόνες της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών. Ε, ε, αυτό δεν συνάδει με το νόημα της Συμφωνίας και πλουτίζουν οι ήδη ευημερούσε κινέζικε εταιρείε. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε πάρα πολύ για το πώ αντιμετωπίζουμε αυτέ τι συμφωνίε ελευθέρων συναλλαγών. Μου φαίνεται τα είπα όλα, κύριε Πρόεδρε, ή τα περισσότερα. Ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στο τελευταίο πάνελ που έχει να κάνει με τις προοπτικές ε, του Νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλίας. Στην περίπτωση αυτή το λόγο έχει ο κύριος Καντέκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τους θαραλέους ε, που είναι ακόμη εδώ με στην αίθουσα από τα Εθνικά Κοινοβούλια και επέλεξαν να έρθουν ε, να συζητήσουν μαζί μας ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα είμαι σύντομος γιατί έχουμε μεγάλη καθυστέρηση, Πρόεδρε, σε σχέση με το πρόγραμμα. Θα ήθελα να εξηγήσω το χρονοδιάγραμμα που προτείνουμε. Παρουσίαση στις 24 Απριλίου του σχεδίου, στις 19 ε, Σεπτεμβρίου επανεξετάστηκε, 28 Νοεμβρίου Επιτροπή και Ιανουάριος 2013 θα ψηφιστεί ε, το σχέδιο στην Ολομέλεια. Ε, το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Θάλασσα και για την Αλληλία είναι προφανώς, απορρέει προφανώς από τον ισχύοντα κανονισμό. Η χρηματοδότηση θα είναι συνάρτηση του περιεχομένου του βασικού κανονισμού. 6,7 δις για την περίοδο 2014 έως 2020 είναι η πρικοδότηση του Ταμείου στα πλαίσια του κοινού στρατηγικού πλαισίου, στα πλαίσια δηλαδή της πολιτικής συνοχής, όπως μας είπαν και οι συνάδελφοι. 376 ε, περίπου εκατομμύρια ευρώ για το Ταμείο. Δηλαδή, είναι αμεληταίο το ποσό σε σχέση με το συνολική προκοδότηση για την πολιτική συνοχή, αλλά αυτά έχουμε. Είναι σίγουρο ότι θα απηχεί ε, η προκοδότηση του Ταμείου το περιεχόμενο του νέου βασικού κανονισμού. Θα ήθελα όμως ήδη να σας κοινοποιήσω κάποιες σκέψεις που έχω κάνει, κάποιες παρατηρήσεις Πρώτον, θα ήθελα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας, το ΕΤΑ, ε, να είναι χρήσιμο για τους αλληλείς ε, και όχι για την ανακύκλωσή τους και την αλλαγή δραστηριότητας ε, ε, δεν θέλω να είμαι υποτιμητικός, ε, αλλά δεν θέλω οι ε, να αρχίσουν να πουλάνε πίτσες ε, ή να ανοίξουν ξενώνες. Και το, δεν το λέω υποτιμητικά. Έχω, τρέφω μεγάλο σεβασμό για όσους πουλάνε πίτσα ή έχουν ξενώνες. Εννοώ ότι κάνουμε κάποιες προσπάθειες για να σώσουμε την αλία και τους αλείς. Ε, ταυτόχρονα θα πρέπει να συμβάλλουμε στη διατήρηση των αποθεμάτων. Νομίζω όλοι θα συμφωνήσουν. Αυτές είναι οι δύο βασικές συνιστώσεις του ζητήματος. Ε, ε, υπάρχουν επίσης ενδιαφέροντα στοιχεία στη νέα πρόταση. Παραδείγματο χάρη η θέση της υδατοκαλλιέργειας, ε, γιατί το είπα και προηγουμένως, ξεχνάμε ότι είτε μιλάμε για την ΚΟΑ, Κοινή Οργάνωση Αγοράς, είτε για το βασικό κανονισμό, είτε για οτιδήποτε, ε, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τι συνθήκε της Λισαβόνα και μετά ισχύει η διαδικασία τη συναπόφασης. Ε, λοιπόν, θα αποφασίσει και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ε, για το πεπρωμένο της πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, θεωρώ ότι είναι ενδιαφέροντα τα στοιχεία σε σχέση με την υδατοκαλλιέργεια, το ίδιο και τα νέα στοιχεία για τι οργανώσει παραγωγών και τις επαγγελματικέ οργανώσει, Είναι ενδιαφέρουσε οι προτάσει τη Επιτροπή. Τώρα, για να υπάρξει ενώτερη συνεργασία ανάμεσα στου επιστήμονε και Και αυτό μου φαίνεται καλή ιδέα. Ε, σε σχέση τώρα με τις ε, εντόπιες ομάδες ε, δράσης, όπως λέγαμε πριν, ο άξονας 4 δηλαδή, ε, αυτού συμφωνούμε. Αλλά στο αντίστοιχο σημείο 1 έχουμε κάποιες διαφωνίες διότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε προφανές αυτό διάφορους τομείς της αλληλευτικής δραστηριότητας αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και τα αναπτυξιακά θέματα και τα θέματα ανταγωνιστικότητας. Ε, ε, ε, σε αυτά θα πρέπει να εστιάσουμε και όχι στην ανακύκλωση σε εισαγωγικά των αλλιέων. Δηλαδή δεν έχουμε λάβει εντολή για να επαναπροσανατολιστούν αυτοί οι επαγγελματίες προς κάποιο άλλο κλάδο. Λάβουμε την εντολή να αναβαθμίσουμε τον αλλιευτικό κλάδο, τον ίδιο. Σε σχέση τώρα με την εισρωή νέων ανθρώπων στον κλάδο θα έπρεπε να διευκολύνουμε την προσφασή τους ε, όποιο και αν είναι αυτό το επάγγελμα, έτσι, και κυρίως για την ερασιτεχνική και την παράκτια αλία, χρειάζεται ιδιαίτερη υποστήριξη για την σύσταση μικρών επιχειρήσεων ε, και για την κατάρτισή τους. Πιστεύω ότι ε, κάτι που είναι ε, απαραίτητο είναι ε, ο μηχανισμός στήριξης ε, για όσους πλήττονται από την κρίση. Σε κανένα σημείο δεν αναφέρεται σε αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, ε, επαναλαμβάνω, θα με συγχωρέσετε, αλλά είναι σημαντικό. Θέλω να ανανεωθεί, ε, να εξυγχρονιστεί ο στόλος και αυτή, αυτό το πριμ για τον παροπλισμό του στόλου θα πρέπει να συνεχιστεί. Είναι απαρχαιωμένος ο στόλος, σας είπα, 27 χρονών είναι κατά μέσο όρο κάθε σκάφος και γίνεται επικίνδυνο για λόγους ασφάλειας, ε, για ε, λόγους ε, ενέργειας, κατανάλωση δηλαδή δίζελ, εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Είναι απαραίτητο να ανανεωθεί ο στόλος γιατί αλλιώς σε 15 χρόνια θα έχουμε κάποιες μεγάλες βιομηχανικές στράτες και τίποτε άλλο. Θα εξαφανιστούν τα υπόλοιπα μικρά σκάφη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς επενδύσεις προτείνει κάτι μόνο, αποκλειστικά και μόνο για την απαγόρευση των απορρίψεων. Ε, εντάξει, ναι, είναι καταπληκτική ιδέα, τελικά όλοι συμφωνούν και εγώ το ίδιο. Όμως σήμερα γνωρίζουμε ότι από τεχνικής πλευράς δεν είναι εφικτή αυτή η λύση, άρα χρειαζόμαστε συνοδευτικά μέτρα για να καταλήξουμε τελικά στις μηδενικές απορρίψεις ε, μελλοντικά. Ακούγοντα την κυρία Δαμανάκη μου δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι έχει μετεξελιχθεί η αρχική πρόταση. Δεν επιδιώκει τη μηδενική απόρριψη όπω ήταν στην αρχή, μου φαίνεται. Ε, αυτό θα ήταν θετικό. Χρειαζόμαστε επίσης ρυθμιστικούς μηχανισμούς ε, πριν για την αποθήκευση. Προτείνει η σταδιακή κατάργησή, τη τώρα, κατάργησή του συγγνώμη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ρυθμίζονται οι τιμέ τη αγορά με κάποιο τρόπο. Επίση, στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, απουσιάζει οποιαδήποτε μνήμα στην ε, ε, περιφερειοποίηση. Η κυρία Πατράου Νέβε ήταν συγγήτρια στην, για την Πράσινη Βίβλο και θυμάμαι ότι έλεγε στην Πράσινη Βίβλο ότι επιδιώκουμε μια ουσιαστική περιφερειοποίηση. Δεν νομίζω ότι θα το αμφισβητήσει κανεί. Δυστυχώ, όμω, δεν βλέπουμε καμία σχετική μνήμα. Αυτό θα ρύθμιζε πολλά προβλήματα. Ε, δηλαδή βρισκόμαστε αντιμέτωποι με κάποιου νομικού φραγμού που προτάσει η Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εντάξει, όντω σε σχέση με τον βασικό κανονισμό υπάρχουν νομικά κολλήματα που σχετίζονται με τι διατάξει περί ενιαία αγορά. Αλλά δεν επαρκεί αυτό και σα έλεγα προηγουμένω, δεν χρειάζεται τώρα να μακρηγορήσω και να σχολιάζουμε μόνο αυτό το θέμα ε, των μεταβιβάσεων, μεταβιβάσιμων παραχωρήσεων έχουν γίνει κάποιες ε, Προτάσει που οδεύουν προ τη σωστή κατεύθυνση, αλλά έχω την εντύπωση ότι χρήζει τεχνική επεξεργασία. αυτή η πρόταση για τι μεταβιβάσιμε παραχωρήσει. Λοιπόν, για να κλείσω την παρέμβασή μου, η πρεκοδότηση του Ταμείου, σα είπα, θα είναι απόλυτη συνάρτηση του περιεχομένου του νέου βασικού κανονισμού. Άρα θα πρέπει να στείλετε όλοι σα τροπολογίε και θέσει ε, για το σχέδιο του νέου κανονισμού. Ε, θα κλείσω και είμαι στη διάθεση αν έχετε ερωτήσει. Ευχαριστώ. Να περάσουμε στις ερωτήσεις. Καταρχήν, ο κύριος Νάουντινς από την Λετωνία. Ευχαριστώ. Κύριε Καντέκ, αγαπητοί συνάδελφοι, θα κάνω ένα σχόλιο που έχει να κάνει σε σχέση με τη θέση της Λετωνίας ε, για το αν υποστηρίζουμε αυτό το μέσο. Είμαστε καταρχήν σίγουροι ότι πρέπει να υποστηρίξουμε μέσα εξεχρονισμού για να έχουμε και ενεργειακή αποδοτικότητα αλλά και ασφάλεια στην αυσιπλοεία. Έτσι λοιπόν ε, θα ε, υποστηρίζαμε να αντικαταστούν μηχανές ε, με μηχανές που είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον και λιγότερο ενεργοβόρες. Όμως ε, το ότι αναφέρθηκε ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια για την αντικατάσταση των μηχανών. Ε, πραγματικά αυτό αντίκειται στους στόχους που έχουμε, τους περιβαλλοντικούς. Ε, δεύτερον, σε ό,τι αφορά τώρα τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας και τη σχετική ενίσχυση, θα πρέπει να δοθεί ενίσχυση και στην διαδικασία παραγωγής για να έχουμε μεγαλύτερη προσθέμενη αξία έτσι ώστε οι μεγάλες εταιρείε ε, μεταποίησης ε, αυτοί που απασχολούν ε, πάρα πολλούς στον κύκλο παραγωγής να μην υπερβαίνουν κάποια κατόφλια και θα πρέπει γιατί να λαμβάνουν ε, τελικά την ίδια ένταση υποστήριξης ενίσχυσης όπως και μικρές επιχειρήσεις. Ε, τέτοιες ε, εταιρείε παρέχουν δουλειά σε ανθρώπους που κατοικούν σε περιοχές που εξαρτώνται από την αλευτική βιομηχανία. Και επίση ε, θα ήθελα να απευθυνθώ στην Επιτροπή Ελία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που οργανώσατε αυτή την εκδήλωση σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τίσκλιν από τη Σουηδία. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κύριο Καντέκ. Όταν ε, συζητούμε το θέμα των ευρωπαϊκών θαλασσών ε, και ε, συζητούμε το θέμα του νέου ταμείου θα πρέπει να διασφαλίσουμε τη συνοχή. Ακόμη και αν μιλάμε για την υποστήριξη μέσω οικοσυστημικής προσέγγισης θα πρέπει να κατανοούμε στην πραγματικότητα τι συμβαίνει. Από σουηδικής πλευράς θεωρούμε ότι η περιβαλλοντική βιωσιμότητα είναι εκ των όνου για να να επιτύχουμε την οικονομική βιωσιμότητα. Επίσης θεωρούμε, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, ε, ε, να ε, μείνουμε στο στόχο για το MSY μέχρι το 2015. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε να συνεχίσουν να ψαρεύουν οι αλληλείς. Από πλευράς μας ε, ξεκάθαρα τέτοιου είδους ε, επιδοτήσεις ε, που αυξάνουν τις θέσεις απασχόλησης και διασφαλίζουν την περιβαλλοντική διασημότητα... είναι οπωσδήποτε προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει να βρούμε φυσικά μια ισορροπία. Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε μόνο στην πλεονάζουσα ικανότητα. Πιστεύω ότι έχουμε περιθώριο λιγμών, μπορούμε να κάνουμε θετικές δράσεις και διάφορους υποκλάδους της αλίας, όπως παραδείγματος χάρη η υδατοκαλλιέργεια και ίσως χρειάζεται μια διαφοροποίηση για να υπάρξει καλύτερη συνεργασία τώρα που συστάθηκε και το νέο ταμείο κυρίως για τη μεταποίηση, για τη βιομηχανία, ε, συγγνώμη, για την αλία μικρής Ε, Πρέπει να όλοι να αντιληφθούμε ότι επικρατούν ιδιαιτερότητες σε αυτούς τους υποκλάδους και να δώσουμε μια ικανοποιητική απάντηση. Ε, είμαστε υπέρ φυσικά της ολοκληρωμένης ε, θαλάσσιας ε, πολιτικής και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η οδηγία σχετικά με τα ύδατα και τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων που συζητείται ταυτόχρονα με το νέο βασικό κανονισμό για την αλία. Χρειαζόμαστε σαφείς στόχους. Λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα στηρίξει ολόκληρο τον κλάδο το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο θάλασσας ε, και αλίας ε, και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει συνεργασία ανάμεσα σε όλους τους παράγοντες ε, του επαγγελματικού αυτού κλάδου. Ευχαριστώ, κυρία Τόβεν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ, κυρία Καντέκ. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Έχω μια ερώτηση. Έχετε δει επιτάπητο στην ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή τις ε, γνωμοδοτήσεις των κρατών μελών σε σχέση με τις δράσεις ε, του Ταμείου Αλίας, του σημερινού. Δηλαδή, ε, αναφέρομαι στις προτεραιότητες ε, των προγραμμάτων ή στις διαδικασίες. Να μας πείτε ποια είναι τα κείμενα που ισχύουν και αυτά που δεν λειτουργούν. από το Γαλλικό Κοινοβούλιο, επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ. Εδώ και 20 χρόνια η κοινή Λευτική πολιτική ε, χρηματοδοτείται από ένα ειδικό ε, μέσο για την αλία, το μέσο προσανατολισμού αλίας, το οποίο είχε πρικοδότηση 4,1 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2000-2006 και μάλιστα χρηματοδοτήθηκε και για την κατασκευή πλοίων, ε, ενώ είχαμε κατόπιν 3,8 εκατομμύρια για το 2007-2013 και τώρα μας ανακοινώνεται ένα ταμείο για τη θάλασσα και την αλία όπου έχουμε κάποια ερωτηματικά ε, τι ακριβώς θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από αυτό το νέο ταμείο. Το Ταμείο Περσανατολισμού Αλίας ε, ήταν αφιερωμένο αποκλειστικά στην Αλία, στους Αλείς και στα εργαλεία παραγωγής. Το 2007 το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας κατήργησε την ενίσχυση για τα εργαλεία παραγωγής ε, για να προωθήσει περισσότερο τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων, δηλαδή την μεταποίηση των προϊόντων ή τον τουρισμό. Όμως ε, αυτή τη φορά με το σχέδιο για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας ε, προχωρούμε σε ένα άλλο επίπεδο και αν δούμε τον κανονισμό βλέπουμε ότι το αντικείμενο του Ταμείου θα ήταν να προωθήσει μια βιώσιμη αλία και υδατοκαλλιέργεια αλλά και να προωθήσει μια ισορροπημένη ανάπτυξη της επικράτειας στις ζώνες που είναι εξαρτημένες από την αλία και να ευνοήσει την εφαρμογή της αλληλευτικής πολιτικής Ένωσης συμπληρώνοντας την πολιτική συνοχής. Αυτό που θα θέλαμε είναι, μπορούμε να έχουμε δεσμεύσεις ότι το τμήμα των κονδυλίων για την αλία θα είναι ανώτερο από ε, το κονδύλι που είχαμε για το προηγούμενο Ταμείο Αλίας. Δηλαδή, πού θα σταματήσει η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, η χρηματοδότηση ε, των ε, παράκτητων περιοχών από ποιον θα γίνει τώρα η ποικιλομορφία, ε, μάλλον η βιοπικιλότητα του θαλάσσιου βυθού ή της κλωρίδας και της πανίδας λαμβάνονται υπόψη. Μπορούμε να κατανοήσουμε τους λόγους μιας τέτοιας εξέλιξης, αλλά παρόλα αυτά αναρωτιόμαστε ποιος θα είναι ο αντίκτυπος στα οικονομικά μέσα που θα ε, αφιερωθούν για την αλευτική πολιτική αυτή καθ' αυτή. Αυτό είναι το ερώτημά μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νίλουγκ από τη Φιλανδία. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστούμε κύριε Καντέκ. Ήταν πολύ καλή και σαφέστατη η παρουσίασή σας. Θα ήθελα να κάνω τέσσερις παρατηρήσεις ε, σε αυτήν την τόσο σημαντική συζήτηση. Ε, στο βόρειο τμήμα της Ευρώπης υπάρχουν πολλά σημαντικά πράγματα. Πρώτον, χρειαζόμαστε νέες επενδύσεις για υποδομήνες, λιμενικές εγκαταστάσεις, χώρους εκφόρτωσης για την παράκτια ε, αλληλεία ε, και την αλία σε, με εσωτερικές υδάτινες ε, οδούς. Ε, έτσι θα υπάρχει ισότιμη πρόσβαση στα αλλιευτικά προϊόντα και νομίζω ότι θα βελτιωθεί και η συνεργασία ανάμεσα στους αλλιείς. Δεύτερον, χρειαζόμαστε ένα πακέτο startup, δηλαδή για τους νέους που εισέρχονται στον κλάδο και θέλουν να στήσουν μικρές επιχειρήσεις. Αυτό το πακέτο στήριξης θα έπρεπε να είναι παρόμοιο όπως αυτό που προβλέπεται στον κανονισμό IMFF για την υδατοκαλλιέργεια, ε, για την παράκτια αλία. Αυξάνονται οι ανάγκες ε, και πολλές ε, εκμεταλλεύσεις θα καταρρεύσουν ακόμη πριν στηθούν, πριν σταθούν στα πόδια τους, αν δεν στηρίξουμε τους νέους αλείς. Υπάρχουν επίσης και άλλα είδη, όπως ακόμη και θαλασσοπούλια, όχι μόνο θαλάσσια είδη, που πρέπει να προστατευθούν για δημοκρατία ε, ε, δεν βρίσκονται απαραίτητα στον φυσικό βιότοπό τους ε, και δημιουργείται πρόβλημα με τις φώκες και τους κόρμοράνους που απειλούν την ύπαρξη αυτών των ειδών. Στη συνέχεια... Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε την προσανατολισμό της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον τομέα της αλληλείας Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Μπούρλουν από την Ιρλανδία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Καντέκ για την παρουσίασή του. Θα κάνω σύντομε παρατηρήσει σε σχέση με τον νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσα και Αλία. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Καντέκ ότι πρέπει να στηρίξουμε ε, του ε, αλληλεί, ε, αλλά όχι μόνο. Τα μέλη του πληρώματο των σκαφών πρέπει να τύχουν υποστήριξη επίση. Επίση, χρηματοδότηση για μέτρα ασφαλεία για τα σκάφη και για του αλληλεί, ώστε ε, γενικά ε, να αυξηθεί η ασφάλεια του στόλου. Στη συνέχεια θα πρέπει όσοι έχουν πληγεί από την παρακμάζουσα ε, οικονομική δραστηριότητα να τύχουν υποστήριξη σε παράκτης περιοχές ή εξόχως απομακρυσμένες περιοχές. Έχουν αποδεκατιστεί κάποιες περιοχές λόγω της παρακμής του κλάδου. Θα πρέπει λοιπόν να επανακατευθύνουμε την υποστήριξή μας και να δούμε πού χωλαίνει η βιομηχανία κοινωνία της ε, αλίας. Όχι όμως μέσω των οργανώσεων παραγωγών, γιατί ξέρετε ότι εκείνοι ασχολούνται ως επιτοπλίστων με τα αλλιεύματα. Αλλιεύουν ναι, και οι ίδιες εξάλλου. Θα έπρεπε η επιδότηση να περνάει από τοπικές εταιρικές σχέσεις ή από τις τοπικές αρχές, ούτως ώστε και στο μέλλον να είναι βιώσιμος ο κλάδος. Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, έχουμε δύο ακόμη ερωτήσεις. Ε, Κύριε Παπαγεωργίου και ο Πίνης μου ζητήσει το λόγο. Αν ε, συμφωνείτε, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Κάντεκ όμως πρώτα, για να απαντήσει και κατόπιν, καθώς έχουμε και την ευκαιρία να πιούμε ένα ποτό, να πιούμε μια κοκακόλα, μπορούμε να συνεχίσουμε με το διάλογο. Ο κύριος Καντέκ, παρακαλώ, σε πέντε λεπτά για να ολοκληρώσετε. Ε, εμένα μου επιτρέψετε να μην πιω κοκακόλα, πρόεδρε, να πιω κάτι άλλο. Λοιπόν, ε, να προσπαθήσω να απαντήσω Κύριε Νάντης, αρχικά κατάλαβα ότι ήσασταν ε, υπέρ και της ε, ενίσχυσης ε, για να αντικατασταθούν οι μηχανές και να έχουμε λιγότερο ενεργοβόρες μηχανές στα σκάφη. Εγώ είμαι υπέρ της πρότασης αυτής. Τώρα για την υδατοκαλλιέργεια, αυτό είναι κάτι σημαντικό και ήδη αυτό υπάρχει στο βασικό κανονισμό. Αποτελεί μια, έναν από τους άξονες της μεταρρύθμισης. Προφανώς θα πρόκειται για μια βιώσιμη και υπεύθυνη υδατοκαλλιέργεια

Ε, τώρα ε, ε, μπορούμε να δούμε και τι έχουν κάνει κάποιοι γειτονέ μα. Ε, να μην του αντιγράψουμε γιατί δεν έχουν ε, προβεί σε βιώσιμη διδοκαλλιέργεια. Μπορώ να σα πω ότι η διδοκαλλιέργεια στην Ευρώπη καλύπτει μόνο το 4% τη παγκοσμίω διδοκαλλιέργεια. Και στην αρχή τη αιτία μου είχα κάνει μια σχετική έκθεση, αλλά φτάνουμε σχεδόν το 70% των ψαριών που καταναλώνουμε είναι εισαγωγή. Έτσι λοιπόν, σίγουρα χρειαζόμαστε να έχουμε και μια υπεύθυνη και μια βιώσιμη αλία, αλλά αυτή να συνοδεύεται από μια βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια. Αυτό μου φαίνεται απαραίτητο. Ο κύριος ε, Τέσκλιν από τη Σουηδία. Είπατε, αναφερθήκατε στην ε, αναγκαιότητα του να λάβουμε υπόψη τις περιβαλλοντικές πτυχές. Νομίζω ότι είναι προφανές ε, αυτό για μας οι περιβαλλοντικέ πτυχέ, οι πτυχέ τη βιοπικιλότητας και τη αηφορία τη ελία ε, Μου φαίνεται απαραίτητο ε, αυτό, γιατί αν δεν υπάρχουν ψάρια, όπως είπαμε, δεν θα υπάρχουν καλείς. Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε και την οικονομική και η κοινωνική δραστηριότητα, γιατί έχουμε 140.000 ε, ε, θέσεις σήμερα στον τομέα της Ελίας στην Ευρώπη, αλλά μιλάμε για άμεσες θέσεις εργασίας και έχουμε και έμεσες θέσεις εργασίας στη μεταποίηση και αλλού. Έτσι λοιπόν αυτή η πτυχή, αν δεν εμφανίζεται στην ε, πρώτη Κομισιόν, πρέπει να τη βάλουμε. Όπως είπατε κύριε Τεσκλίνς, είναι λεπτή ισορροπία, δεν είναι εύκολο να την βρούμε και πιστεύω ότι ακριβώς αυτός είναι ο ρόλος μας. Μιλήσατε για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο, αλλά ε, θα σημειώσετε, το είπε και ο συνάδελφος, ε, ότι ε, μιλάμε για Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας. Δεν μιλάμε μόνο για την Αλία εδώ. Έτσι λοιπόν δεν πρέπει εδώ το ένα να είναι εις βάρος του άλλου. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί εδώ. Μου τέθηκε και η ερώτηση σχετικά με τον προπολογισμό του, του ΦΕΠ, του Ταμείου Αλίας, ε, κυρία Γιώτοβα. Υπάρχει ένα έγγραφο πολύ ενδιαφέρον, ε, η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου, η οποία ουσιαστικά κάνει τον απολογισμό της χρήσης ε, του, των Ευρωπαϊκών Ταμείων τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν κάποια θετικά, κάποια αρνητικά, υπάρχουν ε, κάποια πράγματα που δεν πήγαν καλά, είναι προφανές, αλλά σας καλώ επίσης ότι αφορά την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου, να τη διαβάσετε και να την ξαναδιαβάσετε. Γιατί όπως και όλες οι εκθέσει ε, του ελεκτικού συνεδρίου ε, μπορούν να ερμηνευτούν με διαφορετικού τρόπου. Πολλέ φορέ έχουμε απριόρι και κάνουμε διαφορετικέ ερμηνείε. Υπάρχουν δηλαδή πολλά αρνητικά που θέλουμε να τα αναλύσουμε διαβάζοντα με ένα συγκεκριμένο τρόπο την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου, αλλά ε, υπάρχουν και κάποια στοιχεία που καθιστούν απαραίτητη την μεταρρύθμιση και σε επίπεδο χρηματοδότηση. Και το είπε και ο συνάδελφος ε, προηγμένως ε, ότι αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας αφορά και τις θαλάσσιες υποθέσει. Είναι Ταμείο Αλίας και Θάλασσας όπως σας είπα. Είναι αλήθεια ότι το Ταμείο αυτό δεν είναι μόνο για την Αλία αλλά φυσικά είναι πιο ε, μεγάλο από το προηγούμενο, η χρηματοδότηση είναι πιο μεγάλη και θα πρέπει ε, βέβαια να έχουμε ενίσχυση της αλίας, όχι μόνο για τη μετατροπή των αλιαίων ε, και όπως ε, είπατε κύριε Πρίγκελ, θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι υπάρχουν κάποιες κοινότητες που θίγονται ιδιαίτερα. Τώρα, συμφωνώ απόλυτα με όσα είπατε υπόθηκαν. Θα προσπαθήσω ε, να τα συμπεριλάβω όσα ακούστηκαν στη δική μου έκθεση, γιατί και εγώ συμφωνώ, κύριε Νίλαν, από το φιλαντικό Κοινοβούλιο. Μας είπατε, και το είπα και εγώ και ο ίδιος προλίγο, γιατί έχω την ίδια ανησυχία, μας είπατε ότι χρειάζεται και μία ενίσχυση για τους νέους αλείς. δεν ε, θα πρέπει να υπάρχει αύξηση του αριθμού των σκαφών των αλλιών, αλλά σίγουρα πρέπει να ανανεώνονται και οι αλλά και τα σκάφη. Γιατί φυσικά και ο μέσος όρος της ηλικία των ε, αλλιέων είναι αρκετά μεγάλος σήμερα. Πρόκειται για μια δουλειά που μπορεί να επιτρέψει ε, σε όσου ε, απασχολούνται στον τομέα τη να κερδίσουν αξιοπρεπώ ε, τη ζωή του. Έτσι λοιπόν πρέπει να το προσέξουμε και αυτό. Ό,τι αφορά όμω και την προστασία των πόρων, δεν είναι μόνο ο άνθρωπο ε, που είναι έκτο στη γη, υπάρχει και ο κορμοράνο, όπω υπόθηκε. Υπάρχουν και φώκε, έχουμε αυτά τα είδη τα οποία είναι κυνηγετικά. Ο κύριο ε, δεν ξέρω αν είναι ακόμα εδώ, γνωρίζει πάρα πολύ καλά το πρόβλημα που τίθεται από τις φώκες και από τους κορμοράνους και είναι προβλήματα γιατί είναι προστατευόμενα ήδη. Έτσι λοιπόν αυτά είναι θέματα που τα θέτουμε στην Επιτροπή εδώ καιρό και ελπίζω ότι κάποια μέρα θα μπορέσουμε να βρούμε μια λύση σε αυτό το πρόβλημα γιατί μιλάμε για είδη πραγματικά κινητικά. Όταν μιλώ για τους αλληλείς, ε, μιλώ και για το πλήρωμα. Δεν μιλώ μόνο ε, για τους ε, αλληλείς, μιλώ στο σύνολό τους. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Τομείο Θάλασσας και Ελίας καλύπτει τους αλληλείς με αλφα κεφαλαίο. Και επίσης είναι απαραίτητο να ξεχρονίσουμε τα σκάφη για να είναι πιο ασφαλή Ξέρετε, έχουμε ατυχήματα κάθε χρόνο και στη Μεσόγειο, στην Άγχη, στη, Βαλτική, στη Μάνχη, στη Βαλτική, στη Βορειοθάλασσα. Πρέπει να ξεχρονίσουμε τα σκάφη μας για να είναι λιγότερο επικίνδυνα. Πιστεύω λοιπόν ότι και αυτό είναι σημαντικό. Είχαμε μία σειρά θετικών στοιχείων, όπως είπα, κυρίως ε, την επιλεκτικότητα των ε, εργαλείων. Αναφέρεται αυτό στην πρόταση, πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό. Είναι καλή αυτή η πρόταση, πρέπει λοιπόν να την διατηρήσουμε να την επιλέξουμε. Και πάλι να σας πω ότι οι προτάσεις σας ε, και οι ιδέες σας είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Σας ευχαριστώ που τις διατυπώσετε εδώ και σας καλώ επίσης ε, να τις επαναδιατυπώσετε αν θέλετε και γραπτός. Γιατί είναι ακόμη καλύτερο για να θα με βοηθήσετε να εργαστώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σας ξαναδίνω το λόγο. Ελπίζω να το χρόνο. Αλλά όπως σας είπα δεν θα πιω κοκακόλα. Ευχαριστώ Αλέν. Μάλιστα, ολοκληρώνουμε εδώ αυτή τη συνεδρίαση. Ήταν εξαιρετική, όπως σας είπα. Και αυτή είναι η στιγμή των συμπερασμάτων. Πιστεύω ότι εδώ έχουμε μια πολύ σημαντική ιδέα που ήταν η συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων, γιατί αναφυσβήτητα εμπλούτιζε τη συζήτηση, υπήρχαν πάρα πολλέ ερωτήσει, 60 παρεμβάσει σχεδόν. Και πιστεύω ότι είναι λοιπόν σημαντικό. Υπάρχουν βέβαια και πολλά επίμαχα σημεία. Ε, έχουμε τις ε, μεταβάσιμες ελευτικές παραχωρήσεις, τις επορρίψεις, ε, το τι θα γίνει με την λευτική προσπάθεια, όλα αυτά είναι επίμαχα ζητήματα και φυσικά όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να σεβόμαστε το περιβάλλον, αλλά πρέπει και να σεβόμαστε και τα δικαιώματα των αλλιών. Πολλές συμφωνίες, πολλές συμφωνίες, πολλές διαφωνίες, κάποιες πιο γενικού χαρακτήρα, κάποιε πιο συγκεκριμένε. Νομίζω ότι μιλήσαμε για πάρα πολλά, για μια ρεαλιστική μεταρρύθμιση, για τι οργανώσει παραγωγών που πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικέ για την την ανανέωση του στόλου, για την ανανέωση των ε, ε, αλλιέων, της γενιάς των αλλιέων, αλλά και κάτι που υπόθηκε πολλές φορές σήμερα είναι το θέμα της αηφορίας, της βιωσιμότητας. Μιλήσαμε για κάτι που όλοι θέλουμε. Θέλουμε να έχουμε και ψάρια στις θάλασσες, αλλά θέλουμε να λειτουργεί και ο κλάδος. Και είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να το κάνουμε και ε, εδώ Θέλουμε φυσικά να συνεισφέρουμε και εμείς ως Επιτροπή Αλίας και φυσικά κάθε συνεισφορά και δική σας θα είναι ευπρόσδεκτη. Κλείνω σας ευχαριστώντας όλους όσους συμμετείχατε στην οργάνωση αυτής της έκτακτης συνεδρίασης σήμερα. Ευχαριστώ την ε, Γραμματεία της Επιτροπής Αλίας, ε, την ε, Αρμόδια Υπηρεσία που έρχεται σε επαφή με τα Εθνικά Κοινοβούλια και φυσικά ο Πρόεδρος και μάλλον λέει θέλω να ευχαριστήσω και τους Γερμινείς, ευχαριστούμε και εμείς. Και σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε εδώ σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα ήθελα να σας ε, καλέσω στον πρώτο όροφο να πιούμε κάτι, αν όχι μια κοκακόλα, ένα ποτήρι κρασί, ό,τι άλλο επιθυμείτε. Σας ευχαριστώ πολύ και θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας ε, εκτός της αίθουσας.